Καλησπέρα σα, συνάδελφοι, λέει ο κύριο Γκουαλτιέρη. Α αρχίσουμε τη συνεδρίαση. Παρακαλώ, πρώτα-πρώτα να εγκρίνουμε την ημερησία διάταξη θεωρώ ότι εγκρίθηκε. Έχω και κάποια ανακοίνωση όσον αφορά το γλυσκό καθεστώ, γιατί επειδή έχουμε σήμερα ε, συνδιαλλαγή για τον προπολογισμό, πάρα πολλέ καμπίνε απουσιάζουν, είναι κλειστέ κατά την δική μα συνεδρίαση την σημερινή. Δανέζικα, Ουγγρικά, Σλοβενικά, Κροατικά και Μαλτέζικα. Ζητούμε συγγνώμη για ε, αυτήν την ενόχληση και επίσης θα πρέπει να εγκρίνουμε τα πρακτικά της προηγουμένης συνεδριάσεω στο, των συνδυάσεων, μάλλον Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου. Θεωρώ ότι εγκρίνονται και σας ευχαριστώ. Πάμε τώρα στο σημείο του παριθμών 4 της ε, ημερησίας διατάξεως που είναι ο νομισματικός διάλογος με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης τον Μάριο Ντράγκη τον οποίο και καλωσορίζουμε. Σας ευχαριστούμε που ξαναήλθατε εις αυτές τις ε, τακτές όσο και επικοδομητικές μας συναντήσεις για διάλογο και επίσης ε, περιμένουμε να μας ενημερώσουν σαν πρόσφατες τις πρόσφατες ε, ε, αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης συγκεκριμένα όσον αφορά τα, το, το πρόγραμμα ABS, τα τιτλοποιημένα δάνεια, τα, τα, ομόλογα, το, τι γίνεται με τους ολογισμούς, επίσης το, την δέσμευση για τα επιπλέον συμβατικά ε, μέσα και εργαλεία οικονομικής πολιτικής εάν χρειαστεί και επίσης οι συντονιστές έχουν επισημάνει κάποια ε, συγκεκριμένα ζητήματα ε, επί των οποίων εργαζόμαστε όσον αφορά το, το πλαίσιο για τα collaterals και επίσης τα μέτρα νομισματικής πολιτικής. Ο συνήθως θα ξεκινήσουμε με μία εισαγωγική δήλωση ο πλευράς του κ. Ντράκη και κατόπιν θα έχουμε το σύνηθες πεντάλεπτο ερωταπαντήσεων. Κύριε Ντράγη, σας ευχαριστούμε και σας δίνουμε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές της Οικονομικής και Νομισματικής Επιτροπής, κυρίες και κύριοι. Είναι μεγάλη χαρά για μένα που επανέρχομαι εδώ στην Επιτροπή σας μετά την ε, τελευταία ακρόαση που είχαμε εδώ το 2014. Αυτή η ακρόαση έρχεται μετά από διάφορες αλλαγές οι οποίες προηγήθηκαν. Επρόκειτο για μία χρονιά νομοθετικών και θεσμικών αλλαγών που έγιναν. Από το 2014 ε, έχουμε την ε, γέννηση της Τραπεζικής Ένωσης με τον ενιαίο μηχανισμό εξυγίανσης. Έχουμε την αρχή του ενιαίου μηχανισμού εποπτείας και ολοκληρώσαμε επιτυχώς επίσης την ε, αξιολόγηση των ισολογισμών των τραπεζών. Και ήταν ε, πράγματι μια χρονιά γεμάτη προκλήσει για την νομισματική πολιτική, διότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα χρειάστηκε να υιοθετήσει διάφορα μέτρα προκειμένου να αντιμετωπίσει του κινδύνου από ε, μια σκοτεινή κάπως οικονομική προοπτική. Επιλέξατε δύο θέματα για σήμερα. Τη σχέση του χρηματοπιστωτικού κατακαιρματισμού και την νομισματική πολιτική, αλλά και το πλαίσιο του ευρωσυστήματος. Εγώ θα ασχοληθώ με τα δύο αυτά θέματα, αλλά επιτρέψτε μου πρώτα απ' όλα να σας εξηγήσω λιγάκι ποια είναι η αξιολόγησή μας όσον αφορά τις οικονομικές προοπτικές. Ο ρυθμός της οικονομικής ανάπτυξης στο ευρώ ήταν πιο αδύνατος τα τελευταία, τους τελευταίους μήνες του καλοκαιριού και οι προβλέψεις είναι προς τα κάτω. Συγχρόνως όμως υπάρχουν προοπτικές για μια ε, μεσαία ανάκαμψη το 2015 και 2016. Η ζήτηση πρέπει να στηριχθεί από διάφορους παράγοντες. Μεταξύ άλλων έχουμε τα μέτρα που έχουμε υιοθετήσει για την νομισματική μας πολιτική και η πρόοδος που έχει γίνει όσον αφορά τη δημοσιονομική εξυγίανση και η μεταρρυθμίσεις που έγιναν σε διάφορες χώρες. Επιπλέον, η υψηλή ανεργία, η δυναμικό το οποίο δεν χρησιμοποιείται είναι παράγοντες οι οποίοι χρειάζονται διόρθωση, διότι αλλιώς θα περιορίσουν ακόμα περισσότερο την ανάκαμψη. Οι κίνδυνοι όσον αφορά τις οικονομικές προοπτικές συνεχίζουν να μας ε, οδηγούν σε πεσοδοξία. Ιδιαίτερα ο αδύναμος ρυθμός ανάπτυξης στην Ευρωζώνη μαζί με τους γεωπολιτικούς κινδύνους έχουν σαν αποτέλεσμα να περιορίζουν την εμπιστοσύνη και άρα να περιορίζουν και τις ιδιωτικές επενδύσεις. Επιπλέον δεν, υπάρχουν δεν υπάρχει αρκετή πρόοδος στις αγροτικές μεταρρυθμίσεις στις χώρες της Ευρωζώνης που οδηγούν σε επιπλέον κινδύνους όσον αφορά τις οικονομικές προοπτικές. Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη παραμένει πολύ χαμηλός. Τον Οκτώβριο ήταν 0,4%. Ε, Αναμένουμε να παραμείνει γύρω στα σημερινά χαμηλά επίπεδα και τους επόμενους μήνες πριν να αυξηθεί σταδιακά κατά τη διάρκεια του 2015 και του 2016. Κοιτώντας προς το μέλλον, ελέγχουμε τους κινδύνους όσον αφορά τις εξελίξεις των τιμών. Τα τελευταία νομισματικά στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει μια περιορισμένη βασική ανάπτυξη όσον αφορά την προσφορά χρήματος. Η ετήσια ανάπτυξη έχει αυξηθεί λίγο τους πρόσφατους μήνες. Και φαίνεται ότι βρισκόμαστε σε μια καμπή όσον αφορά την ε, αύξηση των πιστώσεων. Επιτρέψτε μου να στραφώ τώρα στον χρηματοπιστωτικό κατακαιρματισμό, το πρώτο θέμα που θέλατε να εξετάσουμε σήμερα. Ο κατακαιρματισμός σε διάφορους τομείς των χρηματοπιστωτικών αγορών είναι ένα μεγάλο εμπόδιο όσον αφορά την ε, εφαρμογή της νομισματικής μας πολιτικής και τελικά προκειμένου να μπορέσουμε να έχουμε αποτελέσματα όσον αφορά την εντολή μας. Επίσης, εξαιτία διαφόρων δράσεων η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που έλαβε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ο κατακαιρματισμός έχει περιοριστεί σημαντικά από τότε που άρχισε η χρηματοπιστωτική κρίση. Τα επίπεδα μη εξασφαλισμένων νομισματικών αγορών περνούν μέσα σε συναλλαγές, σε λογικά spreads και έχουν απομακρυνθεί από το υψηλό σημείο που βρισκόντουσαν το 2012. Οι εξελίξεις αυτές δείχνουν επίσης επιστροφή της εμπιστοσύνης των επενδυτών στην Ευρωζώνη. Όμως, εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση όπου ο πρόσφορος προσανατολισμός νομισματικής πολιτικής μας δεν έχει φτάσει ακόμα εκεί που θα θέλαμε στην Ευρωζώνη. Αυτό συμβαίνει επειδή οι πιστοτικές αγορές σε ορισμένα μέρη της Ευρωζώνης εξακολουθούν να δυσκολεύονται και έχουμε μόνο μερικά πολύ δειλά δείγματα ανάκαμψης. Το αποτέλεσμα είναι ότι η ανάπτυξη πιστώσεων, η αύξηση πιστώσεων εξακολουθεί να είναι περιορισμένη και οι συνθήκε πιστώσεων, παρόλο που έχουν διευκολυνθεί κάπως, παραμένουν δύσκολες. Κάτι πολύ σημαντικό είναι ότι το κόστος της χρηματοδότησης τραπεζών έχει βελτιωθεί, αλλά εξακολουθεί να είναι κάτι ιδιαίτερα ψηλό σε πολλές χώρες μέλη. Εκεί όπου είναι χαμηλότερα δεν ε, καταφέρνουν να επηρεάσουν πλήρως την πραγματική οικονομία. Τα μέτρα νομισματικής πολιτικής που αποφασίστηκαν τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο φέτος με μακροπρόθεσμες ε, δράσεις αναχρηματοδότησης και αγορά προγραμμάτων ε, τίτλων εξασφαλισμένων με περιουσιακά στοιχεία και καλυμμένων ομολόγων σχεδιάστηκαν για να ξεπεραστούν τα εμπόδια αυτά θα ενισχύσουν την εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής, την ε, παροχή πιστώσεων στην οικονομία της Ευρωζώνης και το αποτέλεσμα θα είναι να έχουμε καλύτερο προσανατολισμό νομισματικής πολιτικής. Βλέπουμε κάποια δείγματα ότι η διευκόλυνση αυτή πιστώσεων αρχίζει να φαίνει αποτελέσματα. Από την αρχή του Ιουνίου η τιμή του χρήματος έχει μειωθεί μέσα στο πλαίσιο της ληξιμότητας. Τώρα η επόμενη καμπή είναι κάτω από το 0 σε ορίζοντα 2 ετών. Το Ιόνια δεν πρόκειται να ξεπεράσει τα 25 βασικά, βασικούς βαθμούς πριν από το 2018. Το τρίμηνο Eurobor, το οποίο είναι ένα σημαντικό στοιχείο της νομισματικής μας πολιτικής για δανεισμό, έπεσε σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα και τώρα είναι κοντά στο 0 και οι πολιτικές αποφάσεις, ιδιαίτερα αυτές που ανακοινώθηκαν το Σεπτέμβριο, οδήγησαν σε μια μείωση των spreads και σε άλλες κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων και των ABS, των καλυμμένων ε, ομολόγων και των κρατικών ομολόγων. Αλλά χρειάζεται περισσότερος χρόνος προκειμένου να υλοποιηθούν ε, πλήρως οι θετικές επιπτώσεις από τα τελευταία μέτρα. Στα πλαίσια αυτά, επιτρέψτε μου να υπογραμμίσω ότι έχουμε δεσμευτεί για όλα μας τα μέτρα, είτε πρόκειται για δράσεις δανεισμού, είτε πρόκειται για τις αγορές κρατικών ομολόγων, σε τέτοιο βαθμό που να μπορούμε να στηρίξουμε όπως πρέπει τον πληθωρισμό και την ανάκαμψη της οικονομίας στην Ευρωζώνη. Όλα αυτά τα μέτρα θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στον ισολογισμό μας που αναμένουμε να φτάσει στα επίπεδα των αρχών του 2012. Αυτό θα διασφαλίσει ότι ο προσανατολισμός της μαθηματικής μας πολιτικής θα συνεχίσει σταδιακά να ανακάμπτει και θα φτάσει με ε, πληθωρισμό που να είναι πολύ κοντά στο 2%, λίγο πιο κάτω αλλά κοντά στο 2%. Παρ' όλα αυτά πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για τους κινδύνους που μπορεί να επηρεάσουν παρετέρω τον πληθωρισμό, ιδιαίτερα αν υπάρξει ένας αδύναμος ρυθμός ε, οικονομικής μεγένθησης. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να παρακολουθούμε στενά και να αξιολογούμε την καταλληλότητα των μέτρων μας νομισματικής πολιτικής. Εάν πρέπει να υπάρξουν αλλαγές, αν υπάρξουν δηλαδή συνεχιζόμενοι κίνδυνοι, τότε το Δικητικό Συμβούλιο ομόφωνα έχει δεσμευτεί να υιοθετήσει επιπλέον μη συμβατικά μέτρα αν χρειαστεί. Στα πλαίσια αυτά, επίσης, Έχουμε αναθέσει στο προσωπικό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των Επιτροπών ε, του Ευρωσυστήματος με έγκαιρη προετοιμασία προκειμένου να υιοθετηθούν επιπλέον μέτρα αν χρειαστεί. Τέτοια μέτρα θα μπορούσαν να συμπεριλαμβάνουν επιπλέον αλλαγές στο μέγεθος και στην σύνθεση του ισολογισμού του ευρωσυστήματος εφόσον χρειάζεται να κάνουμε περισσότερα πράγματα για να πετύχουμε σταθερότητα τιμών μεσοπρόθεσμα. Από μόνη της όμως η νομισματική πολιτική δεν μπορεί να ξεπεράσει τον χρηματοπιστωτικό κατακαιρματισμό στην Ευρωζώνη. Ο κατακαιρματισμός μεταξύ εθνικών συνόρων δείχνει ότι υπάρχουν εθνικές ανισορροπίες και θεσμικές αδυναμίες. Για να τα ξεπεράσουμε αυτά χρειάζονται αποφασιστικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις από πλευράς των εθνικών κυβερνήσεων προκειμένου να βελτιωθεί το επιχειρηματικό περιβάλλον και να υπάρξουν κίνητρα για επενδύσεις με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικότητας, τη δημιουργία απασχόλησης και την αύξηση της οικονομικής μεγέθυνσης στην οικονομία μας. Επίσης, Όσον αφορά την χρηματο... τον χρηματοπιστωτικό κατακαιρματισμό, απαιτείται και αντιμετώπιση άλλων ελλείψεων σε οικονομική και χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση. Τώρα έχουμε προχωρήσει πολύ φέτος. Όσον αφορά την Τραπεζική Ένωση, όσον αφορά την συνολική αξιολόγηση και τον SSM. Αυτό σημαίνει ότι ιδιαίτερα Όσον αφορά τον SRM, θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε περισσότερο με τον ενιαίο δηλαδή ε, Ταμείο και θα μπορέσουμε έτσι να καλύψουμε περισσότερο τις ανάγκες μας. Τώρα αν κοιτάξουμε πιο πέρα. Μια μεγαλύτερη ολοκλήρωση των ε, χρηματοπιστωτικών αγορών, αυτό που ονομάζουμε Ένωση Αγορών Κεφαλαίου, είναι κάτι δικαιολογημένο προκειμένου να μειωθεί περισσότερο ο κατακαιρματισμός των χρηματοπιστωτικών αγορών και θα βελτιωθεί έτσι και η χρηματοδότηση του SME, κάτι το οποίο θέλουμε. Δεν έχω καμία αμφιβολία λοιπόν ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που είναι συνομοθέτης θα παίξει και πάλι ένα αποφασιστικό ρόλο επ' αυτού. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ τώρα στο δεύτερο θέμα. Το πλαίσιο αυτού του ευρωσυστήματος σχεδιάστηκε έτσι ώστε να πετύχουμε συγχρόνως δύο στόχους. Πρώτον, να προστατεύσουμε το ευρωσύστημα από απώλειες. Αυτό ζητάει και το ίδιο το καταστατικό τη ευρωπαϊκή Κεντρικής Τράπεζας και δεύτερον προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι οι πράξεις πιστώσεων του ευρωσυστήματος μπορούν να λάβουν χώρα χωρίς προβλήματα και με αρκετές εγγύσεις. η πρόσφατη εμπειρία μας έχει δείξει ότι αυτό το δίδυμο ήταν πάρα πολύ αποτελεσματικό. Μέχρι τώρα το ευρωσύστημα ποτέ δεν χρειάστηκε να αναγνωρίσει απώλειες εξαιτίας των πιστοτικών ε, δράσεων του ευρωσυστήματος. Σε λίγες περιπτώσεις όπου οι αντισυμβαλόμενοι ε, οδηγήθηκαν σε πτώξεις, σε περίπτωση, για παράδειγμα, της Lehman Brothers, τότε το ευρωσύστημα μπόρεσε να καλύψει πλήρως την έκθεσή του, χρησιμοποιώντας τις εγγύσεις το εγκυτικό πλαίσιο. Συγχρόνως, το εγγυητικό πλαίσιο διασφάλισε ότι οι τράπεζες μπόρεσαν να έχουν αρκετή ρευστότητα από την Κεντρική Τράπεζα καθ' όλη τη διάρκεια της κρίσης. Αυτό έγινε περισσότερο ορατό στα πλαίσια δύο πολύ μεγάλων σε χρονικό διάστημα ε, πράξεων αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας το 2011 και 2012. Πήραν λοιπόν έτσι τέτοια εγκυμένη ρευστότητα η τράπεζα στις τάξεις των 524 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα σε 10 μόνο εβδομάδες. Αυτό το βασικό πλαίσιο λοιπόν του εγκαιτικού πλαισίου παρέμεινε το ίδιο από την αρχή της Νομισματικής Ένωσης. Τα τρία μέρη του, ευρω... του εγγυητικού αυτού πλαισίου του ευρωσυστήματος. Πρώτα απ' όλα το πλαίσιο των αντισυμβαλόμενων, το, τα βασικά κριτήρια για τα βασικά περιουσιακά στοιχεία και τρίτον τα μέτρα ελέγχου κινδύνου παρέμειναν αμετάβλητα. Το ευρωσύστημα εξακολουθεί να έχει ένα ευρύ πλαίσιο με κριτήρια τα οποία παραμένουν όπως είχαν. Αυτό δείχνει ότι ο σχεδιασμός του εγγυητικού πλαισίου του ευρωσυστήματος παραμένει εύρωστο. Παρ' όλα αυτά χρειάστηκαν κάποιες αλλαγές για να διασφαλίσουμε την ε, καλή εφαρμογή της νομισματική μας πολιτικής σε περιόδους πίεσης των χρηματοπιστωτικών ε, αγορών προκειμένου υπάρχει πρόσβαση σε ρευστότητα. Πρώτα απ' όλα, το πλαίσιο αυτό ποτέ δεν πρέπει να δρά ε, προκυκλικά. Ο περιορισμός της ρευστότητας των τραπεζών, για παράδειγμα, μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο όχι μάλιστα μόνο στις πιο ευάλωτες τράπεζες, αλλά σε ολόκληρο το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Τελικά αυτό θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο στον ισολογισμό των κεντρικών τραπεζών και όχι να τις προστατεύσει. Οπότε προκειμένου να οι πολλοί αντισυμβαλόμενοι να μπορούν να συμμετέχουν στην ε, δράσει αναχρηματοδότησης, το σύστημα ε, χαλάρωσε κάπως τα κριτήρια για τα βασικά περιουσιακά στοιχεία και αυτό έγινε πολλές φορές. Για παράδειγμα, από το 2008 μέχρι το 2011 και μετά από το 2012 όπου δεχτήκαμε ε, σε ξένο νόμισμα ε, εμπορεύσιμα περιουσιακά στοιχεία. Το 2012 δημιουργήσαμε ένα, το Additional Credit Claims πλαίσιο ιδιαίτερα προκειμένου το MBS να μπορέσει να καλύψει τα απαιτούμενα κριτήρια. Το ηγετικό πλαίσιο του ευρωσυστήματος ήταν περίπλοκο από την αρχή και όχι μόνο επειδή τα εθνικά πλαίσια που προηγήθηκαν αυτού διέφεραν μεταξύ τους, αλλά και γιατί ο στόχος της Νομισματικής Ένωσης ήταν να δοθεί πρόσβαση σε ένα μεγάλο έύρο αντισυμβαλόμενων, σε αντίθεση με τι κεντρικές τράπεζε όπου συμμετέχουν λίγοι αντισυμβαλόμενοι. Οπότε το κεντρικό πλαίσιο έπρεπε να λάβει υπόψη τα διάφορα εθνικά τραπεζικά συστήματα και χρηματοπιστωτικές αγορές. Μερικέ εθνικέ κεντρικέ τράπεζε, για παράδειγμα, δέχονταν ισχυρισμού ω εγγύηση, ενώ άλλε όχι. Για να υπάρχουν κοινέ προδιαγραφές, θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη όλα τα χαρακτηριστικά, ενώ συγχρόνω θα έπρεπε να διασφαλίσουμε επαρκείς εγγύσεις. Συνεπώς, τώρα ποια είναι η πρόκληση που έχουμε μπροστά μας. Είναι το κεντρικό πλήσιο να γίνει πιο απλό, περισσότερο διάφανο και να μην εμποδίζει του αντισυμβαλόμενους να έχουν πρόσβαση. Συνεπώς, κύριε και κύριοι, το 2014 ήταν, όπως είπα και στην αρχή, μια χρονιά μεγάλων αλλαγών. Όσα πετύχαμε μέχρι τώρα όμως δεν φτάνουν. Το 2015 πρέπει να είναι η χρονιά όπου όλοι οι φορείς της Ευρωζώνης, των κυβερνήσεων και των ευρωπαϊκών θεσμών μαζί θα ενώσουν τις δυνάμεις τους ώστε οι οικονομίες μας να μπουν και πάλι στον καλό δρόμο. Η νομισματική πολιτική από μόνη της δεν θα τα καταφέρει και γι' αυτό Επιγόντως υπάρχει ανάγκη να συμφωνήσουμε βραχυπρόθεσμα σε δεσμεύσεις για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στις χώρες μέλη και καλή εφαρμογή του Συμφώνου Ανάπτυξης και Σταθερότητας να συμφωνήσουμε επίση για του σωστού προσανατολισμού τη νομισματική μα πολιτική στην Ευρωζώνη και μια στρατηγική επενδύσεων προκειμένου να διασφαλίσουμε την βιωσιμότητα της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης. Προσβλέπω λοιπόν στη συζήτησή μας και συγγνώμη αν μίλησα περισσότερο από ό,τι συνηθίζω. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ Πρόεδρε Ντράγκη για την σημαντική αυτή παρουσίαση και ας ακούσουμε τον πρώτο μιλητή του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Παύλος Αλβοδίδη ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Ντράγκη. Καλώς ορίσατε και σας ευχαριστούμε για όσα μας είπατε. Εγώ θα ήθελα τώρα να αναφερθώ σε αυτά τα οποία εσείς έχετε πει κάποια στιγμή όσον αφορά την αύξηση του, αυτού του 3 ευρώ όσον αφορά τα, τα, τα χρήματα. Είπα ότι αυτό είναι προσδοκία, δεν είναι στόχος. Τι θέλετε να πείτε. Τι εννοείτε προσδοκία. Επίσης, σε σχέση με αυτά τώρα που μας είπατε, φυσικά συμφωνώ 100% ότι η νομισματική πολιτική μόνη της δεν είναι δυνατόν να δώσει όθηση προς ανάπτυξη και προς δημιουργία απασχόληση και ότι όπως είπατε και εσείς αυτό το οποίο χρειάζεται είναι κάποιες μεταρρυθμίσεις και ανάληψη δράσης αποφασιστική με τους άλλους εμπλεκομένους. Αυτό που θα ήθελα να ξέρω είναι αν μπορείτε πέστε μας τη γνώμη σας πιο συγκεκριμένα, πέστε μας δυο λόγια τι γίνεται, ποιες χώρες ή και θεσμικά όργανα θα πρέπει να αναλάβουν δράση κατά αυτόν τον τρόπο και συγκεκριμένα τι, τι, τι μέτρα θα πρέπει κατά τη γνώμη σας να ληφθούν ώστε η νομισματική πολιτική να μπορέσει να έχει κάποια αποτελέσματα ή να έχει πιο απτά αποτελέσματα όσον αφορά την πρόθεση της απασχόλησης και της οικονομικής ανάπτυξης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο Μεταξύ Ιουνίου και Σεπτεμβρίου στο έχουμε πάρει μια σειρά από διάφορα μέτρα ε, ε, από το τέλτρος μέχρι την απόφαση σε σχέση με την εξαγορά αυτών των ομολόγων των καλυμμένων των ABS και εμείς ε, πιστεύουμε ότι τα μέτρα αυτά τα οποία έχουν ληφθεί πρόκειται να βοηθήσουν ούτως ώστε να πετύχουμε τις προσδοκίες ε, σε σχέση με τον πληθωρισμό, δηλαδή περί το 2% ή κάτω από αυτό. Εάν επομένως εμείς κάτσουμε να αξιολογήσουμε και καταλήξουμε ότι αυτά τα μέτρα δεν αρκούν για να επιτύχουν αυτό το στόχο και έτσι ε, οι προσδοκίες, οι μεσοπρόθεσμες πρόκειται να λάβουν κατεύθυνση προς τα χείρο, τότε σε αυτή την περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως σας είπα, ομόφωνο είναι ότι πρόκειται να ληφθούν και άλλα επιπλέον μέτρα τα οποία δεν θα είναι συμβατικού χαρακτήρα. Οπότε εμεί θεωρούμε ότι αυτού του είδους ο ισολογισμός θα προσεγγίσει τα επίπεδα του Μαρτίου του 2012. Όπως σας προείπα, είμαι θα έτοιμοι να πάρουμε νέα μέτρα εάν η κατάσταση για τον πληθωρισμό μέσω πρόθεσμα ε, πάει ταχύρω για να αποδειχθεί ότι δεν αρκούν τα μέτρα τα οποία έχουμε ήδη πάρει ούτως ώστε να ανασχέσουμε αυτή την επιδείνωση στον πρώτο μέτωπο του πληθωρισμού. Για το δεύτερο σημείο τώρα νομίζω έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο τώρα πια ότι και η επεκτατική ε, ε, νομισματική αλλά και δημοσιονομική πολιτική έχουν επιπτώσεις περιορισμένες όσον αφορά την οικονομία. Άπαξ και το, η οικονομική συγκυρία, το οικονομικό περιβάλλον δεν είναι ευεπίφορο ή τις επενδύσεις. Οπότε, γι' αυτό το λόγο έχουμε επανειλημμένα πει ότι οι διαρθωτικές αλλαγές είναι πάρα πολύ σημαντικές. Κάθε χώρα δε έχει το δικό της θεματολόγιο και τις δικές της ανάγκες. Γενικώ πάντως δύο κατηγορίες έχουμε τέτοιες ε, ε, αλλαγές. Πρώτα-πρώτα τον ανταγωνισμό, η αγορά, ούτως ώστε να πάμε προς την ολοκλήρωση της ε, νομοθεσίας για την ενιαία αγορά. Εκεί θα πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα. Δεύτερον, έχουμε και την αγορά εργασίας. Οπότε διαπιστώνουμε ότι οι χώρες που έχουν προβεί σε τέτοιου είδους μεταρρυθμίσεις τώρα έχουν ωφεληθεί, έχουν πάει προς την ανάκαμψη. Επομένως, είναι ακόμα νωρίς να πούμε για το κατά πόσον υπάρχει ένα συσχετισμός άμεσος, έντονος μεταξύ των δύο μεταβλητών, αλλά υπάρχει, ένα, υπάρχει σχέση. Οι χώρες οι οποίες έχουν ε, καταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης είναι εκείνες όπου έχουν αναλυφθεί ε, των κάποιες μεταρρυθμίσεις διαρθωτικές. Ευχαριστώ να σας τα πω στα πορτογαλικά. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Και συμπαθάτε με γιατί δεν θα μπορέσω να κάτσω μέχρι το τέλος της συνεδριάσεως γιατί έχω κάποια υποχρέωση και πρέπει κάπου να πάω. Έχω όμως την εξής ερώτηση. Η νομισματική πολιτική και τα επιτόκια που ανέκαθεν ήταν το εργαλείο για την ε, ανάκαμψη της, ε, του ενίου νομίσματος. Ε, σχεδόν τώρα μας εξαντλήθηκαν ή βρισκόμαστε εκεί κοντά στο σημείο εξάντλησής τους. Επομένως, η σημερινή μας συγκυρία με αυτές τις τόσο εντυπωσιακε ανισορροπίες σε κάποιες χώρες, με κάποιο διαρθρωτική ανεργία τεραστίων διαστάσεων. Και έχουμε επίσης κάποιες οικονομίες που έχουν αναλάβει τις μεταρρυθμίσεις, όπως είπατε κι εσείς υπάρχει παρόλα αυτά μία μεγάλη δυσκολία από πλευράς ζήτησης. Άρα αυτές οι μεταβλητές δεν είναι αρκετά σημαντικές ούτως ώστε να φτάσουμε εκεί που θέλαμε στο 2012. Δηλαδή να βρεθούν οι πρόεδροι των βασικών ε, ε, οργάνων ε, χρηματοπιστωτικών και να, όπως τότε μαζί με τα ευρωπαϊκά όργανα στο πιο υψηλό επίπεδο να συμφωνήσουν, να κλείσουν μια συμφωνία όσον αφορά μια πολιτική ανάκαψη για την Ευρώπη. Και, εν πάση περιπτώσει, να δοθεί μια όθηση για τις επενδύσεις. Όχι μόνο στο εσωτερικό των χωρών, αλλά και γενικότερα στην Ευρωζώνη. Άρα η κατάσταση είναι πάρα πολύ σοβαρή και θα πρέπει να δούμε πώς οι, οι θύνοντες, οι, πιο υψηλά ειστάμενε στα χρηματοπιστωτικά θα πρέπει να βρεθούν και να τα βρουν γιατί η Κεντρική Τράπεζα δεν μπορεί να τα κάνει όλα μόνη της. Ναι, δεν μπορώ να συμφωνήσω μαζί σας. Η νομισματική πολιτική έχει καταφέρει πολλά και μπορεί να καταφέρει ακόμη περισσότερα εάν οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις αναλυφθούν. Αλλά όμως δεν μπορούμε έτσι να τα καταφέρουμε όλα. Επομένως χρειάζεται ε, δημοσιονομική πολιτική. Και επίσης ο τρίτος πυλώνας για αυτό το πλαίσιο πολιτικής είναι οι διερευνητικές ε, μεταρρυθμίσεις. Όμως αυτό το οποίο επιπλέον χρειάζεται είναι το να επιστρέψει η εμπιστοσύνη όσον αφορά το οικονομικό περιβάλλον και εμπιστοσύνη προς την Ευρωζώνη. Και για να συμβεί κάτι τέτοιο, αυτό το οποίο χρειάζεται κυρίως είναι το να υπάρχει από πολιτική και οικονομική πλευρά μια τέτοια δομή που να δείχνει, να δείχνει σε όλο τον κόσμο ότι μπορούμε να συνεργαστούμε, να κινηθούμε μαζί προς μια περισσότερη ολοκλήρωση. Να, πώς θα υπάρξει η εμπιστοσύνη. Δεν έχει να κάνει με το χρήμα, με τα οικονομικά, κάθε αυτά αλλά περισσότερο με την μακρόπνοη σταθερότητα του πλαισίου που έχουμε. Yes, you have the time. Ε, como ainda tenho tempo, Αφού πιέζει ο χρόνος, έχω μόνο μία επιπρόσθετη ερώτηση, λέει κυρία Φερέ, για κάτι άλλο το οποίο εσείς αναφέρατε. Μας ενημερώσατε όσον αφορά τι γίνεται το backstop για το Ταμείο επίλυση των διαφορών και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ βασικό για τα, ε, ε, για τα κράτη-μέλη. Αυτό για τον μηχανισμό στήριξης δηλαδή. Πολλές μεταβολές έχουν γίνει όσον αφορά τον μηχανισμό στήριξης και όλων των άλλων σταθερών. Είναι πολύ σημαντικό το, αυτό το όργανο, το Resolution Fund. Και επίσης τώρα υπάρχει περισσότερη κεφαλαιακή επάρκεια μετά από όσα έγιναν Επίσης έχουν αλλάξει πάρα πολλοί κανόνες για τη λειτουργία του, οπότε τώρα η, η δυνατότητα του τραπεζικού συστήματος να απορροφήσει τις, τους κλονισμούς και τις, τις ζημίες είναι καλύτερη. Επίσης λέμε τώρα ότι έχουμε 50 δις που έχει πρικοδότηση αυτό το ταμείο και το ρώτημα είναι αν αυτά φτάνουν. Εγώ θα έλεγα ότι είναι σαφές ότι είναι σαφής η συμφωνία ότι έχουμε ενισχύσει τις δυνατότητες του Ταμείου Στήριξη. Ο κύριος Νότης Μαριάς. Για το Όπως προκύπτει από την έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2013, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εφαρμόζοντας το πρόγραμμα για τις αγορές τίτλων S&P αγόρασε στη δευτερογενή αγορά με σημαντική έκπτωση κρατικά ομόλογα της ελλάδας της ιταλίας της πορτογαλίας της ισπανίας και της ιρλανδίας ύψους 219,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. πλην όμως κάθε φορά η ΕΚΤ απαιτεί και επιτυγχάνει την εξόφληση των ομολόγων αυτών στην ονομαστική τους αξία κερδοσκοπώντας έτσι ασύστολα χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της πατρίδος μου της ελλάδος καθώς η ΕΚΤ αγόρασε κατά τη διάρκεια της κρίσης ομόλογα του ελληνικού δημοσίου στην δευτερογενή αγορά με έκπτωση τουλάχιστον 40% καταβάλλοντας 35 δις ευρώ πλην όμως απαιτεί να εξοφληθεί στην ονομαστική αξία των ομολόγων αυτών που ανέρχονται σε 57 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή η ΕΚΤ θέλει να βγάλει κέρδος 22 δις ευρώ κερδοσκοπώντας σε βάρος του φτωχοποιημένου από τα μνημόνια ελληνικού λαού. Για φέτος η ελληνική κυβέρνηση με τις εντολές της Τρόικας, δηλαδή και της ΕΚΤ, επέβαλε δυσβάστακτους φόρους στους Έλληνες πολίτες για να πληρώσει στην ΕΚΤ και μάλιστα στην ονομαστική τους αξία ομόλογα ύψους 10 δις ευρώ, ενώ η ίδια η ΕΚΤ κύριε Ντράγκη τα αγόρασε πληρώνοντας 6 δι ευρώ. Αυτό όμως είναι καθαρή κερδοσκοπία και μην μου πείτε κύριε Ντράγκη ότι η ΕΚΤ επιστρέφει δήθεν τα κέρδη στην Ελλάδα. Διότι πρώτον, η όποια επιστροφή αφορά μόνο μικρό μέρος των κερδών και όχι όλα τα κέρδη. Δεύτερον, τα εν λόγω επιστρεφόμενα κέρδη πηγαίνουν αποκλειστικά για την εξόφληση του χρέους, άρα επιστρέφουν πίσω στους δανειστές. Τρίτον, η όποια ενδεχόμενη επιστροφή μέρους των κερδών γίνεται υπό την προϋπόθεση εφαρμογής διαφόρων σκληρών μνημονιακών μέτρων. Τέσσερα, για να πληρωθούν στην ονομαστική τους αξία τα κερδοσκοπικά ομόλογα της ΕΚΤ η Ελλάδα δανείζεται κάθε φορά τα αντίστοιχα ποσά από τον EFSF και έτσι διαιωνίζεται η παρουσία της Τρόικας και των Μνημονίων. Πέντε, μόνο για το 2014 η ΕΚΤ δεν έχει επιστρέψει μέχρι στιγμής κέρδη 1,7 δισεκατομμυρίων ευρώ δημιουργώντας χρηματοδοτικό κενό στην Ελλάδα. Προτείνω λοιπόν κύριε Ντράγκη να δεχθείτε να μην εξοφληθούν τα ελληνικά ομόλογα στην ονομαστική τους αξία αλλά η ΕΚΤ να πληρωθεί μόνο το ποσό που πλήρωσε για την αγορά των ομολόγων αυτών, συν τον νόμιμο τόπο. Αυτό θα σημάνει μείωση του ελληνικού χρέους κατά 22 δισεκατομμύρια ευρώ, χωρίς η ΕΚΤ να υποστεί καμία ζημιά. Συμφωνείτε με την πρόταση αυτή. Αλλιώς κύριε Ντράγκη, πώς δικαιολογείται με βάση τις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το γεγονός ότι η ΕΚΤ κερδοσκοπεί σε βάρος του ελληνικού λαού. Στραματίστε λοιπόν κύριε Ντράγκη να κερδοσκοπείτε κατά του φτωχοποιημένου ελληνικού λαού και των λαών του Ευρωπαϊκού Νότου. Ευχαριστώ. Well, I, I would not agree. Δεν ε, θα συμφωνήσω ότι η συζήτηση για την αναδιάρθρωση ή για την ανακούφιση είναι σωστό να γίνει τώρα. Πρέπει η Ελλάδα να στοχεύσει ακόμα στις μεταρρυθμίσεις για να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά της και η πραγματικότητα δείχνει ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές αρχίζουν και αποδίδουν και τα ευεργετήματα είναι όλο και μεγαλύτερα. Στο τρίτο τρίμηνο φάνηκε στην έκθεση σημαντική πρόοδος. Φαίνεται λοιπόν καθαρά ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε σωστή πορεία, σε σωστή πορεία και εκπληρεί τους στόχους για τα επόμενα χρόνια. Τα κέρδη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας έχουν επανέλθει μέσω των εθνικών τραπεζών και μέσω ημών στην Ελλάδα. Σας ευχαριστώ. Έχω και άλλο χρόνο Έχω και άλλο χρόνο στο σλότ Σας ρώτησα κάτι πολύ απλό. Για φέτος η Ελλάδα θα πληρώσει 10 δισεκατομμύρια στα ομόλογα της ΕΚΤ. Με την πρόταση που σας κάνω θα πρέπει να πληρώσει η Ελλάδα μόνο 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή τα χρήματα που έβαλε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τα υπόλοιπα τέσσερα δισεκατομμύρια μπορούν να αξιοποιηθούν από την Ελλάδα για το χτύπημα της ανεργίας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σας έθεσα πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα με συγκεκριμένους αριθμούς. Γιατί συνεχίζετε λοιπόν να καλύπτετε και να δέχεστε την κερδοσκοπική πολιτική της ίδιας τη Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ευχαριστώ λέτε και πάλι ότι πρέπει να αναδιαρθρωθεί το χρέος. Δεν θεωρούμε ότι είναι το σωστό πράγμα να γίνει και δεν θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο και δεν, δεν θεωρούμε ότι θα είναι και χρήσιμο. Μακάρτι, όχι με συγχωρείτε, Πέτερ Γέσεκ από τους Ελευθέρους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στο ιστορικό της ποσοτικής διευκόλυνσης φαίνεται να εμφανίζονται κάποιες ανησυχίες σχετικά με τη δυνατότητα των χωρών μελών να προχωρήσουν σε εξυγίανση των ε, δημοσίων οικονομικών τους και ε, να κάνουν σχετικές μεταρρυθμίσεις. Από την άλλη μεριά, χώρες με μεγαλύτερο φορολογικά περιθώρια φαίνεται να είναι επιθυμούν ε, να κάνουν παραγωγικές επενδύσεις. Ίσως το δεύτερο ωστόσο βραχυπρόθεσμα να είναι πιο ενισχυτικό, διότι η ανάπτυξη δεν θα προκύψει αυτόματα καθώς έρχεται και ο χειμώνας, πρέπει να δημιουργηθεί για να, και να διατηρηθεί. Λαμβάνονται και μέτρα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αυτά δηλαδή της ε, πιστοτικής διευκόνησης, Άκουσα, άκουσα την δήλωσή σας σχετικά με την ομοφωνία και βέβαια η ομάδα Άλτε θεωρεί την συνοχή μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σημαντική και την ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας απαραίτητη. Ποιο είναι το μήνυμά σας για αυτά τα θέματα που κατά κάποιο τρόπο συνδέονται. Πρόεδρος δεν κατανόησα απόλυτα το νόημα της ερωτήσεώς σας. Για να το πω πιο συγκεκριμένα. Μέτρα υπάρχουν ακόμη στον αγωγό για το quantitative easing. Ίσως ορισμένα τα μέτρα αυτά να αποθαρρύνουν ορισμένες χώρες να εξηγιάνουν τα δημόσια οικονομικά τους και μπορεί να αποθαρρύνει και ορισμένες που έχουν περισσότερα διαθέσιμα να επενδύσουν. Πρόεδρος. Το επιχείρημα ότι η νομισματική πολιτική στερεί τα κίνητρα από τις κυβερνήσεις των χωρών μελών να κάνουν τα σωστά πράγματα, είτε πρόκειται για εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών, είτε πρόκειται για επενδύσεις κλπ. Έχει ακουστεί συχνά. Η απάντηση στο επιχείρημα αυτό έχει βέβαια κάποια σκέλη. Το πρώτο είναι ότι ειλικρινά εμεί έχουμε στο κάτω τη γραφή την εντολή μα και η εντολή μας είναι η διατήρηση σταθερότητα των τιμών και αυτό σημαίνει τώρα να επανέλθει ο πληθωρισμό λίγο κάτω από το 2%. Αλλιώς αρχίζουμε να εξαρτώμεθα από τις κυβερνητικέ δράσει. και εμείς θέλουμε να διατηρήσουμε την ανεξαρτησία μας της νομισματικής πολιτικής. Επομένως, νομικά αλλά και κατά την έννοια τα δύο, τα δύο αυτά ε, θέματα είναι ξεχωριστά. Όμως και ουσιοδός είναι αλήθεια ότι οι κυβερνήσεις δεν έδρασαν ή δεν αναλαμβάνουν δράση διότι τους έχουμε περιχύσει με τόσο πολύ χρήμα που έχασαν το ενδιαφέρον τους να κάνουν οποιαδήποτε μεταρρύθμιση. Εάν εξετάσουμε τα πρόσφατα στοιχεία, αυτό δεν είναι απόλυτα σωστό. Είδαμε χώρες να μεταρρυθμίζουν τις αγορές εργασίας των και με πολύ χαμηλά επιτόκια. Υπάρχει ένα σύνολο μεταρρυθμίσεων που πραγματικά δεν έχουν σχέση με την νομισματική πολιτική. Όλες οι μεταρρυθμίσεις που έχουν σχέση με το πολιτικό σύστημα ή με τα συστήματα υγείας και ούτω καθεξής. Αλλά υπάρχει ένας τομέας όπου η σχέση αυτή μεταξύ νομισματικής πολιτικής και κινήτρων ίσως έχει κάποια αιτιολόγηση και αυτό είναι ο δημοσιονομικός, ο τομέας του προϋπολογισμού. Ίσως υπάρχει κάποια διασύνθεση μεταξύ των ε, εξοικονομήσεων μπορεί να κάνει η χώρα στη βάση των χαμηλών επιτοκίων και στην οικονομική πολιτική που ασκεί. Κατά τα άλλα δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλά στοιχεία που να δείχνουν ότι οι χώρες καθυστερούν τα μέτρα για την ολοκλήρωση της νέας αγοράς, για παράδειγμα, επειδή τα ε, επιτόκια είναι πολύ χαμηλά ή και πολύ ψηλά ενδεχομένως. Μακάρτι, ενωτική αριστερά. Κύριε Ντράγκη, πρόσφατα η Κεντρική Τράπεζα έδωσε στη δημοσιότητα επιστολές μεταξύ του κυρίου Τρισέ και του πρώην Ιρλανδού Υπουργού, Υπουργού Οικονομικών. Θα ήθελα να, ρωτήσω να κάνω ορισμένες ερωτήσεις σχετικά με τις επιστολές αυτές. Πρώτα, Μάρτιο και Μάιο φέτος η Κεντρική Τράπεζα δήλωσε κατηγορηματικά ότι δεν πιστεύει ότι θα είναι ορθό να δημοσιοποιηθεί αυτή η αλληλογραφία. Τι άραγε, άλλαξε στο, μεταξύ, ποιες συζητήσεις προηγήθηκαν και έγιναν συζητήσεις με το Υπουργείο Οικονομικών στο Δουβλίνο και ποια, ήταν η φύση των συζητήσεων αυτών και σε ποιο χρονικό πλαίσιο έγιναν. Σε μία από τις επιστολές στον, προς τον Υπουργό Brian Λέναν του Οκτωβρίου του 2010 ο τότε πρόεδρός σας Jean-Claude Trichet δηλώνει ότι εκτιμά την δέσμευση της Ιρλανδικής κυβερνήσεως σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να προωθήσει μια μακροπρόθεσμη δημοσιονομική πολιτική. Τι είδους διαβουλεύσεις είχαν ήδη γίνει στο χρονικό εκείνο σημείο. Γνωρίζετε λεπτομέρειες, γνωρίζετε πότε άρχισαν οι συζητήσεις εκείνες. Και θα ήθελα να ρωτήσω εγώ ξεχωριστά, εάν γνωρίζετε, εάν πριν από την αποστολή των επιστολών αυτών είχε προηγηθεί μελέτη των ενδεχομένων επιπτώσεων, από πλευρά τη ΕΚΤ δηλαδή, μελέτη των επιπτώσεων που θα, είχαν, ε, που θα είχε άσκηση τη πολιτική αυτή από την Ιρλανδική κυβέρνηση. Και αν γνωρίζετε τα αποτελέσματα τέτοιων εκτιμήσεων, και δέχεστε ότι τώρα ότι ήταν σφάλμα της Κεντρικής Τράπεζας η πολιτική που υπαγόρευσε τότε στην Ιρλανδική κυβέρνηση και η αναδρομική ανακεφαλαίωση, η ανακεφαλαιοποίηση των Ιρλανδικών τραπεζών αν ήταν ρεαλιστική όχι και αν γνωρίζετε αν η Ιρλανδική κυβέρνηση προτίθεται να υποβάλει σχετική αίτηση και στην περίπτωση αυτή ποια θα ήταν η στάση της Κεντρικής Τράπεζας. Σας ευχαριστώ. Ε, κάνατε πολλές ερωτήσεις. Ελπίζω να μπορέσω να σας απαντήσω σε όλες. Πρώτη ερώτηση, γιατί αλλάξαμε γνώμη. Δεν αλλάξαμε γνώμη στην πραγματικότητα. Είπαμε στην αρχική επιστολή ότι όσο γινόταν η αξιολόγηση η δημοσιοποίηση της αλληλογραφίας εκείνης μπορούσε να οδηγήσει σε κάποια ε, αποσταθεροποίηση, οικονομική αποσταθεροποίηση. Γι' αυτό και περιμέναμε. Σχολιάζω τα άλλα θέματα που αναφέρατε. Είναι πολύ σημαντικό να υπενθυμίσω ότι πριν από την έτσι Ιρλανδίας να μπει στο πρόγραμμα Βεβαίω, και η δημοσιοποίηση ολόκληρη της αλληλογραφίας μεταξύ του πρώην Προέδρου της κεντρική Τράπεζας και του πρώην Υπουργού Οικονομικών περιλαμβάνει τα στοιχεία αυτά με τρόπο σύντομο. Δεν ήταν λοιπόν η ίδια η επιστολή, αλλά πρώτα η κυβερνητική εγγύηση των υποχρεώσεων των τραπεζών. Δεύτερον, η έκταση της κρίσης. Τρίτο, οι εξωτερικοί παράγοντες που οδηγούσαν σε επιδείνωση της κρίσης. Και τέταρτο, η απώλεια εμπιστοσύνη των αγορών, που καθιστούσε αναπόφευκτο η Ιρλανδία να ζητήσει να μπει σε πρόγραμμα στήριξης. Σε ό,τι αφορά το ρόλο του ευρωσυστήματος, τονίζω ότι για πολλά χρόνια πριν από την έναρξη του προγράμματος προσαρμογής Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, καθώς και στην περίοδο αμέσως μετά, το επίπεδο ρευστότητας που πρόσφερε το ευρωσύστημα για στήριξη του Ιρλανδικού τραπεζικού συστήματος ήταν σε εξαιρετικά ύψη. Τη στιγμή που απεστάλλει η επιστολή την οποία συζητούμε τώρα, ήταν περίπου της τάξης του 85% του Ιρλανδικού ακαθάριστου εθνικού προϊόντος και ένα τέταρτο τη συνολική χορήγηση ρευστότητα από, το από, την, από το σύστημα. Το τέταρτο συνολικά το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας πάντοτε τήρησε τα όρια των, της εντολής του και τους κανόνες για το σύνολο της ε, ζώνης ευρώ. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και όρια στην στήριξη που μπορεί να προσφέρει το ευρωσύστημα σε τράπεζες των χωρών μελών. Και τα όρια αυτά καλύπτονται από τους γενικά αποδεκτούς κανόνες και υπενθυμίζονται στην επιστολή του πρώην Προέδρου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας με ημερομηνία 15 Δεκάτου 2010 προς τον πρώην Υπουργό Οικονομικών. Αρχάς Νοεμβρίου 2010 και όπως διαλαμβάνεται στην επόμενη επιστολή την οποία στέλνει ο τότε Υπουργό Οικονομικών στον πρώην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Άπεδας 4 Νοεμβρίου 2010 η κατάσταση στην Ιρλανδία ήδη έχει επιδεινωθεί σημαντικά και ταχύτατα και το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας είχε καθήκον να αντιμετωπίσει την κατάσταση αυτή. Συνεπώς, η επιστολή, η επιστολή στην οποία αναφέρεστε, αποστέλλεται από τον πρώην πρόεδρο της Κεντρικής Τράπεζας, τον πρώην Υπουργό Οικονομικών, στις 19 Νοεμβρίου πλέον 2010 και στην απάντησή του του Νοεμβρίου 21 της 21ης Νοεμβρίου, ο Υπουργός Οικονομικών της Ιρλανδίας δηλώνει ότι κατανοεί απολύτως τις ανησυχίες που αναφέρει στην επιστολή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ντράγκη στα Ισπανικά. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Γι' αυτό το τελευταίο που μόλις αναφέρατε θέλω να αναφερθώ και εγώ στις επιστολές αυτές που δημοσιεύτηκα σε σχέση με την Ιρλανδία. Για την ομάδα μου, και αυτό είναι το βασικό κύριε Ντράγκη, αυτό που έγινε δεν ήταν διάλογος μεταξύ της κυβέρνησης και της τράπεζας, της Βουβακής Κεντρικής Τράπεζας, όπως το παρουσιάσατε. Κατά τη γνώμη μου ήταν μια απειλή για κάθε κανόνα ε, γιατί ουσιαστικά εκβιάσατε την Ιρλανδική κυβέρνηση ότι δεν θα βοηθήσετε αν δεν δεχτούν. Αυτό ξεπερνάει την εντολή όμως, όπως συμβαίνει συχνά με την τράπεζα. Κάτι το οποίο οδηγεί σε μεγάλη ανησυχία την κοινή γνώμη για τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεστε τα ζητήματα αυτά και πολλούς από εμά εδώ που θέλουμε να ενημερωνόμαστε και όχι τόσο αργά. Λοιπόν, έχω να σα δώσω το εξή. Πρώτον, όσον αφορά το 2010 και τι συνεδριάσει τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, βάσει ποιου άρθρου του καταστατικού τη Τράπεζα δράσατε προκειμένου να αναγκάσετε την Ιρλανδία να ζητήσει οικονομική ενίσχυση. Γιατί εγώ δεν νομίζω ότι έχετε τέτοια εντολή. Δεύτερον, θα ήθελα να μου πείτε αν θεωρείτε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ε, προχωράει σε όλε αυτέ τι δράσει έχοντα τη στήριξη τη κοινή γνώμη ή όχι. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ντάγκη, συγγνώμη, η ερώτησή σας ποια ακριβώς είναι. Η ερώτηση είναι με ποια ιδιότητα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ζήτησε είπε στην, Ευρωπαϊκή, στην Ιρλανδική κυβέρνηση ότι θα πάρει βοήθεια εφόσον ε, το ζητήσει κάτω από τους όρους που ζητήσατε εσείς. Θα σας ξαναδιαβάσω την ε, επιστολή, την απάντηση που έδωσα και πριν. Όταν στηρίζεται με 85% ρευστότητα σε σχέση με το ΕΠ της χώρας, ένα τέταρτο της ρευστότητας στο σύνολο του ευρωσυστήματος, η Ευρώπη θέλει να είναι σίγουρη ότι δεν υπάρχει συστημική απειλή για τη σταθερότητα ολόκληρου του ευρωσυστήματος. Δεν νομίζετε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα έπρεπε να ανησυχεί επ' αυτού. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λοιπόν όφιλε να ζητήσει να εφαρμοστούν οι πολιτικές εκείνες οι οποίες θα διασφάλιζαν ότι η κατάσταση σιγά σιγά θα σταθεροποιότανε. Δεν νομίζετε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει χρέο απέναντι στι υπόλοιπε χώρε που δίνουν, προσφέρουν τη ρευστότητα αυτή να το κάνει. Αυτό ακριβώ έκανε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Σα ε, τα παρουσίασα πριν όλα τα βήματα δεν ήταν κάτι ανορθολογικό από πλευράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ούτε καμιά αυταρχική πράξη. Αποτελεί μέρος ενός συνολικού πολιτικού διαλόγου ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τις Ιρλανδικές Αρχές. Οι Ιρλανδικές Αρχές κάποια στιγμή ζήτησαν πρόγραμμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Μεσματικό Ταμείο. Πρόεδρος. Α, συνεχίζει με την ερώτηση του Ευρωβουλευτή. Κύριε Ντράγκη, μια που έχω λίγα λεφτά ακόμα στη διάθεσή μου, όσον αφορά το στόχο τώρα που αφορά τον πληθωρισμό. Κύριο στόχο είναι η σταθερότητα τιμών τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αλλά ε, επαφείεται στο Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει το ακριβέ ε, επίπεδο, αν θα είναι κάτω από το 2% και πόσο κάτω από 2%. Στο σημερινό πλαίσιο, και σε σχέση με το στόχο της συνθήκης είναι κάτι το οποίο μπορεί να τροποποιηθεί και έχει συζητηθεί καθόλου αυτό στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ντράγκη, όχι. Δεν υπάρχει περίπτωση να τροποποιηθεί. Δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο. Θα παραμείνει αμετάβλητο. Μάρκο Τζάνι τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, τρεις ερωτήσεις έχω, παρακαλώ. Πρώτη, έχει να κάνει με το σκάνδαλο των φοροποφυγών στο Λουξεμβούργο, το LuxLeaks όπως το είπαμε και η εποπτεία των μεγάλων ευρωπαϊκών τραπεζών. Ποια είναι η γνώμη σας για το σκάνδαλο αυτό, μια που η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα χρησιμοποιεί τα προγράμματα αυτά μαζικά, τα οποία επιτρέπουν να αποφεύγονται ε, φόροι από τα κέρδη αυτά. Τι θα μπορούσε να γίνει για να αποφευθεί το φαινόμενο αυτό και τι θα μπορούσε να κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Έρχομαι τώρα και στις δοκιμές αντοχής των τραπεζών και στην ανάλυση το, της ποιότητας του ενεργητικού έγιναν, αλλά σε μερικές περιπτώσεις τα αποτελέσματα δεν ήταν ικανοποιητικά. Ποια είναι η γνώμη σας, λοιπόν, τι πιστεύετε για τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε στις δοκιμές αυτές αντοχής και στην αξιολόγηση της ποιότητας του ενεργητικού. Η μεθοδολογία αυτή ε, μήπως δεν έλαβε υπόψη τους κινδύνους που ελοχεύουν ε, αναφέρομαι ιδιαίτερα εδώ στα χρηματοοικονομικά παράγωγα. Δεν πιστεύετε ότι άπαξ και καλυφθεί το ε, κενό όσον αφορά τα κεφάλαια ότι η Ευρώπη θα έπρεπε να μπορεί να αντισταθεί σε νέε κρίσεις στη Lehman Brothers. Σύμφωνα με την άλλη ανάλυση είναι σωστό να πούμε ότι μια τράπεζα όπως η Deutsche Bank ηχμένη σε χρηματοοικονομικά παράγωγα με 75 δισεκατομμύρια ευρώ είναι σωστό να πούμε ότι δεν εκτίθεται τόσο ή δεν είναι τόσο επικίνδυνη όσο μια μικρή τράπεζα όπως είναι η Κόμετ Σαν Και τι πιστεύετε για τη δημιουργία ενός δημοσίου οργανισμού παρόμοιο με αυτόν που έχουν Ηνωμένε Πολιτείε μετά το 2008 που θα μπορούσε κάθε τρεις μήνες να υποβάλει έκθεση με εκτιμήσεις όσον αφορά την έκθεση σε χρηματοπιστωτικά παράγωγα από πλευρά των Ευρωπαϊκών Τραπεζών. Τέλος για το ευρώ. Πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες είναι αλήθεια ότι δεν είναι πλέον ενθουσιώδεις όσον αφορά το ευρώ και κάποιες χώρες κάποια μέρα θα αποφασίσουν μονομερός να φύγουν από την Ευρωζώνη. Στι 25 Μαΐου ψήφισαν οι Ευρωπαίοι πολίτες για κινήματα και κόμματα που είχαν στο πρόγραμμά τους είτε δημοψήφισμα είτε έξοδο από το ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πιστεύει ότι μπορούμε να καλύψουμε το νομοθετικό κενό που υπάρχει όσον αφορά την έξοδο από το ευρώ, να μπορεί να δημιουργήσει δηλαδή μηχανισμούς που θα επιτρέπουν στις χώρες μέλη που το επιθυμούν να φύγουν δημοκρατικά από το ευρώ. Στην ακρόασή του ο κύριος Δομπρόφσκι που θα ασχοληθεί με το ευρώ είπε ότι εάν μια χώρα θέλει να βγει από το ευρώ, κανένα δεν μπορεί να την εμποδίσει και ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα βοηθήσει τεχνικά. Αλλά όλα αυτά διαψεύστηκαν την επόμενη μέρα μέσω ε, ενό δελτίου τύπου. Ποια είναι η δικιά σα άποψη από αυτού. Ευχαριστώ, λέει ο κύριο Δράγκη. Θα δούμε σιγά σιγά τις ερωτήσεις σας. Πρώτα απ' όλα όσον αφορά το LuxLeaks. Δεν έχουμε εμεί κανένα ρόλο έχει να κάνει με τη φορολογική ε, ενιοποίηση, έχει να κάνει με την αναρμόνιση μάλλον τη φορολογική. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μπορεί να έχει πολλές εξουσίες, αλλά το φορολογικό δεν το έχει. Δεύτερον, όσον αφορά τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε στα τεστ αντοχής και στην συνολική αξιολόγηση. θα σχολιάσω ίσως και αργότερα από αυτού. Συνολικά πάντως η αξιολόγηση ήταν μια αξιόπιστη άσκηση που καλύπτεται από πλήρη διαφάνεια και είναι κάτι το οποίο καλοδέχτηκε ένα μεγάλο μέρος, το μεγαλύτερο μέρος της κοινή γνώμης, θεώρησε ότι πρόκειται για μια πρόοδο προκειμένου να ενισχυθεί ο συλλογισμός των μεγάλων ευρωπαϊκών τραπεζών της Ευρωζώνης. Από αυτή την άποψη λοιπόν θα φέρει πολλά ωφέλη. Ένα από αυτά είναι όντω την ενίσχυση της εφαρμογής της νομισματικής μας πολιτικής. Από την άλλη μεριά όμως θα αποτελέσει και μια πολύ καλή βάση για την βελτίωση της ρευστότητας μέσα στους επόμενους μήνες. Τώρα, κατά πόσο κερδίσαμε τον πόλεμο και τελείωσε... Η ερώτησή σας μπορεί να τεθεί και διαφορετικά. Μπορούμε να πούμε έχουμε ε, συνθήκες ε, απόλυτα ισότιμες όσον αφορά το τραπεζικό τομέα παντού. Ε, η απάντηση είναι όχι. Έχει επιτεθεί μεγάλη πρόοδος, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο και θα σας δώσω κάποια παραδείγματα. Πρώτον, γιατί δεν έχουμε ίσους όρους παντού. Γιατί σε διαφορετικές χώρες έχουμε διαφορετική νομοθεσία. Πρόκειται για εθνική νομοθεσία η οποία αναγνωρίστηκε από τον Ευρωπαίο νομοθέτη. Οπότε προς το παρόν αυτή είναι η κατάσταση, αυτή η νομοθεσία ισχύει και η συνολική αξιολόγηση έπρεπε να το λάβει αυτό υπόψη. Παραδείγματα. Η μεταχείριση του goodwill, treatment of goodwill, ή τρίτα περιουσιακά στοιχεία είναι μερικά παραδείγματα. Και έχουμε και σε εσά εναρμόνιση των ε, κινδύνων περιουσιακά στοιχεία ή ισότιμη μεταχείριση ε, εσωτερικών μοντέλων. Συνεπώς χρειάζεται επιπλέον δουλειά προκειμένου να πετύχουμε ισότιμους όρους και το SSM, η κυρία Νουγή και η κυρία Λάντους Λέγερ και ολόκληρο το Διοικητικό Συμβούλιο του Ενίου Αποπτικού Μηχανισμού έχουν δεσμευτεί όπως έχουν πει και ξαναπεί επανειλημμένως. Φτάνουν αυτά για να αποφύγουμε οποιαδήποτε μελλοντική κρίση που θα μας έρθει από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Όχι βέβαια. Ασφαλώς όχι. Κάναμε πολλή δουλειά για να ξεπεράσουμε την οικονομική κρίση. Οι προπτικές δεν είναι ας μαντέψουμε ποια θα είναι η επόμενη κρίση και να δουλέψουμε βάση μια τέτοια επόμενη κρίση, Όχι, αυτό που θέλουμε να κάνουμε και γι' αυτό δουλέψαμε είναι για να κάνουμε πιο ανθεκτικό το σύστημα. Αν λοιπόν έρθει μια άλλη κρίση, το σύστημα θα είναι ισχυρότερο. Είμαι όμως απολύτως σίγουρος ότι το σύστημα ήδη τώρα μάλλον μπορώ όμως να σας πω ότι δεν μπορούμε 100% να είμαστε σίγουροι ότι θα έχει πλήρη ασυλία από οποιαδήποτε μελλοντική κρίση το σύστημα. Πάντως χρειάζεται παραπάνω δουλειά. Γι' αυτό ακριβώς και γι' αυτό η δράση μας επικεντρώνεται στην ρύθμιση του τραπεζικού συστήματος. Όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει βέβαια και το σκιώδες τραπεζικό σύστημα, το οποίο εξελίσσεται επίσης πολύ γρήγορα. Το επόμενο τώρα ερώτημά σας ήταν για την Deutsche Bank. Δεν σχολιάζω για επιμέρους τράπεζες. Όσον αφορά το ευρώ, Είσαστε πεπισμένος από ό,τι φαίνεται, για σας είναι σαφές, όχι όμως και για μένα, ότι κάποιες χώρες θα θελήσουν να φύγουν από το ευρώ. Όσον αφορά εμάς, βεβαίως. Πρώτον, δεν έχουμε νομοθετικές εξουσίες. Έχουμε αρκετές εξουσίες. Αν θέλετε να μας αναθέσετε και νομοθετικές εξουσίες για να αποφασίσουμε αν μια χώρα θα βγει ή δεν θα βγει από το ευρώ, Ίσως, αλλά δεν έχουμε τέτοιες εξουσίες τώρα. Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το έχω πει και ξαναπεί ότι το ευρώ είναι μη αναστρέψιμο και ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα κάνει ό,τι χρειάζεται στα πλαίσια της εντολής της. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος. Ο κ. Ντομπρόσκης έκανε σαφέστατη δήλωση σχετικά με την θέση του για την ε, ακαιρεότητα της Ευρωζώνης η οποία δεν είναι επιστρεπτή. Αυτά για τον κύριο Τομπρόσκη. Κύριε Μπάρμπαρα Κάπελ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε Ντράγκη, από τα πιο αμφισβητούμενα μέτρα που έχουν ληφθεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τη σταθεροποίηση των, ε, των αγορών ήταν και το πρόγραμμα του Αυγούστου 2012 και τον επόμενο χρόνο. Με την αγορά κρατικών ομολόγων υποτίθεται ότι προσφέρεται στήριξη και αυξάνεται ο ισολογισμός της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε 3 εκατομμύρια Δεν συμφώνησαν όμως όλες οι χώρες και δεν ακολούθησαν οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις σε όλες τις χώρες μέλη σύμφωνα και με έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πολλές χώρες δεν προβαίνουν στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Ερώτηση. Συμφωνείτε μαζί μου ότι η αγορά κρατικών ομολόγων από πλευρά κεντρικής τράπεζας από χώρε οι οποίες αποδείχνονται απρόθυμες να προβούν στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις δίνει εσφαλμένε εντυπώσεις και κίνητρα με την έννοια ότι δεν εφαρμόζουν τις μεταρρυθμίσει οι χώρες στον ε, τομέα του προπολογισμού, διότι μπορούν να έχουν φθηνότερο χρήμα για να εκπληρώνουν τις υποχρώσεις τους. Ο κλάδος έχει τελικώς αναλάβει περισσότερες υποχρώσεις. Για την υλοποίηση της ε, ε, Τραπεζικής Ένωσης για το μέλλον θα σημαίνει ότι τα, και τα ε, οι ευρωπαϊκές τράπεζες θα πρέπει να έχουν πολύ μεγαλύτερες ζώνες προστασίας, buffer δηλαδή, με χρήμα το οποίο θα λαμβάνουν από αλλού, από τον ιδιωτικό τομέα. Θα υπάρξουν αρνητικές συνέπειες για τη Βασιλεία 3 και για τις τράπεζες. Θα υπάρξει αρνητική επίπτωση στη χρηματοδότηση των μικρών και μεσών επιχειρήσεων. Λαμβάνει μέτρα, υποτίθεται να λάβει μέτρα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τη βελτίωση χρηματοδότηση των μικρών και μεσών επιχειρήσεων. Για την πρώτη σας ερώτηση, μεταξύ Ιουνίου και Σεπτεμβρίου, όπως είπα και στην αρχική μου ομιλία, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έλαβε πληθώρα μέτρων και για ε, την ε, αγορά κρατικών ομολόγων και ABS. Είμαστε πεπισμένοι ότι με τα μέτρα αυτά βοηθήσαμε στον να σταθεροποιηθεί πληθωρισμός και αναμένουμε ότι θα έχουμε αρκετά μεγάλη επίπτωση στον ισολογισμό μας που θα τίνει να φτάσει στο ύψος που είχε το Μάρτιο του 2012. Τούτου λεχθέντος, εάν τα μέτρα αυτά αποδειχθεί ότι δεν είναι επαρκή έτσι ώστε ο αναμενόμενος πληθωρισμός να φτάσει σχεδόν στο 2% ή ενδεχομένως και να αντιμετωπιστεί και επιδίνωση του προσδοκόμενου πληθωρισμού ή αν ο πληθωρισμός αρχίσει να επιδεινώνεται από μόνος του, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι διατεθειμένο και πανέτοιμο να αναλάβει δράση. Είπα και πριν ότι είναι ομόφωνο στο να αναλάβει και άλλα μη συμβατικά μέτρα πέραν των μέτρων που έχουν ήδη αποφασιστεί. Και είναι και διατεθειμένο να αναλάβει δράση. Με την έννοια ότι στην τελευταία του συνεδρίαση ζήτησε από το προσωπικό της Κεντρικής Τράπεζας αλλά και από τις ε, σχετικές επιτροπές που απαρτίζονται από προσωπικό των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών να μελετήσουν τα σχετικά συμβατικά, α, μη συμβατικά μέτρα. Ε, τούτου λεχθέντος έχουμε και μια εντολή. Η εντολή λέει ότι ο στόχος του πληθωρισμού θα πρέπει να φτάνει το πολύ στο 2%. Εμεί, και απάντησα και σε άλλη ερώτηση σχετική προηγούμενα, θα εξετάσουμε τι γίνεται σε άλλε χώρε Αυτό είναι ξεχωριστό. Το εάν έχουν κίνητρα για να προχωρήσουν ή όχι είναι σημαντικό. Αλλά δεν είναι ζήτημα το οποίο άπτεται τη εντολή μα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν έχει δημιουργηθεί για να εξασφαλίσει ότι οι κυβερνήσει θα πράττουν το σωστό. Το γνωρίζουμε. Είναι σημαντικό για την αποτελεσματικότητα τη νομισματική μα πολιτική. Όπω είπα και πριν, τα μέτρα μας έχουν το σκοπό να κάνουν τη συμβατική πολιτική πιο αποτελεσματική, αλλά όπως είπα περιοριζόμαστε από την εντολή μας. Άλλα μη συμβατικά μέτρα μπορούν να σημάνουν και την αγορά άλλων προϊόντων και ενδεχομένως και κρατικών ομολόγων. Ο κύριος Κύριε Πρόεδρε, είπατε και το επαναλάβατε τώρα ότι η νομισματική πολιτική από μόνη της δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματα. Μιλήσατε για διαφορετικές αλλαγές, μεγαλύτερη παραγωγικότητα και ούτω καθεξής. Σωστά είναι αυτά σίγουρα. Όμως η κοινή γνώμη συζητεί και άλλα θέματα που δεν ε, έχουν απαραίτητα σχέση με το παρελθόν αλλά με το μέλλον. Για παράδειγμα, συζήτηση την οποία ξεκίνησε η κυρία Λαγκάρντ και σας θέτω και εγώ εσά το ερώτημα και παρακαλώ να απαντήσετε. Δεν θεωρείται αναγκαίο να αναθεωρηθούν οι κανόνες του 1995 που οδήγησαν σε αύξηση του χρέους κατά 25% παγκοσμίω. Κάτι που σημαίνει ότι και η νέα χρέωση δεν θα πρέπει το περιθώριο να αυξηθεί και το περιθώριο, περιθώριο του νέου χρέους να μειωθεί. Και βάζω εδώ και το ζήτημα του πληθωρισμού. Θέλει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να ασκήσει πολιτική αντίθετη με τις πραγματικά μειούμενες τιμές του πετρελαίου και άλλων πρώτων υλών. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση τώρα. Η ποσοτική χαλάρωση και τα άλλα μέτρα που λάβατε δεν οδήγησαν σε επιτυχία τώρα. Η κοινή γνώμη συζητεί με την ανάληψη κινδύνων από τις τράπεζες και την ελάφρυνση των κυβερνήσεων, η κεντρική τράπεζα ενδεχομένως θα, καταστεί, θα να είναι bad bank. Η ρευστότητα, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι τόσο το πρόβλημα, αλλά ενδεχόμενα υψηλότερε απαιτήσει. Και τέλος, η πιο πρόσφατη πρόταση που ακούστηκε τούτο το Σαββατοκύριακο, για την απομάκρυνση για το, για το μεγάλωμα του χάσματος ευθύνονται κυρίως οι μισθοί. Εδώ υπάρχουν μόνο τρεις δυνατότητες. Πληθωρισμός, αποπληθωρισμός ή μείωση της αξίας του νομίσματος, κάτι το οποίο αποκλείεται βεβαίως. Άρα τώρα υποτίθεται ότι θα πρέπει να εγκριθεί ένας μηχανισμός Αντισταθμιστικό. Εσεί τι γνώμη έχετε γι' αυτό. Νομίζω ότι κατανόησα δύο από τις τρεις ερωτήσεις. Δεν είμαι βέβαιος ότι κατανόησα καλά την τρίτη. Να προσπαθήσω να απαντήσω στο πρώτο πάντως. Οι κανόνες μας είναι αυτοί που θεμελιώνουν την εμπιστοσύνη και επομένως πρέπει να τηρούνται και συγγράφηκαν περιλαμβάνοντας και ένα στοιχείο ευελιξίας ή ευκαμψίας με το οποίο μπορούν να εφαρμοστούν. Ας αναρωτηθούμε ποια πράγματα πήγαν στραβά το 2003 και το 2005. Άλλαξαν οι κανόνες λόγω του συμφέροντος ορισμένων χωρών των και όχι μέσα από μια συλλογική κοινωτική διαδικασία. Οι αλλαγές στους κανόνες οδήγησαν σε χρέωση, έτσι ώστε όταν ξέσπασε η μεγάλη οικονομική κρίση, ήδη τα επίπεδα του χρέους ήταν πολύ υψηλά και ανέβηκαν κι άλλο μετά από το ξέσπασμα της κρίσης. Το θέμα λοιπόν εδώ είναι θα πρέπει να ανατρέψουμε τους κανόνες συνολικά όπως φαίνεται να προτείνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και να ξαναρχίσουμε μια συζήτηση από την αρχή ή θα πρέπει απλώ να τηρήσουμε τους κανόνες θεωρώντας ότι είναι σημαντικότερο για να υπάρξει αμοιβαία εμπιστοσύνη και αξιοπιστία να τηρούμε και να σεβόμαστε του κανόνε. που όπω είπα είναι γραμμένοι με αρκετή προσοχή. Η Κεντρική Τράπεζα τάσσεται μάλλον υπέρ της δεύτερη επιλογής. Η Κεντρική Τράπεζα δεν επιθυμεί να προχωρήσει μια συζήτηση που θα αλλάξει όλους τους κανόνες άρδιν. Εξάλλου δεν είμαι βέβαιος ότι συμφωνώ μαζί σας όταν λέτε ότι η νομισματική μας πολιτική δεν απέδωσε. Εγώ θα έλεγα μάλιστα το αντίθετο. Η νομισματική μας πολιτική απεδείχθη εξαιρετικά επιτυχής. Όλα μας τα επιτόκια είναι χαμηλότερα από ό,τι ήταν Και τα χαμηλότερα από αυτά είναι χαμηλότερα και από εκείνα των Ηνωμένων Πολιτειών. Και σε, όλο, σε, σε κάθε είδους ορίζοντα, σε όλες τις ληξιμότητες. Και στην κρίση του ευρώ του 2012. Μειώσαμε τα επιτοκιά μας και έχουμε και ένα deposit facility rate που τώρα πλέον οι τράπεζες καλούνται να πληρώσουν εάν θέλουν να παρκάρουν το σαγικών τα χρήματά τους στην κεντρική τράπεζα και όχι να τα δανείσουν στην πραγματική οικονομία. Βέβαια, η νομισματική μας πολιτική πέτυχε να ξαναβάλει μπρος την πραγματική οικονομία στη ζώνη ευρώ. Απάντηση είναι όχι. Χρειαζόμαστε χρόνο έτσι ώστε τα νομισματικά αυτά κίνητρα να αρχίσουν να χαράζουν μια πορεία μέσα στην πραγματική οικονομία. Είπαμε βέβαια κατά επανάληψη ότι χρειάζονται και άλλοι δυο πυλώνες διαρθρωτικές αλλαγές και μια σωστή δημοσιονομική πολιτική. Εγώ θα έλεγα λοιπόν ότι υπήρξαμε επιτυχής από την πλευρά των αγορών, επιτυχής από την άποψη της σταθεροποίησης του τραπεζικού συστήματο, που είτε μα αρέσει είτε όχι εξακολουθούν να υπάρχουν τραπεζέ και παίζουν το διαμεσολαβητικό ρόλο στο 80% των ε, ροών στην πραγματική οικονομία. Απαντώ σε μια ερώτηση που δεν απίτησα ακριβώ πριν. Όταν είπαμε τι θα κάνουμε για να δανείσουμε περισσότερα στι μικρέ και μεσαίε επιχειρήσει, ένα από τα πράγματα που κάνουμε είναι η συνολική αξιολόγηση, comprehensive assessment. Δηλαδή, να διαπιστώσουμε, να φροντίσουμε ώστε να είναι ισχυρότερο και υγιέστερο το τραπεζικό σύστημα τώρα και να μπορεί να διαθέσει περισσότερα κεφάλαια στις ΜΜΕ. Την τελευταία ερώτηση για του πραγματικού μισθού δεν την κατανόησα, Δυστυχώ. Η τελευταία μου ερώτηση είχε το εξή νόημα. Σχετικά με τι προτάσει που προέρχονται από πολιτικού αλλά και από οικονομικού επιστήμονε, ότι η απροθυμία μεταρρυθμίσεων σε ορισμένε χώρες μέλη δεν αντιμετωπίζεται με χαμηλότερα επιτόκια, ούτε με παρατάσεις, αν έχουν ξεπεράσει το 95%, διότι θα φτάσουν τότε στο 60% του ΑΕΠ τους ως χρέος το 2050. Ερώτηση. Υπάρχει ένας διορθωτικός παράγοντας που να είναι νοητός, που να μπορεί να προταθεί και ο οποίος να μπορεί να βελτιώσει τις σχέσεις και να τις προσαρμόσει γιατί έχουν όπως είπα συγγραφεί από το Μάιο του 1998. Απάντηση. Θα το επεξεργαστούμε και θα το συζητήσουμε. Δεν έχουμε άποψη για την ώρα επ' αυτού. Για το εάν η νομισματική μας πολιτική τώρα στερεί τα κίνητρα από τις χώρες μέλη για να κάνουν τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις και αυτό απίτησα προηγουμένως πράγματι στον δημοσιονομικό τομέα, το τομέα του προπολογισμού, δηλαδή αφού πληρώνουν χαμηλότερου τόκους, θεωρούν ίσω όντω ότι μπορούν να καθυστερήσουν μέτρα τα οποία θα μείωναν τι κρατικέ δαπάνε. Σε όλου του υπόλοιπου τομεί όμω, δεν διαθέτουμε στοιχεία που να δείχνουν ότι υπάρχει κάποιο συσχετισμό μεταξύ τη αδράνεια από τη μια μεριά και των επιτοκίων από την άλλη. Ρενάτο Σόρου. Σας ευχαριστούμε. Το λόγο έχει κύριος Σόρο. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Ε, πάντοτε είναι πάρα πολύ χρήσιμο να ξέρουμε τις απόψεις σας και να μπορούμε έτσι να έχουμε μια πιο ξεκαθαρή εικόνα για την κατάσταση και στην απάντησή σας ήδη απαντήσατε κάτι πριν σε ρωτήσω στην Ευρώπη το 80% των πόρων των επιχειρήσεων περνούν μέσα από τις τράπεζες. Θεωρείτε ότι θα μπορούσε αυτό να έχει άλλος και να έχουμε περισσότερη χρηματοδότηση κατά τον τρόπο για τις επιχειρήσεις. Επίσης, όσον αφορά την ανάλυση του Ευρωπαϊκού Τραπεζικού Συστήματος, όπως έγινε, μας κατέληξε ότι υπάρχει κεφαλουχική επάρκεια αλλά ε, δεν δίνονται αρκετά, δεν είναι στις ΜΜΕ. Γιατί τέτοιου είδους χρηματοδότηση απαιτεί μεγαλύτερη επάρκεια. Μπορείτε κάτι να κάνετε γι' αυτό. Τέλος, στη συνέχεια στο ίδιο όσον αφορά την ε, νομισματική πολιτική η οποία βοήθησε πάρα πολύ για την συρρήγνωση των επιτοκίων αλλά από μόνη της δεν αρκεί. Όπως είπατε και εσείς, μπορεί να γίνουν περισσότερο από την νομισματική πολιτική, αν έχουμε κάποιες μεταρρυθμίσεις, ούτως ώστε να είναι πιο ανταγωνιστικές οι οικονομίες. Ιδίως να γίνει κάτι για την ε, ε, αγορά εργασίας, αλλά και γενικότερα στην αγορά. Και έτσι υπάρχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη από πλευράς όλων. Όμως, χρειάζεται μια δημοσιονομική πολιτική πραγματικά κοινή. Τι γίνεται με αυτά τα 300 δις, δεν ξέρουμε πώς θα προκύψουν. Επίσης μιλούμε για τελευταίες μέρες για αυτό το νέο ταμείο επενδύσεων το οποίο μπορεί να ε, χρησιμοποιεί με πολλούς τρόπους ούτως ώστε να έχουμε τέλος κάποιες ε, επενδύσεις και του κρατικού και του ιδιωτικού τομέα. Πώς θα εμπλακεί επομένω σε αυτή την ιδέα Γιούγκερ η Ευρωπαϊκή Κοινωνική Τράπεζα. Όντως είναι κάτι το ανέκλητο το ευρώ. Αλλά τι θα γίνει με την οικονομία, τι θα γίνει με την απασχόληση. που έχουν γίνει τα πράγματα τόσο δύσκολα σε όλα αυτά τα μέτωπα σε πολλές χώρες της Ευρώπης, Σας ευχαριστώ. Η Ευρωζώνη ενδιαφέρει πάρα πολύ από ό,τι είπα. Διότι 80% των πιστώσεων περνούν μέσα από το τραπεζικό σύστημα, ενώ στις ΗΠΑ έχουμε το αντίστροφο. Έχουμε περίπου 30% ίσως και λιγότερο ε, των πιστώσεων και των δανείων που περνούν μέσα από τις τράπεζες. Τώρα, ποιο σύστημα είναι καλύτερο. Το μάθημα που έχουμε αντιλήσει από την συγκυρία τελευταία είναι ότι εάν οι τράπεζες για κάποιο λόγο βρίσκονται σε αδύναμη θέση, σε αρκετή ε, χρονική διάρκεια, σταματούν να δίνουν πιστώσεις και δάνεια. Ό,τι και να κάνει η κεντρική τράπεζα. Όσο επεκτατική να είναι η πολιτική δεν δίνονται πιστό στην πραγματική οικονομία γιατί απλά έχει στεγνώσει ο διάβλος χορήγηση δανείων. Ευτυχώ είχαμε το εξή όμω αυτή την τελευταία δύσκολη τριετία τετραετία. Είδαμε το 2011 και το 2012 και το 2013 τα δάνεια να μειώνονται πάρα πολύ, απελπιστικά πολύ. Βλέπουμε όμως τώρα ότι το, χειρότερο σημείο είναι πίσω μας και επομένως όπως έγινε αυτή η, η, αξιολόγηση οδήγησε στο να αρχίσουν να χώνονται πάλι δάνεια. Έχουμε ομόλογα που εκδίδονται έχουμε άλλα αξιόγραφα τα οποία επίσης όλα αυτά κατατείνουν στο ότι οι αγορές δηλαδή αλλά και οι εταιρείε ε, τελικά ε, αντιστάθμισαν αυτού του είδους τη μείωση των ε, δανειών της τράπεζας τελευταία τη τριετία και αυτό μας οδηγεί στις εξής σκέψεις πρώτα πρώτα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν πρόσβαση στις κεφάλαια αγορές. Άρα, όπως έχουν τώρα τα πράγματα, έχουμε χρηματοδότηση σε μεγάλες θερίες αλόγους σε ΜΜΕ. Και η ΜΜΕ είναι μεταξύ 70 και 80% της απασχόλησης στην Ευρωζώνη. Όμως, δεύτερο συμπέρασμα είναι το εξής. Θα έπρεπε η πολιτική μας να κατατείνει στο να έχουμε πιο ισχυρή κεφαλαιόρα από ό,τι σήμερα και κατά αυτόν τον τρόπο η οικονομία μας να στηρίζεται λιγότερο στις τράπεζες στο μέλλον. Η απάντηση είναι 100% καταφατική. Οπότε και συμφωνούμε με την πρόταση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να υπάρχει μια τέτοια ένωση των αγορών οπότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, να επεξεργαστούν αυτή την πρόταση κατά το επόμενο έτος. Τώρα όσον αφορά το πρόγραμμα επενδύσεων που παρουσιάζει ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, φυσικά και το θεωρούμε κάτι πολύ θετικό, αλλά δεν μπορεί σε αυτό να εμπλακεί με χρηματοδότηση η Ευρωκεντρική Τράπεζα. Θα περιμένουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει τις λεπτομέρειες και σας ευχαριστώ. Γκολτιέρη. Ευχαριστώ. Δεν το έχουμε την επόμενη ομιλήτρια. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα τράγκη. Όταν μας είπατε ότι είναι πρόθεση της τράπεζας να συνεχίσει και να, να ξεκινήσει τελικά τα EBS, τι γίνεται όσον αφορά με ναι, αυτά τα μέτρα σε σχέση με τις εγγύησεις. Και είπατε αυτά τα, αυτές οι ενδιάμεσες δόσεις θα πρέπει να έχουν εγγύησεις κρατών μελών. Έτσι είχατε αναγγείλει. Όμως, όμως, για αυτού τους εγγύησεις είδαμε ότι ελάχιστα ενδιαφέρονται τα κρατή μέλη. Επίσης είπατε ότι η ΕΚΤ συνεχίζει στην πορεία αυτή ό,τι και συμβαίνει. Εσείς τι λέτε. Τι θα κάνετε, θα συνεχίσετε πέραν του τα κράτη-μέλη δεν θέλουν τέτοιες εγγύσεις. Θα μπορούσαν τα κράτη-μέλη να υποφεληθούν από την ασφάλεια των στοιχείων των τραπεζών. Επίσης όσον αφορά την macroprudential policy, το SSM είναι ένα εργαλείο εποπτικό. Ο μηχανισμός αυτός έχει αρμοδιότητα του να θέτει και φολοχέ πιο απαιτητικέ. και επίσης και άλλα μέτρα για να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι οι μακροοικονομικοί. Άρα είναι βασικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιο είναι το μέλλον λοιπόν του SSM Ποιο είναι το μέλλον της μακροπροληπτικής πολιτικής. Ντράγκη. Νομίζω την επόμενη φορά θα συζητήσουμε για τη δεύτερη ερώτηση, αλλά για την πρώτη σας ερώτηση έχω να πω το εξής. Είπατε ότι η ΕΚΤ μπορεί να γίνει κακή τράπεζα. Δυσκολεύομαι να κατανοήσω όμως πώς προκύπτει κάτι τέτοιο. Να σας εξηγήσω τι κάνουμε. Ναι, το ABS με τα τριτλοποιημένα δάνεια. Το πρώτο το οποίο έχουμε κατά νου, να δώσουμε το ίδιο όνομα σε πράγματα όλος διαφορετικά. Στη ΣΥΠΑ τα ABS ήταν κυρίως τα subprime τέτοια δάνεια στεγαστικά τα οποία δεν υπάρχουν στην Ευρώπη. Και εάν πάρουμε επομένω όλη τη χρηματοδότηση μεταξύ 2007 και 2013 όλοι όμως τότε έχουμε 18,4% εκτόγιους ενώ εδώ έχουμε 1,5%. Άρα εδώ πέρα δίνουμε το ίδιο όνομα σε δύο διαφορετικά πράγματα. Δεν αγοράζουμε όμως ε, όλα τα τίτλοπνένα δάνεια, αλλά μόνο συγκεκριμένα. Ας πούμε τα στεγαστικά κατοικίας ε, έχουν default rate 0,1%. Καταναλωτικά δάνεια και τέτοια αγοράζουμε. 0,04% είναι το default rate αυτόν. Αλλά δεν ακούμαστε ούτε σε αυτό αγοράζουμε μόνο τα ανώτερα κομμάτια, τα ανώτερα τμήματα, όπου το default rate είναι ακόμα πιο χαμηλό. Άρα η χρήση του όρου Bank, τράπεζα για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την αδικεί. Το να πούμε το λιγότερο. Τώρα να αφορά αυτό το μέζαν είναι αυτό το ενδιάμεσο, ε, έχει κάποιο κίνδυνο αλλά όχι τον μεγαλύτερο όσον αφορά τα διτολμένα δανεία. Και γι' αυτό είπαμε ότι η ΕΚΤ e θα τα αγοράσει μόνο από τη βάση εγγύησεων, από τη βάση κάποιων ασφαλιών. Αυτό δεν έχει αλλάξει. Αυτή την πολιτική έχουμε τώρα. Ξέρω ότι εκ πρώτης όψεως οι περισσότερες κυβερνήσεις, κάποιες κυβερνήσεις αυτών είπαν ε, όχι, αλλά κάποιες ε, άλλες κυβερνήσεις είναι υπέρ. Και τα περισσότερα κράτη, αν όχι όλα, ήδη έχουν προχωρήσει προς τα εκεί, ήδη προσφέρουν εγγύσεις και ασφάλειες για το μεζανίν μέσω συγκεκριμένων ε, ταμείων παρακατοπτικών και στην ΤΕΠΟ, Κάζα την στην Ιταλία και στη Γαλλία και το διηγείται σε Ισπανία και Γερμανία. Οπότε εδώ το θέμα είναι ο συντονισμός το να μάθουμε να προχωρούμε από κοινού κλπ. Έχουμε ξεκίνησει μόνο με το ανώτερο κομμάτι των αγορών αυτών των δανείων και θα δούμε πού θα πάει. Ο κύριος Πέτερ Σιμών έχει το λόγο. Τα επιτόκια της Κεντρικής Τράπεζας τίνουν προς το μηδέν. Διαπιστώνουμε ωστόσο ότι στην πραγματική οικονομία οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις δεν λαμβάνουν τα χρήματα δεν φτάνει μέχρι εκεί, μέχρι εκεί πιστώσεις. Από πλευράς Κεντρικής Τράπεζας, τι είναι δυνατόν να κάνει η ίδια από την πλευρά της ή να προτείνει, ώστε να φτάσουν οι πιστώσεις στι στις ίδιες τις μικρές και μέσες επιχειρήσεις. Και τι θα προτείνατε σε εμά του Ευρωπαίους νομοθέτες, πέραν από τις διαφορετικές μεταρρυθμίσεις που ζητείτε από τις χώρες μέλη να κάνουν, τι άλλο μπορείτε να προτείνετε για να πληρωθεί το κενό αυτό. Δηλαδή, αφενός συχνά οι τράπεζες διαθέτουν ρευστότητα, από την άλλη μεριά δεν, είτε δεν ζητούνται είτε δεν προσφέρονται στις μικρές και μέσες επιχειρήσεις. Δεύτερη σύντομη ερώτηση, πάλι με το ίδιο ιστορικό αλλά με άλλη κατεύθυνση. Τραπεζική Ένωση. Στόχος της Τραπεζικής Ένωσης είναι να βελτιωθεί η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και να καταστεί και πιο ανεξάρτητη από την τραπεζική χρηματοδότηση. Ποια στοιχεία θεωρείτε εσείς προσωπικά ως απαραίτητα για την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης και ποιον ρόλο βλέπετε μέσα στην προσπάθεια αυτή για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρος Δράγκη, ευχαριστώ. Να πω πρώτα ότι η κατάσταση βελτιώνεται και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Υπάρχουν δύο έρευνες, αφενός αυτή που κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και αφετέρου άλλη ειδική έρευνα την οποία νομίζω κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, SFE. Αυτές δείχνουν ότι αυτές οι δύο έρευνες δείχνουν ότι όντως έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Ότι οι χρηματοδοτήσεις είναι λιγότερο σφιχτές από ό,τι ήταν στο παρελθόν, ότι η αντίληψη του κινδύνου από πλευρά του τραπεζικού συστήματος έχει βελτιωθεί σημαντικά. Βέβαια, τούτου λεχθέντος οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε και το γεγονός ότι η πίστη έχει δύο πτυχές. Ζήτηση και προσφορά. Για αυτό το λόγο, όσο ναι μεν οι περιορισμοί, και οφείλω να το πω προσεκτικά, οι περιορισμοί είναι λιγότερο σφιχτοί στις διάφορες έρευνες που έχουμε κάνει τον τελευταίο 1,5 χρόνο, εξακολουθούν ωστόσο ιστορικά να είναι σφιχτοί. Αν τους εξετάσετε μέσα σε ευρύτερο χρονικό πλαίσιο από την άλλη μεριά πρέπει να υπάρξει και κάποια ανάκαμψη της ζήτησης πίστης για επένδυση. Εκεί βλέπουμε να αργοπορούν πολύ. Βεβαίως πάντα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στις διαπιστώσεις μας. Υπάρχουν κάποια στοιχεία που δείχνουν ότι ο κύκλος αρχίζει να βελτιώνεται, αλλά δεν έχουμε δει ακόμα σαφώς τις επιπτώσεις της ΜΜΕ. Πρέπει βεβαίως να λάβουμε υπόψη και άλλα δύο πράγματα για τη ΜΜΕ. Δεν είναι εύκολο να χορηγηθούν πιστώσεις στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, διότι ιστορικά σε ορισμένες χώρες μέλη οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ιστορικά έχουν υπερβολικό leverage και είναι πολύ περιορισμένη η χρηματοδότησή τους. Εξάλλου όλες οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο. Ακόμα και στις χώρες εκείνες όπου οι ΜΜΕ παίζουν κυρίως ρόλο σε εξαγωγές τα πάνε πολύ καλά. Είναι λοιπόν πρόβλημα κυρίως, κυρίως εσωτερικής ζήτησης. Και οι ΜΜΕ που δουλεύουν για την εσωτερική ζήτηση εξακολουθούν να είναι αδύναμες. Δεν έχουν αρκετή ρευστότητα και δεν υποβάλλουν πολλές αιτήσει για χρηματοδότηση πιστεύουμε ότι η νομισματική μας πολιτική θα φτάσει τελικά μέχρι την πραγματική οικονομία. Και αυτός ο παράγοντας μαζί με άλλους όπως οι χαμηλές τιμές πρώτων υλών θα στηρίξουν την ζήτηση. Αλλά βέβαια είναι μια αργή διαδικασία όπως έχουμε δει ως τώρα. Τώρα για την ενοποίηση των κεφαλαίων ρωτήσατε ποιος θα είναι ο ρόλος της Κεντρικής Τράπεζας. Η Κεντρική Τράπεζα είναι υπέρ της μείωσης της ε, εξάρτησης ε, της Ευρωζώνης από τις τράπεζες και να ενισχυθούν ε, και να ενισχυθεί και η προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο σημαντικό αυτό τομέα. Λούντεκ Μάιερ Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Ντράγκη, σας εύχομαι καλή επιτυχία στη νέα σας αποστολή με τον SSM. Νομίζω ότι είναι συναρπαστική εξέλιξη αυτή για την Κεντρική Τράπεζα που αναλαμβάνει την εποπτεία. Θα έχετε περισσότερες εξουσίες, όπως είπατε και πριν. Επανέρχομαι στην εισαγωγική σας ομιλία, όπου είπατε ότι θα θέλατε να δείτε συγκεκριμένες βραχυπρόθεσμες μεταρρυθμίσεις που να αναλυθούν από πολλές χώρες έτσι ώστε να βελτιωθεί η οικονομία. Και αν δεν έκανα λάθος, είπατε ότι θα θέλατε περισσότερο μακροπρόθεσμο όραμα. Ερώτηση λοιπόν, μπορείτε να μου πείτε μερικά συγκεκριμένα παραδείγματα των βραχυπρόθεσμων δεσμεύσεων που επιθυμείτε να δείτε και ποια θα θέλατε να είναι η εμπλοκή των συστημάτων οικονομικής διακυβέρνησης στην Ευρώπη. Το άλλο είναι η... το quantitative easing, η ποσοτική χαλάρωση. Είπατε ποιοι πρέπει να είναι όροι στην αρχή για την open market facility. Προφανώς είναι σωστό και τα κάνατε ως τώρα πολύ καλά τα πράγματα. Πώς βλέπετε την εμπλοκή του μηχανισμού κατεπίγουσας χρηματοδότησης, χορήγηση ρευστότητας δηλαδή, για το μέλλον του τραπεζικού συστήματος. Δράγκη, για την πρώτη σας ερώτηση. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν βραχυπρόθεσμες υποχρώσεις και μακροπρόθεσμες υποχρώσεις που θα πρέπει να, να ληφθούν. Οι βραχυπρόθεσμες αναφέρονται στις διαθωτικές αλλαγές που έχουμε συζητήσει κατά επανάληψη στο παρελθόν. Ολοκλήρωση της νομοθεσίας της ενιαίας αγοράς, αύξηση της ανταγωνιστικότητας, αλλαγές στην αγορά εργασίας, αλλά αυτές είναι πολύ ευρείες κατηγορίες. Κάθε χώρα μέλος έχει και το δικό της θεματολόγιο αλλαγών. Αυτό που λέω είναι απλό. Έχουμε σκεφτεί ξανά και ξανά, έχουμε προβληματιστεί, έχουμε αναλύσει τις μεταρρυθμίσεις αυτές. Ωστόσο λίγα πράγματα είναι γνωστά έως τώρα. Και αυτά τα είπαμε, αλλά πρέπει τώρα πια να αναλάβουμε δράση και να πάρουμε τι σχετικές αποφάσεις, που βεβαίω είναι δύσκολε αποφάσεις, γιατί καμιά φορά αλλάζουν σε βάθος την οργάνωση τη κοινωνία, όπω αυτή ισχύει εδώ και πολλά χρόνια. Είναι όμω σαφέ ότι οι αποφάσει αυτέ πρέπει να ληφθούν. Για το δεύτερο θέμα είναι οι μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις δηλαδή. Εάν επιστρέψετε και εξετάσετε την εμπειρία των τελευταίων 30-40 ετών. Οδηγήστε στο συμπέρασμα ότι η διαδικασία ολοκλήρωσης έχει περάσει μέσα από το χρόνο πάντα σε μια βάση, την ε, κοινή κυριαρχία. Βαθμιδών μοιραζόμαστε όλο και περισσότερο κυριαρχία σε διάφορους τομείς. Για παράδειγμα, στην νομισματική πολιτική. Πριν από την δημιουργία του ευρώ, οι περισσότερες χώρες της ζώνης ευρώ είχαν χάσει τελείως την νομισματική τους κυριαρχία για διαφόρους λόγους. Ε, η δημιουργία του ευρώ και η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας οδήγησε όλες αυτές στην κοινή διαχείριση αυτής της νομισματικής πολιτικής μέσα στα πλαίσια των οργάνων αυτών. Το ίδιο για την νομισματική ένωση. Σιγά σιγά έχασαν την κυριαρχία που πήγε στις αγορές. Ακόμα περισσότερο στην ε, Budgetary Union που από το να μην έχουμε καθόλου κοινού κανόνες έχουμε τώρα πραγματικά ένα κλάδο της ε, δημοσιονομικής πτυχής με κοινού κανόνες και ούτω καθεξής. Είναι σαφές ότι αυτή είναι η εμπειρία μας και πάνω σε αυτή την εμπειρία θα πρέπει να βασίσουμε τα επόμενα βήματα. Αυτό το οποίο εννοούσα όταν έλεγα μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις με δύο τρόπους, αφενός επέκταση του χώρου των κοινών κανόνων, όπου μπορούν να περιληφθούν και κάποιες κοινέ διακυβερνήσεις κοινών δομών και δεύτερο και πιο περίπλοκο βέβαια είναι να περάσουμε από τους κοινούς κανόνες σε κοινούς θεσμούς. Και εδώ σταματώ, διότι δεν είναι ούτε καθήκον μου, ούτε άλλωστε ε, ε, ε υπάγει τις αρμοδιότητες μου να υπαγορεύσω ποια θα πρέπει να είναι τα επόμενα βήματα. Ευχαριστούμε. Αλφισάντ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε Ντράγκη, πρώτα απ' όλα να εκφράσω το θαυμασμό μου για τον τρόπο με το οποίο φέρατε σε μια ισορροπία της αντιφάσεις της πολιτικής και της αποφάσεις που χρειάστηκε να πάρετε. Τώρα έχετε πολιτικές, μάλλον δεν έχετε πολιτικές ευθύνες ούτε εθνικές ούτε ευρωπαϊκές. Οι επιπτώσεις όμως είναι σημαντικές και έχετε κάνει δηλώσεις με τεράστια πολιτική σημασία όπως κάνατε και τώρα. Οι πολιτικοί που παίρνουν αποφάσεις φαίνεται ότι περιμένουν τις δικές σας δηλώσεις για να ε, καταλήξουν στον προσανατολισμό της δικιάς τους πολιτικής ευρωπαϊκή πολιτική βασίζεται λοιπόν σε δηλώσεις που μερικές φορές ξεπερνούν τις αρμοδιότητές σας προκειμένου να διακανιστούν τα θέματα της Ευρώπης. Έχετε πει ότι επιγόντως πρέπει να ενισχυθούν οι νομισματικοί θεσμοί της Ευρωζώνης και αναβαθύνουμε περισσότερο στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Αυτό σημαίνει περισσότερη ομοσπονδιοποίηση των ευρωπαϊκών θεσμών είναι ένα παράδοξο. Η Ευρώπη είναι, οι Ευρωπαίοι είναι υπέρ του ευρώ, όμως δεν θέλουν να μια ομόσπονδη Ευρώπη. Συγχρόνως οι οικονομικές αποκλήσεις στις διάφορες περιοχές και χώρες αυξάνονται και δεν μειώνονται. Ευάθυνση λοιπόν της ονέκατο από αυτές τις συνθήκες μάλλον θα επιτείνει τις αποκλήσεις. Από στρατηγικής πλευράς. Αυτά τα παράδοξα και αντιφάσεις μπορούν να παραμείνουν για πολύ καιρό ακόμα. Μέχρι τώρα οι πολιτικές επιλογές ήταν ε, κάποια βελτίωση επιφανειακή. Τώρα όμω, μήπω θα έπρεπε να εξετάσουν περισσότερο σε βάθο τι επιλογέ για το μέλλον τη Ευρωζώνης, δεδομένου ότι η οικονομικά δεν έχει τις επιδόσεις που έχουν άλλες οικονομικές περιφέρειες. Ποια είναι η αποψή σας γι' αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα για τα καλά σας λόγια όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τον Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου. Όλα αυτά οφείλονται βέβαια στους ιδρυτές ε, πατέρες περισσότερο και όχι στα σημερινά μέλη. Επιτρέψτε μου να προσθέσω ότι είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν εκφραζόμαστε στα πλαίσια της εντολής μας. Υπάρχουν διάφορες πτυχές της πολιτικής μας ή της πολιτικής άλλων που επηρεάζουν είτε την οικονομική σταθερότητα είτε ή μάλλον κατά πρώτον τη σταθερότητα τιμών. Έτσι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρέπει, οφείλει να μιλάει. Και επιτρέψτε με εδώ να αναφερθώ σε ένα ζήτημα μόνο για να απαντήσω στις σημαντικές σας παρατηρήσεις είπαμε ότι η εμβάθυνση στην ε, ΟΝΕ θα τίνει να ενισχύσει τις αποκλίσεις μεταξύ χωρών μελών. Εμείς συμφωνούμε για το ότι η Ευρωζώνη πρέπει να αναπτυχθεί περισσότερο. Οι σημερινές επιδόσεις είναι ελάχιστες και η ανεργία είναι ιδιαίτερα υψηλή, απαράδεκτα υψηλή. Ιδιαίτερα η ανεργία των νέων. κάτι το οποίο κοινωνικά είναι απαράδεκτο. Συνεπώς, συμφωνούμε ότι η Ευρωζώνη πρέπει να αναπτυχθεί περισσότερο. Αλλά πιστεύετε πραγματικά ότι φταίει το ευρώ και δεν υπάρχει αυτή η ανάπτυξη. Και εδώ είναι που δυσκολεύομαι να συμφωνήσω με την επιχειρηματολογία σας. Αν δείτε το τελευταίο τρίμηνο, τα στοιχεία του ΕΠ βλέπουμε ότι 14 14 χώρες είχαν θετική ανάπτυξη. Για κάποιες από αυτές μεταξύ 2 και 4% σε τίσια βάση. Βλέπουμε δύο χώρες σε ύφεση και βλέπουμε και δύο χώρες, αν δεν απατώμε, που να είναι σε σταθερή κατάσταση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Brian Hayes τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρε Ντράκη, την τελευταία φορά που ήρθατε στην Επιτροπή μας, σας ρώτησα σχετικά με τις Ιρλανδικές έρευνες όσον αφορά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η Ιρλανδία διασώθηκε και τι ακριβώς έγινε με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που παρενέβη. Σας ευχαριστώ για τη δημοσίευση των επιστολών που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι θετικό ο Ιρλανδικός λαός να μπορεί να ενημερωθεί και να βάζει τα πράγματα μέσα στο σωστό πλαίσιο. Βέβαια, καταλαβαίνω ότι όλα αυτά δεν έγιναν μόνο από εσά, έγιναν από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δέχομαι επίση ότι ένα πρόγραμμα οικονομική ενίσχυση το 2010 ε, δεν ήταν τίποτα άλλο από μια πραγματικότητα, γιατί δύο χρόνια οδήγησαν στην κρίση αυτή και η κατάσταση δεν μπορούσε να επιληθεί αλλιώ. Εγώ δεν θέλω να σα ρωτήσω τόσο πολύ για το παρελθόν, όσο για το μέλλον. Και όπως ρώτησαν και οι συνάδελφοι, θέλω και εγώ να μου μιλήσετε για την ανάμειξη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην Ιρλανδική έρευνα που λαμβάνει χώρα από το Ιρλανδικό Κοινοβούλιο. Η έρευνα αυτή δεν είναι κυνήγημα γησών. Είναι σημαντικό όμω οι Ιρλανδοί να γνωρίζουν την αλήθεια. Είναι επίση σημαντικό και για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, γιατί όπω είπατε πολύ σωστά πατώντα άλλου συναδέρφου, λογοδοτεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα και πρέπει να το κάνει όταν 25% της αρρωγής πήγε σε μία χώρα εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή, δεδομένη της καταστροφικής κατάστασης που βρισκόταν η χώρα και δεν μπορούσε να εγγυθεί το τραπεζικό σύστημα. Ρωτάω λοιπόν, μπορείτε να επιβεβαιώσετε εδώ στην Επιτροπή μας ότι συμφωνείτε με την ε, έρευνα που θα ελέγξει την ανάμειξη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και θεωρήσετε κάποιον υψηλό αξιωματούχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για να αποτελέσει τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στην Ιρλανδία και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και η τεκμηρίωση που έχει στη διάθεσή της Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για όλα αυτά τα θέματα από το 2008, 2009, 2010 θα διατεθεί για την έρευνα εφόσον η έρευνα χρειαστεί την τεκμηρίωση αυτή. Και τέλος, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, είπατε και εσείς ότι λογοδοτεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συμφωνώ. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όμως λογοδοτεί σε όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρόσθετα εγώ. Και δεδομένου ότι υπάρχει μια Ιρλανδική έρευνα χωρίς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, θα ήταν σαν να μην έχουμε ολόκληρο το οικοδόμημα και να κάνουμε μισές δουλειές. Τράγκη, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λογοδοτεί σε εσά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Άρα, επίσημα δεν θα συμμετάσχουμε σε μία επίσημη έρευνα Εθνικού Κοινοβουλίου. Δεν έχουμε συζητήσει ακόμα τι είδους μορφή θα πάρει τελικά η συμμετοχή η δικιά μας. Θα προβληματιστούμε, θα το συζητήσουμε. Επίσης, πριν από δέκα μέρες η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην ιστοσελίδα της δημοσίευσε διάφορα έγγραφα σχετικά με την Ιρλανδία. Και όλα αυτά περιλαμβάνουν όχι μόνο την ανταλλαγή επιστολών ανάμεσα στον πρόεδρο Τρισέ και τον κύριο Λένιχαμ, αλλά και διάφορες νομικές νομοδοτήσεις οι ομιλίες και λοιπά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Συνεπώς, επί του παρόντος, προχωρήσαμε στην δημοσίευση αυτή. Συζητάμε και θα δούμε. Να επανέλθω παρακαλώ για αυτό το θέμα. Όταν λέτε ότι επίσημα δεν θα συμμετέχετε στην έρευνα για το θέμα του συνδετικού Κρίκου που θα συνεργαστεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με την Ιρλανδία και για την τεκμηρίωση που μπορεί να χρειαστεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αυτά θα τα διαθέσετε. Πρόεδρος Δράκη, λέτε τι μορφή θα έχει επίσημη συμμετοχή μας. Ε, απάντησα σε αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει να το ξαναπώ. Δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα τίποτα σχετικό. Ούτε έχουμε ορίσει κάποιον αξιωματούχο, ούτε ξέρουμε τι τεκμηρίωση ενδεχομένως θα διαθέταμε. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Ναι, ευχαριστώ για αυτά που είπατε για το ότι λογοδοτείτε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που εκπροσωπεί τους Ευρωπαίους πολίτες. Περβάνς Μπερές τώρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρόεδρε Ντράγκη, τώρα που έχουμε την Τραπεζική Ένωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έχει αρχίσει η συζήτηση για τη δομή των τραπεζών. Θα ήθελα λοιπόν τη δικιά σας εκτίμηση για την ε, σημασία που μπορεί να έχει αυτή η δομή, τι μορφή θα έχει αυτή η δομή και τι είναι αυτό που ενδιαφέρει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου. Εσείς ο ίδιος είπατε ότι η ευρωπαϊκή οικονομία δίχως άλλο χρηματοδοτήθηκε υπερβολικά από το τραπεζικό σύστημα. Όμως η διασφάλιση του τραπεζικού συστήματος κόστισε στις οικονομίες των χωρών μελών πάρα πολλά και στο ευρωπαϊκό σύστημα στο σύνολό του. Έγιναν πάρα πολλά για να σωθούν οι τράπεζες. Και αν δεν σώθηκαν οι τράπεζες για να χρηματοδοτήσουν την οικονομία, τότε το τίμημα δεν είναι υπερβολικά ακριβό. Απλώς και μόνο, σε εισαγωγικά το απλώς, να αποφύγουμε συστημικό κίνδυνο. Και επιτρέψτε μου επίσης και μια ακόμα ερώτηση. Η κυρία Νογή δήλωσε πρόσφατα ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα μπορούσε να αγοράσει ε, κρατικά δάνεια αν ε, είναι αναγκαίο. Μπορείτε να σχολιάσετε παρακαλώ την δήλωση αυτή της Χριστίνου Αγία. Όσον αφορά το πρώτο σημείο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν έχει ακόμα υιοθετήσει γνωμοδότηση για το σημείο το σημαντικό το οποίο θέσατε όσον αφορά την ιδεώδη δομή των τραπεζών στην Ευρωζώνη. Η γνωμοδότηση αυτή πάντως θα υιοθετηθεί σύντομα και σίγουρα θα ενημερωθείτε μόλις την έχουμε. Ο λόγος για τον οποίο δεν είναι προφανές να το αποφασίσει κανείς είναι λίγο πολύ και απάντησε στη δεύτερη ερώτησή σας. Φυσικά και θέλουμε να έχουμε μια κατάσταση όπου μειώνονται οι συστημικοί κίνδυνοι και δεν επεκτείνονται εξαιτίας της δομής των τραπεζών μας. Συγχρόνως πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για το τι δραστηριότητες αυξάνουν το συστημικό κίνδυνο και άρα θα πρέπει να διαχωριστούν από το υπόλοιπο τραπεζικό σύστημα και ποιε όχι. Και αυτό το λέω για να καταδείξω τη δυσκολία του εγχειρήματο και γιατί δεν έχουμε ακόμα γνωμοδοτήσει. Κάτι το οποίο, όπως είπα, πολύ σύντομα θα γίνει γιατί οι κύριες συζητήσει έχουν ήδη ολοκληρωθεί για τη γνωμοδότηση αυτή. Και έρχομαι στην τελευταία σας ερώτηση. Η απάντηση είναι ναι είναι στα πλαίσια της εντολής μας. Και όπως είπα και πριν, το Συμβουλίο θέλει να ξεκαθαρίσει ότι υπάρχει δέσμευση να δράσει, δηλαδή να υιοθετήσει και άλλα μη συμβατικά μέτρα εφόσον ο κίνδυνος επιδεινώνεται, αλλά συγχρόνως στέλνει μηνύματα που δείχνει ότι είναι έτοιμη να δράσει, ζητώντας από το προσωπικό και τις σχετικές επιτροπές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να μελετήσουν και να προετοιμαστούν και να προετοιμάσουν και τεκμηρίωση. Παρακαλώ. Μια στιγμή, όταν λέτε ότι πρέπει να δούμε ποια είναι η δραστηριότητα των τραπεζών ε, από την οποία ελοχεύει ο μεγαλύτερο κίνδυνο, υποθέτω ότι δανείζουν σε επιχειρήσει για τη δικιά του ανάπτυξη οι τράπεζε και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε συστημικό κίνδυνο. Και ακριβώ γι' αυτό φτιάξαμε και τους κανόνε που φτιάξαμε. Όμω συχνά το θέμα της προσφυγής στην Κεφαλαϊκή Ένωση σε άλλο τρόπο χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων εμφανίζεται σαν εναλλακτική λύση. Αν λοιπόν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν μπορεί να δανείσει στην πραγματική οικονομία για να ενισχύσει την χρηματοδότηση, τότε τι νόημα έχει. Σωστά τα λέτε, λέει ο κύριος Ντράγκη. Συμφωνώ. Αλλά επιτρέψτε μου. Το μάθημα που πήραμε είναι ότι οι τράπεζες μπορεί να βρεθούν σε μια κατάσταση που να μην μπορούν πια να λειτουργούν. Δεν θέλουμε να το επαναλάβουμε αυτό. Δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε κάτι τέτοιο. Και το στόχο αυτό τον πετύχαμε με δύο τρόπους. Πρώτον, οι τράπεζες πρέπει να γίνουν πιο ανθεκτικές, πιο ισχυρές, με καλύτερη κεφαλαιοποίηση με καλύτερη δομή. Και δεύτερον, ακόμα και τότε δεν επαφιόμαστε απολύτως, αλλά θέλουμε να έχουμε και ένα άλλο κανάλι χρηματοδότησης της οικονομίας μας. Αυτή είναι η μελλοντική μας στρατηγική, γιατί την εμπειρία δυστυχώς την έχουμε και ήταν πολύ επώδυνη, όπως είπατε κι εσείς. Πρόεδρος, ωραία, τελευταίος ομιλητής, Μαρκοσέλο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσουμε κύριε Ντραγή. Διότι διαλέξατε την Νάπολη για να προβείτε στις σχετικές σας δηλώσεις. Είναι η ιδιαίτερη πατρίδα μου. Οπότε βεβαίω και με χρονοποιεί πάρα πολύ. Θα τώρα για μας όσον αφορά το τεστ αντοχής, τα στρες τεστ. Έχουμε την περίπτωση Μόντε Πάσχη της ε, Σιένα. Πρόκειται για μια τράπεζα της ε, Τοσκάνης η οποία έχει αυξήσει κατά 1,5 δις το κεφαλαιό της. Όμως, όσον αφορά τις μετοχές της, υπάρχει μεγάλη ανησυχία. Τι λέτε εσείς. Τι είναι με αυτή την αύξηση κεφαλαίου. Έχω τώρα μια άλλη ερώτηση να σας υποβάλω. Έχουμε εννέα τράπεζες οι οποίες πέρασαν επιτυχώς το τεστ αντοχής. Έχουν όμως προβλήματα με τον ηγετικό τους. Εάν συνεχιστεί η οικονομική κρίση, ιδίως από την ε, αύξηση της ε, πίεσης ε, στο στοιχείο των ιδιωτών τραπεζών λόγω της ε, συντήρησης της Βασιλεία υπαριθμών 3 υπάρχει πρόβλημα. Εσεί για αυτά τα τραπεζικά πιστοτικά ιδρύματα τι λύση θα προτείνατε. Μήπως θα πρέπει να προβούν σε πώληση κάποιων στοιχείων του ενεργητικού. Έχουμε επίση έξι διεθνείς σημαντικές τράπεζες στις οποίες επιβλήθηκαν πρόστιμα και φτάσαμε στα 4 δις. Γι' αυτό όσον αφορά κάποιες ισοτιμίες, όσον αφορά επίσης ε, κάποιες εντολές πελατών και άλλα θέματα ε, στα οποία είχαν σωστή συμπεριφορά. Η ΕΚΤ τι μπορεί να κάνει τόσο ώστε να ε, καταπολεμήσει αυτού του την χειραγώγηση των ισοτιμιών σε διεθνές επίπεδο. Και μιλάμε τώρα για το τι γίνεται εκτός Ευρωζώνης Δράγη. Ναι, όσον αφορά την πρώτη πρόταση ε, την αναλύουμε, την αξιολογούμε, τώρα που μιλάμε. Και όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, τότε θα δημοσιοποιήσουμε τα αποτελέσματα. Δεν είμαι βέβαιος πάντως για το κατά πόσο υπάρχει καθορισμένη μια ημερομηνία μέχρι την οποία θα πρέπει να έχουμε τοποθετηθεί. Πάντως ε, αυτό το οποίο είναι σαφές όσον αφορά τον χρόνο της ε, υλοποίησης έχουμε έξι μήνες αν έχει επισημανθεί το πρόβλημα ε, του, του, του ενεργητικού αν αυτό έχει γίνει από το, την, μελέτη αξιολόγησης και εννέα μήνες αν πρόκειται για το τεστ αντοχής το, είδε. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει στην περίπτωση ε, που έχουμε τον ενίο μηχανισμό μηχανισμό ε, που θα πρέπει να διαπιστώσει αν υπάρχει αξιοπιστία. Θα πρέπει τέλο πάντων για να μην γίνει τίποτα να πληρεί και τι τρει προποθέσει. Τώρα, όσον αφορά την ΕΚΤ, εμεί ε, και στο μέτωπο το θεσμικό και στο μέτωπο της ε, ιδιωτικής αγοράς προσπαθούμε να προωθήσουμε το να υπάρχουν κάποια κριτήρια και για τις ισοτιμίες, κάποιοι κανόνες ε, και αυτό βάσει πραγματικών συναλλαγών και όχι επί τη βάση κάποιων μοντέλων ή κάποιων εξατομικευμένων προβλέψεων και Εργαζόμαστε έτσι σε στενή συνεργασία με τις ε, κεντρικές τράπεζες παγκοσμίω και με την FSB. Δεν κατάλαβα πάντως το, το δεύτερο ερώτημά σας. Μπορείτε να το επαναλάβετε βεβαίω, λέει ο βουλευτής. να ναι, γνωρίζουμε ότι οι τράπεζες που περάσαν ε, αυτήν, αυτό το τεστ 19 δηλαδή, Κάποιοι από αυτές 19 περίπου έχουν, είναι προβληματικές με όσον αφορά το ενεργητικό τους και εάν η κρίση επιδεινωθεί ακριβώς λόγω της θέσεως ισχύω της ε, συμφωνίας της Βασιλείας Παριθμού 3 θα στριμωχτούν πολλοί αυτές οι τράπεζες. Επομένως, πώς θα μπορούσαν ε, αυτές οι τράπεζες να ξεπεράσουν αυτό το πρόβλημα πρέπει κάποια χαρτοφυλάκια να απολυθούν δραγή. Ναι. Είπαμε, θα πρέπει να γινει εξαιρούς εξαιρούση πρώτα-πρώτα των στοιχείων του εννοητικού, asset quality review και κατόπιν το αντοχή, αντοχής, οπότε και έτσι έχουμε ε, την τιμωρία, ιδίω εκεί που έχουμε ύφεση πολύ καιρό, οπότε το stress test τους ε, πλήσει ακόμη περισσότερο. Οπότε ε, έχουν περάσει αυτές οι τράπεζες κάποια αυστηρά τεστ όσον αφορά το, το πόσο... Συγγνώμη, γιατί ανακατεύω τις γλώσσες. Ε, αλλά τι να κάνουμε, τα τελικά είναι η μητρική μου γλώσσα, γι' αυτό τα ανακατεύουμε τα αγγλικά. Και επομένως η ουσία των όσων θέλω να σας πω είναι ότι έχει γίνει κάποιο είδους ε, τεστ δοκιμασία αντοχής, σκληρή για αυτές τις τράπεζες και είδαμε ότι ε, συμμορφώνονται και τώρα τι θα γίνει ε, αποκλείουμε οποιοδήποτε εκτροπή στο μέλλον δεν μπορούμε να αποκλείσουμε και θα πρέπει να γίνει συνεργασία του ενιαίου πολιτικού μηχανισμού με τους εθνικούς εποπτικούς φορείς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πρόεδρε Δράγη, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους. Τώρα η συζήτηση για τον Μηζονικό Διάλογο ολοκληρώθηκε το 2014. 2015 θα γίνει ο επόμενο διάλογο. Θα σα ε, γνωστοποιήσουμε το πότε θα γίνει, ποια ημερομηνία. Και πάμε τώρα ευθύ αμέσω. Πώ? Όχι, θα κάνουμε ένα δίλεπτο διάλειμμα. Και θα επανέλθουμε στο σημείο 5 τη μεσή διατάξεω. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ας αρχίσουμε πάλι με το επόμενο θέμα τώρα της ημερησίας διατάξεώς μας, που είναι η δημόσια κρόαση με παρουσία του Μάριο Ντράγκη, αλλά ως Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ε, Αξιολόγηση του Κινδύνου. Πρόεδρε, μέλη της Οικονομικής και Επιτροπής, κυρίες και κύριοι, με μεγάλη μου χαρά εμφανίζομαι ενώπιόν σα εδώ σε αυτή την επιτροπή που συνοδεύει σώμα τώρα πρόσφατα ή στην ιδιότητά μου, υπό την ιδιότητά μου μάλλον ως πρόεδρος του ESRB και για εσάς που είστε καινούργοι εδώ ελπίζω ότι πρόκειται να σας ενημερώσω αυτό το όσα θα πω γιατί το ECRB, αυτό το Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου παίζει σημαντικό ε, ρόλο όσον αφορά το να έχουμε ένα υγιέστερο ε, χρηματοοικονομικό, χρηματοπιστωτικό σύστημα που χρειάζεται για να έχουμε μια ανάκαμψη στην οικονομία της Ευρώπης γιατί οι ευρωπαϊκές αρχές έχουν πασχίσει πάρα πολύ ούτως ώστε να αναβιώσουν την εμπιστοσύνη στο ευρωπαϊκό σύστημα και αυτές ε, οι, οι προσπάθειες κατατείνουν στο έχουμε αυτό το τεστ αντοχής με το συντονισμό της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, σημαντικό τραπεζών υπό την ε, αιγίδα της Ευρωπαϊκή Εθνικής Τραπέζης και το Συμβούλιο Κινδύνου έχει συμβάλει ε, σημαντικά εδώ και πρόκειται και στο μέλλον να κάνει το ίδιο διότι επίσης ε, προδιαγράψαμε ποιο είναι το, το κακό μακρονομικό σενάριο για το τεστ αντοχής και έτσι θα δούμε ποιε είναι οι οι συνέπειες όσον αφορά την αντίστοιχη των τραπεζών στις εξελίξεις μακροοικονομικές. Επίσης το Συμβούλιο ε, εξετάζει αυτή την υπόθεση της αντιδιδολογική συμπεριφοράς και του κινδύνου την αντιδιδολογική συμπεριφορά ε, στο τραπεζικό τομείο και θα πρέπει οι τράπεζες επομένω να, υποστούν χρηματικές ποινές και άλλες κυρώσεις λόγω του ότι δεν ε, ετήρησαν τους κανόνες διοντολογίας Οπότε αυτού, ο χαρακτήρας, η φύση αυτού του κινδύνου είναι κατά το λέμε tail event και αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα όσον αφορά την αποδοτικότητα και τη φερεγγύη τραπεζών. Και έχουμε έτσι ένα τέτοιο κίνδυνο, το οποίο προέρχεται από πολλού ε, παράγοντε. Πολλέ φορέ αυτά τα θέματα ιδιωτική συμπεριφορά αναδύονται από τι αγορέ, αλλά και σε συστημικά σημαντικέ τράπεζε. Το δε κόστο είναι ολοένα και περισσότερο σε μια συγκυρία κρίση και γι' αυτό και οι επιπτώσει είναι τέτοιε που ευνοούν τη, τη κλικά φαινόμενα για τέλος αυτή η αντιδιωτική συμπεριφορά είναι κακή για την εμπιστοσύνη στις ε, χρηματοπιστωτικές αγορές και στα ιδρύματα για να λειτουργήσει όλο το σύστημα. Και γι' αυτό και θέλουμε σύμφωνα μαζί και με την αρχή των τραπεζών να έχουμε μια ελαχίστη μεθοδολογία ώστε οι τράπεζες να την εφαρμόζουν όταν θέλουν να υπολογίσουν το, πόσο κοστίζει σε, σε καταστάσεις πίεσης αυτού είδους η μη ιδιωτική συμπεριφορά και αυτό επίσης θα οδηγήσει σε μια ε, υγιή αξιολόγηση για όλες τις τράπεζες και θα έχουμε επίσης ε, και, κάποιο, και, και κάποια σχέδια διάσωσης, plan B για όλα τα κράτη και αυτό επίσης θα πρέπει να ε, αφορά και να καλυφθεί αυτού του είδους ο κίνδυνος και από τα μελλοντικά τεστ αντοχής. Να σου πω τώρα με την μακροπροληπτική πολιτική, γιατί άλλωστε αυτό είναι και μια ερώτηση που υπευλήθη προηγουμένως. Από τότε που είχαμε τους νέους κανόνες αστικής ε, διαχείρισης. Είχαμε την οδηγία για τις ε, ε, την οδηγία αλλά και τον κανονισμό για τις κεβολοχικές απαιτήσει και από τότε έχουμε τα, τα νέα μέσα μακροπολιτικής πολιτικής όπως επίσης το αντικυκλικό απόθεμα ασφαλείας τον Ιούνιο του 2014 το Συμβούλιο Κινδύνου ε, εξέδωσε μία σύσταση για το τι θα κάνουμε με, με, με αυτού του είδους το απόθεμα ασφαλείας, σε ποιο ύψος θα πρέπει να κυμαίνεται, είχαμε αποφάσεις σε σχέση με τις ε, ενδυνάμει ζημίες και σε σχέση με το πόσο θα μπορούσε να αυξηθεί ο συστημικός κίνδυνος και γι' αυτό είπαμε να έχουμε κάποιο είδους ε, περιθώριο τέτοιο ε, η πραγματική οικονομία μέσω του, του οικονομικού κύκλου και επίσης είπαμε ότι θα πρέπει να έχουμε τις, ε, τις εκτροπές αυτού του είδους της αναλογίας μεταξύ πίστοσης και ΕΠ που αυτό θα αφορά την αφετηρία για τις αποφάσεις μας ιδίως όσον αφορά τη φάση της ώρες των κινδύνων και επίσης έχουμε επισημάνει κάποιες περιπτώσεις όπου είχαμε και κάποιες άλλες μεταβλητές όπως κάποιες άλλες μεταβλητές των πιέσεων στις αγορές που χρηματοδοτούν τι τράπεζες και κάποιου δείκτες γενικού συστημικού κινδύνου ιδίως τις ε, κάποιες πρώτες χώρες που σε αυτό το πλαίσιο είδανε ότι αυτό το, το απόθεμα ασφαλείας είχε πάει στο 1% στη Σουηδία και 0% στην Τσεχική Δημοκρατία, Σλοβακία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Το Συμβούλιο Κινδύνου επίσης ε, αναθεώρησε μια σύσταση που είχαμε πει να υπάρχουν εθνικές αρχές μακροπροληπτικές και με αυτή την σύσταση βοηθήσαμε τις ε, εθνικές, ε, την εθνική αρμοδιότητα πάνω σε αυτό και επίσης γενικότερα την αποτελεσματικότητα του μακροπολιπτικού ε, μέσου. Γενικότερα θεωρήσαμε ότι αυτό είναι θετικό και ενθαρρύνουμε τα εκεί που Εκεί έχει καθυστερήσει αυτή η δικασία, ε, δηλαδή η Ιταλία, Λουξεμβούργο, Πολωνία, Ρωμανία και Ισπανία, να επιταχύνουν και να μπορέσουν να θεσπίσουν τη σχετική εθνική νομοθεσία του συντομότερο δυνατών. Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, διάφορα θεσμικά πρότυπα έχουν χρησιμοποιήσει, περισσότερε περιπτώσει έχουμε τι μακροπολιτικέ αρμοδιότητε, τι οποίε έχει η Κεντρική Τράπεζα ακριβώ όπω το Συμβούλιο στην Κινδύνου έχει συστήσει και σε πολλέ περιπτώσει η Εποπτική Αρχή και σε λίγε περιπτώσεις επιτροπές που, που προεδρεύει αυτόν η κυβέρνηση <clears throat> έμεσα ή άμεσα. Και τελευταία κάποια κρατημέλη έχουν χρησιμοποιήσει αυτό το πλαίσιο το μακροπροληπτικό. Η δε, το, το ΔΕ Συμβούλιο Κινδύνου έχει εξετάσει περίπου 30 τέτοια εθνικά μέτρα ε, συστημικού κινδύνου με μακροπροληπτικά. Ε, γενικώ αυτά τα μέτρα είναι δύο ειδών. Πρώτα-πρώτα όσον αφορά υπερβολική αύξηση των πιστώσεων, όσον αφορά τη μόχλευση και σχετικά με τον συστημικό κίνδυνο για κάποιο είδου ομίλου ε, τραπεζών που είναι πολύ μεγάλη και περίπλοκη. Ε, αυτού του είδου το απόθεμα ασφαλεία ανήκει στην πρώτη κατηγορία και εφόσον αυτού του είδου το περιθώριο, το απόθεμα αφορά κάποιου είδου εξελίξει για την πίστοση, έχει λιγότερο προσυδειάζει σε συγκεκριμένους κλάδους ε, όπως ε, τον τομέα της, ε, των, των ακινήτων, real estate και την κτήματα αγορά Επομένω, έχουμε πάρα πολλά κρατημέλη που έχουν υλοποιήσει τέτοια μέτρα, τα οποία ακριβώ στοχεύουν σε τέτοια, στην αγορά ή στην κτήματα αγορά κινήτων, Βέλγιο, Σουηδία και επίση κάποια άλλα κρατημέλη, Ουγγαρία, Ιρλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο, έχουν πιο αυστηρά κριτήρια για τον δανεισμό, loan to value, loan to income και επίσης ε, την εξυπηρέτηση, του, το ρυθμό εξυπηρέτηση ε, του, του, του, δανεισμού. Η δεύτερη κατηγορία τέτοιων μέτρων εστιάζεται στο πώ θα λυθεί το περίφημο πρόβλημα too big to fail, πολύ μεγάλο για να πτωχεύσει πρόβλημα και αυτό αφορά κάποιο είδου ε, ιδιαίτερε υψημένε κεφαλικέ απαιτήσει για τράπεζε που μπορεί να αποσταθροπήσουν το χρηματοοικονομικό σύστημα όταν υπάρχει κάποιο είδου στόχευση. Και έχουμε κάποια κρατημέλη, Τσεχία, Δανία, Κροατία και κάτω χώρε που έχουν ακολουθήσει αυτή την συνταγή. Κύριε Πρόεδρε και αξιότιμοι βουλευτέ, εν κατακλείδη, για να ρίξουμε μια ματιά στο μέλλον τώρα που έχει ολοκληρωθεί το τεστ αντοχή για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλω να δούμε τι γίνεται όσον αφορά του κινδύνου εκτό ε, τραπεζικού κλάδου. Γιατί οι αγορέ και όλε οι αρχέ, ε, όλο και περισσότερο προσέχουν το πόσο μετάβολες είναι οι χρηματαγορές και, και, και, ε, και οι πιστοτικές αγορές και αυτό γιατί πολλές φορές δεν υπάρχει αρκετή ρευστότητα γιατί οι υπηρεσίες ρευστότητος ε, στηρίζονται από αυτούς που διαμορφώνουν τις αγορές και γι' αυτό έχουμε κάποιο κατάλογο λίστα των ε, αξιογράφων ομολόγων μετοχών που υφίστανται συναλλαγή. Πάρα πολλοί παράγοντες έχουν βγει σε μια συρρήγνωση αυτών των ε, συναλλασσομένων. Η τεχνολογία πάντως μας επιτρέπει να έχουμε rollover και να το κάνουμε πολύ πιο γρήγορα και γι' αυτό έχουμε περισσότερο ανταγωνισμό και αυτό μας έχει οδηγήσει σε ε, holding ε, lower inventory σε, σε, σε λιγότερο επαρκείς τέτοιους καταλόγους και τέτοιες λίστες και αυτό γίνεται τώρα όποτε έχουμε πάρα πολλούς τόπους που γίνονται οι συναλλαγές και βέβαια ο κάθε τόπος συναλλαγής έχει δικά του χαρακτηριστικά. Οπότε γι' αυτό οι υπηρεσίες ε, ρευστότητος ε, έχουν ε, αυξηθεί λόγω του ότι είναι όλο ένα και πιο σημαντικοί οι διαχειριστές των στοιχείων του ενεργητικού. Και παθητικά και ενεργητικά έχουμε τα exchange trade funds, τα ETFs και αυτό γιατί Πρέπει να υπάρχει παρακολούθηση των κινήσεων στην αγορά, αγορώντας ή πολλώντας στοιχεία ενεργητικού και αυτό γίνεται γιατί γίνεται ε, επίσης συχνά ε, η κίνηση των συναλλαγών, οι πωλήσει και αγορές. Γι' αυτό και έχουμε λιγότερη προσφορά και περισσότερη ζήτηση και οπότε έχουμε σε κάποιες αγορές λιγότερη ρευστότητα και γι' αυτό έχουμε κάποιο είδους ε, ταραχές στην αγορά, διαταράξεις, αναταράξεις λόγω της ρευστότητας. Οπότε θα, όλα αυτά πρόκειται να τα ερευνήσει το Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου και ε, πρέπει να σας πω ότι την επόμενη συνάντησή μας θα σας ενημερώσω. Τέλος, θα πρέπει να σας πω ότι αρχάς επομένου έτους πρόκειται να δημοσιοποιήσουν η έκθεση όσον αφορά ε, το τι γίνεται με την ε, έκθεση προς το, σε σχέση με, την, με τις κανονιστικές αρχές. Και γι' αυτό πρόκειται για το, το μοναδικό τέτοιο, ε, τέτοια επίσημη έκθεση που έχουμε. Και αυτό πρόκειται να μας δώσει μια εποπτεία του τοπίου όσον αφορά τους κινδύνους ε, και το πόσο ε, έχουμε έκθεση σε κίνδυνο των τραπεζών αλλά και των ασφαλιστικών εταιριών και αυτό θα, θα περιλαμβάνει στοιχεία από το τελευταίο τεστ αντοχής οπότε θα, θα έχουμε σε αυτή την έκθεση και πώς μπορούμε με πολιτι, κάποιες πολιτικές μέσω πρόθεσμα να αντιδράσουμε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Thank you very much. Πρόεδρος Γκουαλτιέρη, ευχαριστώ. Είναι ενδιαφέρουσα τα θέματα. Δυστυχώς δεν έχουμε πολύ χρόνο. Θα παρακαλέσω λοιπόν τους συναδέλφους και τις συναδέλφους βέβαια να περιοριστούν σε τέσσερα λεπτά το πολύ και δυνατόν και λιγότερο. Και πρώτος είναι ο κ. Κύρτσος. Thank you, Δύο ερωτήσει, κύριε Πρόεδρε. Υπάρχει κίνδυνος να γίνει εξαντλητική υποπτία του τραπεζικού τομέα χωρίς να εποπτευθεί επαρκώς το shadow banking, έτσι αυξάνοντας τους συστημικούς κινδύνους. Και δεύτερο, τι γίνεται με την πολιτική των Αμερικανικών αρχών που επιβάλλουν τεράστια πρόστιμα σε ύψους δισεκατομμυρίων σε μεγάλες Αμερικανικές και Ευρωπαϊκές τράπεζες. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να εφαρμόσουμε αυστηρότερο καθεστώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να αποφευθούν ανεπίτρεπτες τραπεζικές συναλλαγές ή να διαμαρτυρηθούμε απέναντι στους Αμερικανούς που παρεμποδίζουν το έργο των Ευρωπαϊκών Τραπεζών. Για την πρώτη ερώτηση. Όλες οι πληροφορίες που ε, συλλέξαμε δείχνουν ότι μεταφέρονται από, από banks σε non-banks. Συγκρίνοντας τη σχέση των τραπεζών με αυτά προ ετών, δείχνει τη σημασία των νέων παικτών. Οι δραστηριότητες non-bank, non-insurance. Επίσης σημαντική είναι η αύξηση των μη παραδοσιακών ασφαλιστικών δραστηριοτήτων. Πριν από λίγα χρόνια σημαντικό ρόλο έπαιζαν τα hedge fund που φάνηκαν ωστόσο να είναι και πιο ανθεκτικά στην τροτότητα. Ήδη αρχίσαμε να ασχολούμαστε με money market funds. Έχουμε μια σύσταση από το 2012. Επίσης αγορές OTC. Είναι σαφές ότι χρειάζεται να ολοκληρώσουμε το νομικό θεματολόγιο και να υποβάλουμε όλους τους τομείς της αγοράς στην ίδια εποπτεία. Συμπληρώνω διότι ε, όχι μόνο το Συμβούλιο, η ανησυχία που εκφράσατε είναι παγκόσμια και γίνεται ε, κάποιο έργο και στο επίπεδο του FSB. Για το δεύτερο θέμα σας, το δεύτερο ερώτημά σας, είναι σαφές και τα τελευταία γεγονότα, τα πιο πρόσφατα γεγονότα δείξανε ότι είναι αρκετά σαφές ότι πρώτα-πρώτα η αντιδοντολογική ε, συμπεριφορά τραπεζών είναι πραγματικό πρόβλημα. Δεν είναι επινόηση των διαφόρων ε, δικαστικών δικαιοδοσιών. Δεύτερο, ότι η ισχύουσα νομοθεσία που αναφέρεται σε συνεργαζόμενες τράπεζες είναι υπερβολικά περίπλοκη. Τρίτο, αυτές οι κυρώσεις που εφαρμόζονται από διαφορετικές δικαιοδοσίες, ε, από διαφορετικά δικαστές, διαφορετικές δικαιοδοσίες με διαφορετικό τρόπο, έτσι ώστε τράπεζες με παγκόσμια λειτουργία εκτίθεται σε διαφορετικές εφαρμογές και διαφορετικά πρόστιμα και αυτό εξαρτάται από το που κρίνεται η περίπτωσή τους δικαστικά. Υπάρχει λοιπόν ένα τεράστιο πεδίο συντονισμού παγκοσμίω και στις αρχές όταν καταγράφηκαν, συγγράφηκαν αυτές οι κυρώσεις, τα βασικά δηλαδή νομικά κείμενα, θα πρέπει να περιλαμβάνουν και προβλέψεις για το πώς θα εναρμονιστεί βαριά λέξη αυτή βέβαια για τις δικαστικές δικαιοδοσίες αλλά που θα υπάρχουν κάποιες συμβατότητες έτσι ώστε να προσεγγίσουν. Ιάκωβος φων Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι ιδιαιτέρως που εξετάζεται την, τις συστημικές αδυναμίες ορισμένων εκθέσεων. Δύο ερωτήσεις. Πρώτα, σχετικά με τις δοκιμασίες αντοχής. Υπό την ιδιότητά σας ως Προέδρου του Συμβουλίου Αξιολόγησης Συστημικού Κινδύνου, θα ότι ο συστημικός κίνδυνος δεν ληφθεί υπόψη αρκετά ή και καθόλου στις δοκιμασίες αντοχής. Υπό την ιδιότητα σας λοιπόν που προανέφερα, πώς βλέπετε την απόφαση σχετικά με μελλοντικέ δοκιμασίε αντοχής, να μην περιλάβουν δηλαδή συστημικά στοιχεία. Δεύτερη ερώτηση αναφέρεται σε μια συναρπαστική έκθεση που συνετάχθη από την Επιστημονική Επιτροπή του Συμβουλίου σας, αξιολογήσεως συστημικού κινδύνου, με τον τίτλο Is Europe Overbanked? Μήπως έχει προβολικά πολλές τράπεζες η Ευρώπη. Από τον περασμένο Ιούνιο και νομίζω ότι η Επιτροπή Οικονομικών δεν είχε ακόμα την ευκαιρία να το συζητήσει μαζί σας. Πριν να υποβάλω την ερώτησή μου, ωστόσο, ήθελα να διαβάσω ένα σύντομο τμήμα της εκθέσεως. Δεν είμαστε οι πρώτοι γιατροί που έρχεται να δει το European ε, Banking System αυτή την ε, περίοδο. Ο ασθενής μας έχει αρχίσει κουράζεται από τα φάρμακα που του δίνουμε, λέει εδώ, και από τη θεραπεία. Ορισμένες θεραπείες πρέπει να χορηγηθούν ωστόσο σε μεγαλύτερη δόση, άλλες δεν έχουν δοκιμαστεί καθόλου. Για να αποκατασταθεί η υγεία του Ευρωπαϊκού Δραπητικού Συστήματος πρέπει να ληφθούν μέτρα ώστε να ξεφουσκώσει συχνά πολλοί θεωρούν ότι είναι πολύ φουσκωμένο το σύστημα, διότι μεγάλε ευρωπαϊκέ τράπεζε έχουν αυξηθεί πολύ ταχύτερα από το καθαρίστο εθνικό προϊόν και πολύ ταχύτερα από αμερικανικέ τράπεζε. Και οι θεραπείες που ζητούνται εδώ είναι μεταξύ αυτών και νομοθεσία antitrust για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Τα θέτω αυτά υπόψη σα διότι εγώ επεξεργάζομαι τμήματα τώρα της ε, νομοθεσίας για τη μεταρρύθμιση των τραπεζών που θα βασιστεί και σε εκθέσεις δικές σας. Από τη δική σας όμως πλευρά του Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου συμφωνείτε με την έκθεση αυτή. Σας ευχαριστώ πλήωνα θέματα. Πρώτον για την ε, έκθεση σε κρατικά ομόλογα, σε κρατικά δάνεια. Λήφθηκε υπόψη αυτό. Υπάρχει μια ενδιαφέρουσα έκθεση από την Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή που θα δημοσιευθεί του χρόνου και η οποία προτείνει ορισμένα μέτρα πολιτικής τα οποία μπορούν να αντιμετωπίσουν την ε, υπερβολική έκθεση των χαρτοφυλακίων των τραπεζών σε κρατικά δάνεια. Με διάφορα κριτήρια, κριτήρια διαφοροποίησης, του πυλώνος 3 για ε, δημοσιοποίηση ορισμένων στοιχείων και την οδηγία Solvency 3. Αυτά είναι σημαντικά, διότι κατά κάποιο τρόπο έχουμε δει πόσο σημαντική είναι η διασύνδεση μεταξύ κρατικών δανείων και τραπεζών. Έχουμε λοιπόν ε, να λάβουμε αυτό υπόψη, αλλά ταυτόχρονα οι αλλαγές αυτές, όπως η Αλλαγέ των εθνικών επιλογών που ανέφερα προηγούμενα στην προηγούμενη παρουσίασή μου, δηλαδή πώς να αντιμετωπίσουμε το λεγόμενο goodwill, τον αέρα που λέμε, των τραπεζών. Πώς να αντιμετωπίσουμε την ανάγκη ενός ε, ε, ισότιμου ανταγωνισμού για ορισμένα στοιχεία του ενεργητικού. Αυτά ενδεχομένως να πρέπει να συμφωνηθούν σε παγκόσμιο επίπεδο, έτσι ώστε να μην δημιουργηθεί ένα μη ανταγωνιστικό περιβάλλον, ένα στρεβλό ανταγωνιστικό περιβάλλον δηλαδή, στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Χρειάζεται λοιπόν πολλή δουλειά ακόμα και στην Επιτροπή Βασιλείας και στην EFSB. Αυτό που πρέπει ίσως να πω είναι ότι το συνολικό κλίμα δεν είναι διόλου εχθρικό απέναντι στις αλλαγές αυτές. Δεν το λέω αυτό με την έννοια ότι βρήκαμε κάποια εχθρική υποδοχή απέναντι στις προτινόμενες αυτές αλλαγές. Όχι. Αλλά αυτό που λέω ιδίω είναι ότι χρειάζεται να υπάρξει παγκόσμια συμφωνία για το ε, ισότιμο ε, πεδίο ανταγωνισμού για τις αλλαγές αυτές. Το δεύτερο που είπα, τη δεύτερη έκθεση που αναφέρατε και συμφωνώ μαζί σας ότι είναι εξαιρετική και θα συζητηθεί βεβαίως ήδη διεξήχθη στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διάσκεψη σεμινάριο για την έκθεση αυτή και θα μελετήσουμε και θα προβληματιστούμε από αυτού, διότι περιλαμβάνει πολλές αλήθειες η έκθεση αυτή και πρέπει βέβαια να πούμε και πιο συγκεκριμένα πράγματα. Εγώ πιστεύω ότι όντω περιλαμβάνει πολλές αλήθειες η έκθεση. Σας ευχαριστώ, ο πρόεδρος Γκουαλτιέρη και η Σουίνμπορν, η επόμενη ομιλητριά μας. Ευχαριστώ. Επειδή είμαι μέλος διαπραγματευτικής ομάδας εδώ, θεωρώ ότι η εντολή G20, G20 για το εμπόριο των παραγόγων είναι σημαντικό για την παρακολούθηση του συστημικού κινδύνου που προέρχεται από τα παγκόσμια αυτά προϊόντα. Καθώς προχωρούμε τώρα ωστόσο στη χορήγηση εντολής για τα παράγωγα, ρίχνουμε ιδιαίτερο βάρος στον κίνδυνο αυτών των CCP, που ε, γίνονται ωστόσο συστημικά πάρα πολύ ε, σημαντικά και προκαλούν συστημικό κίνδυνο. πολλές από τις τράπεζες οι οποίες ε, υπόκεινται σε αυτό και επειδή και εμείς στην BRD έχουμε παρόμοια ε, εργαλεία, μήπως θα πρέπει να εξετάσουμε μέτρα για την απορρόφηση των κραδασμών, απορρόφηση δηλαδή των ε, απολειών για να σταθεροποιηθούν τράπεζες στο μέλλον. Η απάντηση είναι ναι συμφωνώ μαζί σας. Το TILAC είναι κέριο μέτρο για να αντιμετωπίσει κανείς ε, περιπτώσεις τραπεζών που είναι υπερβολικά μεγάλες για να τους επιτραπεί να πτωχεύσουν και βεβαίως ο κίνδυνος τότε αναλαμβάνεται, πρέπει να αναλαμβάνεται από τους μετόχους και όχι από τους φορολογούμενους. Το σύνολο της ε, ικανότητας απορρόφηση κρατασμών θα πρέπει να είναι μεταξύ 16 και 20% των συνολικών ενεργητικών ως ελάχιστη απέτηση του πυλώνα 1 και βεβαίως μετά από μελέτη επιπτώσεων και ε, εποπτείας της αγοράς. Όπως γνωρίζετε η FSB έχει αρχίσει εγχείρημα στάθμισης και συνεργαζόμαστε και εμείς. Μια ερώτηση ακόμη. Θα τα εφαρμόσετε αυτά και στα CCP. Αυτό, κοιτάξτε, πρέπει να το επαληθεύσω πρώτα. Θα έλεγα προχείρως ότι υπάρχουν λόγοι για να γίνει αυτό. Αλλά η FSP έχει κάνει τώρα πρόταση για να εφαρμοστεί ο TILAC στα CCP. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω, δεν μπορώ να σας δώσω οριστική απάντηση από αυτού. Ευχαριστώ. Λεν Ευχαριστώ, Πρόεδρε Ντράγκη. Και εγώ έχω δύο ερωτήσει. Παρακαλώ. Τους τελευταίους μήνες η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μείωσε τα επιτόκια σε βαθμό ρεκόρ. Επεκτείνει τον ισολογισμό από ό,τι φαίνεται με OTM για τίτλους και για το CP3 και για άλλα προγράμματα. Ακούσαμε κάποιες κερδοσκοπικές προσπάθειες για ομόλογα, ακόμα και για κρατικά ομόλογα. Στην Ιταλία και την Ισπανία είδαμε αύξηση στην ε, έκδοση Τζάνκερ ομολόγων που δεν έγινε για χρόνια. Εσείς συμφωνείτε με τις ανησυχίες που εκφράστηκαν από διάφορες κεντρικές τράπεζες τους τελευταίους μήνες μεταξύ άλλων και της Bundesbank και του Ηνωμένου Αλυσίου. Ηνωμένου Ασλού που λέει ότι η πολιτική αυτή οδηγεί σε αποθάνηση των επενδυτών, κάτι το οποίο θα οδηγούσε νέες φούσκες και νέα, νέο ηθικό κίνδυνο. Θεωρείτε και εσείς ότι όλα αυτά αποτελούν ε, απειλή για τους στόχους μακροπροληπτικής πολιτικής όσον αφορά τώρα τις κεφαλαϊκές απαιτήσει. Τον Ιούλιο του 2014 Υπήρξε έκθεση για τι διάφορες κοινοποίησει. Πολλές από αυτές είχαν να κάνουν με χώρε οι οποίες επέβαιναν ασφάλειες ε, συστημικού κινδύνου με απόθεμα το οποίο χρησιμοποιόταν ε, σαν υποκατάστατο των ε, τακτικών αποθεματικών ασφάλειας με αποτέλεσμα συστημικό κίνδυνο. Θα μπορούσαν όμως από το 2016 και μετά να επιβάλλονταν. Στη δικιά σας έκθεση του Ιουλίου εκφράσατε κάποιες ανησυχίες για το ότι πολλές χώρες χρησιμοποιούν το ESRB και το εφαρμόζουν σε διάφορες τράπεζες ως υποκατάστατο τακτικών ε, ECR απαιτήσεων. Ανησυχείτε για τις εξελίξεις αυτές και τι μέτρα θα εφαρμόσετε έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να χρησιμοποιείται Συγγνώμη, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου να χρησιμοποιείται όπως πρέπει από τις χώρες. Δράκη, Μια χαλαρή νομισματική πολιτική θα μπορούσε να οδηγήσει σε υψηλότερους κινδύνους για χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει ακουστεί από διάφορες νομολογίες που επέκτηναν τον ισολογισμό τους πολύ περισσότερο αναλογικά με εμάς. Αλλά εδώ πρέπει να κάνουμε τρεις διαφοροποίησεις. Πρώτον, υπάρχουν κατηγορίες ε, χρηματοπιστωτικών ε, φορέων που είναι περισσότερο εκτεθειμένοι. Ιδίω εκείνοι οι οποίοι διασφαλίζουν σταθερά κέρδη. Αυτό έχει να κάνει με τις ασφαλείς ζωής, με τις δακτυλωτικά ταμεία και διάφορες άλλες αγορές ΣΥΝΑΠ. Δεύτερον, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες υπάρχουν κινήσεις σε πραγματικές τιμές που οφείλονται και σε διαρθρωτικούς λόγους, νέα ε, νομικοί περιορισμοί, ε, φορολογία, αλλά και σε προβλήματα ρευστότητας υπέρ των επενδύσεων. Έπειτα, η αστάθεια δεν μπορεί να αποκλειστεί. Τα χαμηλά επιτόκια ενθαρρύνουν κάτι τέτοιο που σημαίνει ότι οι τιμές των περιουσιακών στοιχείων έχουν να κάνουν περισσότερο με το συνέστημα παρά με την πραγματική αξία. Προς το παρόν δεν βλέπουμε πάντως πώς ε, μπορεί να υπάρχει συστηματική υπεραξιολόγηση. Υπάρχουν κάποιες εκτιμήσεις των αγορών ακινήτων από εμά, από το διεθνές Συνατικό Ταμείο, δεν δείχνουν ένα ιδιαίτερα έντονο πρόβλημα αυτή την εποχή. Και βέβαια, αν δούμε τι έγινε τους τελευταίους μήνες, βλέπουμε ότι υπήρξαν και διορθώσεις στις υπεραξιολογήσεις αυτές. Συνεπώς παραμένουμε προσεκτικοί. Πάντως, παρόλα αυτά, πιστεύουμε ότι η δικιά μας νομισματική πολιτική είναι καταλληλότερη όσον αφορά την εντολή μας, που είναι πληθωρισμός κάτω αλλά κοντά στο 2%. Και η κίνδυνη οικονομικής αστάθειας είναι πράγματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν με μακροπροληπτικά εργαλεία. Αυτή είναι η πρώτη, στην πρώτη γραμμή μας. Δεύτερον, είναι αλήθεια ότι χρησιμοποιήθηκε το απόθεμα ασφαλείας αντί για το εσωτερικό απόθεμα ασφάλειας για τις μεγάλες τράπεζες, αλλά είναι περισσότερο θέμα διαδικασιών και αναμφίβολα χρησιμοποιήθηκε ο πιο εύκολος δρόμος. Οικονομικά όμως συμφωνούμε με τα μέτρα και συνέβη σε πολλές χώρες, μία από αυτές είναι οι κάτω χώρες. Ευχαριστώ. Πρόεδρος να συγκεντρώσουμε κάπως τις ερωτήσεις γιατί έχει ένα αεροπλάνο όπου πρέπει να προλάβει ο κύριος Δράγκη. Οπότε παρακαλώ τους συναδέρφους να είσαστε σύντομοι. Επόμενη ερώτηση, Ματ Κάρτι. Τρει ερωτήσεις θα ακούσω μαζί. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και πάλι κύριε Δράγκη σας ευχαριστώ. Είμαι καινούριο στην Επιτροπή αυτή και προσπαθώ να καταλάβω πώς λειτουργεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου και τον ρόλο που παίζει. Ένα από τα πράγματα που με εξέπληξαν, όταν φτιάχτηκε η Μπέρντ για παράδειγμα είναι πόσο κεντρική είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και πώς εσείς είσαστε πρόεδρος και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του ΕΣΚΑ. Γι' αυτό και θέλω να ρωτήσω Υπάρχει, μπορεί να υπάρξει σύγκρουση συμφερόντων με την έννοια ότι θα μπορούσαν αποφάσει της Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να οδηγήσουν σε συστημικούς κινδύνους. Οπότε πώς θα τους αντιμετώπιζε τότε ο ΕΣΚ. Νωρίτερα αναφερθήκαμε στο Ιρλανδικό τραπεζικό σύστημα και την τραπεζική κρίση στην Ιρλανδία. Συμφωνώ ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έπαιξε ένα ρόλο στην δημιουργία αυτής της κρίσης. Με... Σίγουρα οι τράπεζες ε, προέβησαν σε υπερδανισμό, αλλά δανείστηκαν και αυτές από αλλού. Πράγματα τα οποία τα ήξερε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και μια συγκεκριμένη τώρα ερώτηση. Νωρίτερα είπατε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα στήριζε μια κεφαλαϊκή ένωση αγορών. Αυτό θα μπορούσε να αυξήσει τον συστημικό κίνδυνο και αν ναι, εσείς τι κινδύνους προβλέπετε και πώς πιστεύετε ότι ο κίνδυνος αυτός μπορεί να περιοριστεί. Ευχαριστώ. Θέλω να σας πω ότι δεν είναι καλό οι μικρές ομάδες τελικά να χάνουν το χρόνο τους συγκεντρώνοντας έτσι τις ερωτήσεις όπως προτείνετε. Έρχομαι όμως στην ερώτησή μου. Κύριε Ντράγκη, Σίγουρα θα έχετε διαβάσει τις εφημερίδες την ομιλία του κύριου Κάμερον, στην οποία έλεγε ότι υπάρχουν πιναλιές ε, στην γενική εικόνα της ε, ευρωπαϊκής οικονομίας. Θέλω λοιπόν να ξέρω κατά πόσο εσείς βλέπετε τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο. Βλέπετε και εσείς τα διακόκκινα φώτα. Ε, έχω μια πολιτική ερώτηση και κάποιες πιο τεχνικές. Πρώτον λοιπόν, Είπατε εσείς ο ίδιος νωρίτερα πόσο σημασία έχει η εμπιστοσύνη για να ενισχυθεί η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Πιστεύετε ότι οι ηγέτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση βοηθούν όταν αναφέρονται στην χρηματοπιστωτική κρίση. Έπειτα ο Καμερό αναφέρθηκε στο χαμηλό βαθμό οικονομικής ε, μεγέθυνσης, τα ευρωομόλογα κτλ. Γενικά τα επίπεδα είναι πάρα πολύ χαμηλά και η εμπιστοσύνη το ίδιο. Συμφωνείτε ότι μηνύματα αντιφατικά μεταξύ τους οδηγούν σε απώλειες και οι επενδυτές πιστεύετε ότι λειτουργούν έχοντας υπόψη τους ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα λειτουργήσει ως μηχανισμό στήριξης. Δράγκη, σας ευχαριστώ. Συγγνώμη, ο πρόεδρος Κύριε κύριε αρχίζω να σας λυπάμαι, ξέρετε. Είσαστε σαν έναν γιατρό που παρέχει ό,τι φάρμακο υπάρχει, αλλά όλο ένα και χειρότερα είναι ο ασθενής λέτε για το συστημικό κίνδυνο και μας λέτε το ρυθμιστικό πλαίσιο δεν μπορεί να ευνοεί ε, το, κυκλικό φαινόμενο, μα τι είναι, είναι τελικά κάτι που οδηγεί σε αστάθεια. Και άμα σταματήσει ο κύκλος τελείως, τότε ξεκινά κανείς μια μακρά περίοδο ε, οικονομικής ύφεσης, η χαμένη δεκαετία δηλαδή. Οπότε και αυτό γιατί δεν είχαμε κάποιο είδους προσοχή ή και μέτρα τέλος πάντων διασφάλιση του χρόνια. Και άρα τελικά ήμασταν χαλαροί όσον αφορά τον κίνδυνο, τον συστημικό τόσο καιρό. Οπότε μήπως θα έπρεπε να πείτε στι κυβερνήσει Ευρωζώνης ότι το κοινό νόμισμα ε, τώρα δεν μπορεί να λειτουργήσει. Τράγκη. Σας ευχαριστώ. Να αρχίσω την τελευταία ερώτηση. Εάν δεν έχετε αντίληση, δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι η κρίση δεν ξεκίνησε στην Ευρωζώνη. Η χρηματοοικονομική κρίση λόγω της χαλαρότητας των κανόνων ξεκίνησε αλλού, σε μια χώρα που την ξέρετε πολύ καλά ποια ήταν. Και τώρα πάμε να δούμε την άλλη σας ερώτηση. Έχουμε σύγκρουση συμφερόντων συμφερόντος μεταξύ των είναι κάποιος πρόεδρος του Συμβουλίου για την κρίση και τις τράπεζες. Ε, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι, καμία στιγμή δεν διαπίστωσα να υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων και αρμοδιοτήτων, δεν ξέρω τώρα, μέχρι το 2015 ε, δούμε τι θα γίνει, δεν ξέρω τι θα ρυθμιστεί, θα δούμε, ό,τι θέλετε. Και υπάρχει κάποια πρόταση να έχουμε κάποιον ε, διευθυντή για τον ε, για το Συμβούλιο Κινδύνου. Εάν συνεχίσει να λειτουργεί στα πλαίσια της Κεντρικής Τράπεζας, αυτό που θέλουμε με αυτό το νέο διαχειριστή, διευθυντή τέλο πάντων, είναι να συντονίζεται με την σημερινή γραμματεία και με την ΕΚΤ. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να συνεχίσει να έχει τον ίδιο πρόεδρο το Συμβουλίο Κινδύνου. Τέλος, εδώ, όπως είπα, όλα απόκεινται στους συνομοθέτες, εσάς και την Κομισιόν. Τώρα, μήπως η Ένωση Κεφαλαιογορών θα αυξήσει τον κίνδυνο. Άνοιξε μια ματιά στην εμπειρία που έχουμε. Τελικά το, η, η απουσία διάβλου χρηματοδότησης έχει αυξήσει την αβεβαιότητα για τον κίνδυνο. Γιατί μπορεί αν έχουμε έναν διάβλο να εκεί έχουμε κάποια εμπλοκή όπως, όπως με τώρα τις τράπεζες και για τις αγορές ίσως θα μπορούσαν να στηρίξουν το πρόβλημα των τραπεζών και με ε, έκδοση μετοχών ε, τελευταίων τα ίδια κεφάλαια οπότε δεν θα πρέπει να στηριζόμαστε μόνο σε ένα διάβλο ε, Τώρα, όσον αφορά το δεύτερο το οποίο είπατε, τι να πω, σε αυτά που λέει ο κόσμος. Ο κόσμος λέει ότι του έρχεται, ότι αισθάνεται. Αλλά για να δούμε εντάχει τον κατάλογο των κινδύνων από πλευράς ε, του Συμβουλίου. Πρώτα-πρώτα, η μακροοικονομική ευαλωτότητα ε, λόγω του, του συνδυασμού χαμηλής ανάπτυξης, ε, χαμηλών επιτοκίων, ε, υψηλό χρέος των νοικοκυριών, των εταιριών και του κράτους. Όταν έχουμε λοιπόν και αυτά τα, τα τρία χρέος, ε, επιτόκια, όταν όλα αυτά ισχύουν σε, σε πολλούς κλάδους, είναι κίνδυνος. Επίσης, δεύτερος κίνδυνος θα μπορεί να αφορά ε, τις, τις παγκόσμιες αγορές που όταν υπάρχει αυτός κίνδυνος τότε μπορεί να μην έχουμε τόσο πολύ ρευστότητα και αυτό είναι κίνδυνος και αυτό είναι ένα σενάριο δηλαδή μπορεί να αλλάξουν τα επιτόκια και το θέμα είναι πώς αυτό θα επιδράσει στην οικονομία και πώς θα αντιδράσουν οι εμπλεκόμενοι λόγω των μεταβολών στο επιτόκιο. Τρίτον, άλλο, άλλο θέμα μπορεί να είναι ε, στους ισολογισμούς που να είναι ευάλωτες εταιρείε. Ακριβώς ότι είπαμε και για την συμπεριφορά εκτός διοντολογίας. Τέταρτος κίνδυνος να γίνει ακόμα χειρότερη η κρίση του κρατικού χρέους και, ή και ελλείμματος. Αυτό έχει να κάνει και με αυτό που είπατε εσείς. Πώς θα αντιδράσουν οι αγορές στην σημερινή κρίση των κρατικών ομολόγων. θα επιδείξουν λογική αγορές. Η απάντηση είναι εξή. Άπαξ και οι κυβερνήσεις συνεχίσουν εξυγίανση των δημοσιονομικών, ιδίως αν συνεχίσουν τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, τότε οι τιμές αν ανταποκρίνονται στους κινδύνους και έχουν βιωσιμότητα. Εάν όμως ξαφνικά είχαμε αντιστροφή, ιδίως όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις, και αν συνεχίσουμε στην χαμηλή ανάπτυξη, τότε οι τιμές θα είναι άσχετες με την πραγματική κατάσταση. Ίσως έχουμε εδώ πέρα ε, κάποια, κάποια ευαισθησία όσον αφορά τα, το πώς μας κάνει βάλωτος το, το χαμηλό επιτόκιο και επίσης κάτι άλλο το οποίο είπατε, μπορεί να έχουμε τέτοιες διαρθωτικές ε, αδυναμίες όσον αφορά ε, την, ε, τη δομή της αγοράς, CCB, που όπως αναφέρατε. Δεν λέω ότι όλα αυτά θα συμβούν. Απλώ αν κάνει ρίξει μια ματιά του και αναζητήσει την επόμενη πηγή κινδύνου, να, ένα κατάλογο πιθανών πηγών κινδύνου. Όχι, με τίποτα δεν θέλω να πω ότι εμεί ε, θεωρούμε ότι αναδύονται αυτοί οι κίνδυνοι που ανέφερα. Και σα ευχαριστώ. Γκολτιέρη. Και τώρα οι τελευταίοι δύο αγορητές. Κύριε Πρόεδρε της ΕΚΤ, από τις 4 Συνδεκάτου είσαστε τώρα ο πραγματικός επικεφαλής των τραπεζών στην Ευρώπη με το SSM και είπαμε ότι είχαμε την τελευταία αξιολόγηση όσον αφορά την οδηγία των τραπεζών. Ήταν μια μεγάλη επιτυχία, όπως εσείς και κύριε Νόρ. Και επίσης όμως είστε και ο πρόεδρος της, ε, του, αυτού του, του Συμβουλίου και ακολουθώ τη μακροπροληπτική, το μακροπροληπτικό έλεγχο για τους θεμικούς κινδύνους. Με όλη αυτή τη σόρευση των αποστολών σας τώρα έχετε Ελέγχετε τα πάντα στην Ευρωζώνη. Το 2012 ε, εκδώσατε κάποιες ε, συστάσεις και έτσι στιγματίσατε το σχεδόν τραπεζικό σύστημα την τιτλοποίηση, δηλαδή που ξεκίνησε το 2007 με ε, την κρίση των subprimes. Εξηγήστε μας, γιατί κάνατε μια στροφή 180 μοίρων για τις σχεδόν τράπεζες και τι θα γίνει με την τιτλοποίηση που ήταν το κλειδί της νομιστικής σας πολιτικής επίσης για το Συμβούλιο ε, της Σταθερότητας το FSB προλίγο είπατε για, για έλεγχο 30 τραπεζών και ευρωπαϊκών ε, γαλλικών και στα πλαίσια του, του τεστ έγιναν γεφαλοποίηση αλλά δεν θα αντέξουν την επόμενη κρίση και όπως το 2013 στην Κύπρο είχατε, είχατε αυτό το μηχανισμό εξηγήνωση έγινε το μπίλιν αυτή η διάσωση με ίδια μέσα και είχαμε αυτό, αυτό ό,τι έγινε με τις καταθέσεις για να ενισχυθούν οι τράπεζες από τα ίδια κεφάλαια. Ο FSB επομένως τώρα τι, γίνεται όσον, τι θα κάνει όσον αφορά τη Συμφωνία της Βασιλείας 3 θα πρέπει το σταθμισμένο 20% των ερητικών να το πλήσουν αυτές οι τράπεζες για να σωθούν ή πώς αλλιώς μπορεί να γίνει αύξηση το κεφαλαίου πάρα πολύ έτσι ε, ευνοείται τις ιδιωτικές ε, τράπεζες αλλά αυτό δεν είναι κοινωνική πολιτική και επομένως ε, ταλαιπωρείται πάρα πολύ και δίδεται κινδύνο τους Ευρωπαίους και ιδίω να αφορά την απασχόληση. Τελευταίος είναι ο κύριος Χόκμαρκ. Ευχαριστώ, λέει ο κύριος Χόκμαρκ. Ακούγοντας τις συζητήσεις αυτές, καμιά φορά αποκτά κανείς το συνέστημα ότι το καλύτερο θα ήταν να μην έχουμε και καθόλου τράπεζες, γιατί τότε δεν θα είχαμε και κίνδυνο στο τραπεζικό τομέα. Όμως σε αυτή τη στιγμή έχουμε τράπεζες, είναι ενδιαφέρον να ακούσουμε από εσά πώς πρέπει να ερμηνευθούν οι εμπειρίες που αποκτήσαμε και από τη δοκιμασία αντοχή. Είπατε ότι θα είμαστε σε καλύτερη μοίρα τώρα και θα έχουμε περισσότερε, μικρότερε τράπεζε, περισσότερε και μικρότερε. και επειδή γίνεται αυτή η σύγκριση συχνά, λιγότερη χρηματοδότηση μέσω τραπεζών όπως γίνεται στις ΗΠΑ. Αντιλαμβάνεστε ότι κάπου το πάω. Αλλά παρόλα αυτά θα ήθελα να ακούσω τις απαντήσεις σας πρώτα. Ο πρόεδρος Δράγκη, για την πρώτη ερώτηση, εάν δούμε, αν εξετάσουμε τι συμβαίνει στον τραπεζικό τομέα, τι συνέβη δηλαδή στα τελευταία 7 χρόνια από την αρχή της κρίσης τέλη του 2007, θα δούμε ότι άλλαξαν πολλά πράγματα. Πανασχεδιάστηκε ολόκληρο το κανονιστικό πλαίσιο εφαρμόστηκε, άλλο μένει να εφαρμοστεί. Πάντως ο προσανατολισμός είναι τώρα ξεκάθαρος. Το τραπεζικό σύστημα σήμερα είναι πιο ανθεκτικό, σίγουρα, από ό,τι ήταν παλαιότερα. Και το τελευταίο, το τελευταίο παράδειγμα είναι και το TILAC που ανέφερα πριν. Επίσης οι πρακτικές του management και τα κίνητρα έχουν αλλάξει βαθιά στον τραπεζικό κλάδο. Το να πει κανείς ότι δεν έχει γίνει τίποτα βρίσκω ότι είναι υπερβολικό. Ταυτόχρονα συμφωνώ ότι δεν πρέπει να επαναπαθούμε και να μην κάνουμε τίποτε περισσότερο. Πρέπει να συνεχίσουμε να εποπτεύουμε και να είμαστε να επαγρυπνούμε για τις εξελίξεις διότι βέβαια ο τραπεζικός και ο ταμέας της οικονομίας δεν είναι στατικός κάθε άλλο. Τώρα στοχεύουμε και στο non-banking τομέα ή shadow banking οι δοκιμασίες αντοχής έδειξα, έδωσαν σημαντικές ενδείξεις σχετικά με την κατάσταση της υγείας του τραπεζικού τομέα στην, στον τομέα της ζώνης ευρώ. Και για πρώτη φορά προσέφεραν πιο εναρμονισμένους ορισμούς, για παράδειγμα για τα δάνεια που δεν αποδίδουν, non-performing loans. Και βέβαια πρέπει να βελτιώσουμε τις πρακτικές μας σε ό,τι αφορά πιο συμβατά ε, κεφαλοχικά μέτρα, αφενός αξιολόγηση του αέρα, goodwill, των ε, στοιχείων του ενεργητικού και των internal rating models των ε, τραπεζών, κυρίως των μεγάλων τραπεζών. Αυτό ως μερική απάντηση για τις γαλλικές τράπεζες. Οι γαλλικές τράπεζες εξάλλου δεν φάνηκε από τις δοκιμασίες ατοχής να είναι υπό, ε, να έχουν ε, χαμηλότερο κεφάλαιο από το απαραίτητο. Μιλούμε για την αρχή μιας μακράς πορείας προς την κατεύθυνση του να υπάρχει ένας επόπτης αλλά και μία εποπτική πρακτική σε ολόκληρη τη ζώνη ευρώ. Για το τελευταίο θέμα, μικρές τράπεζες ή μεγάλες τράπεζες είναι πολύ δύσκολο ερώτημα. Εφόσον οι τράπεζες είναι πάρα πολύ μικρές, είναι σαφές ότι οι συστημικές επιπτώσεις θα είναι μικρότερες, πιθανά, από του να πτωχεύσει μια πολύ μεγάλη τράπεζα. Ωστόσο, μέχρι ενός μεγέθους είναι δυνατόν να γίνουν οικονομίες κλίμακος και οι οικονομίες εύρους που θα επιτρέψουν μέχρι ένα σημείο καλύτερους οικονομικούς όρους υπέρ της πραγματικής οικονομίας και από την άποψη των τιμών, της, ε, των ποσοτήτων, των τεχνικών συμβουλών κλπ. Από μια στιγμή και μετά όμως, από κάποιο μέγεθος και μετά, η περιπλοκότητα παίρνει το πάνω χέρι και γίνεται πολύ πιο δύσκολο να ε, γίνει η διαχείριση του συστήματος, αλλά ταυτόχρονα και πιο επικίνδυνη. Το ερώτημα λοιπόν είναι μάλλον ποιον ρωτάτε. Αν ρωτήσετε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και που είναι κυρίως μικρές, προτιμούν τις μικρές τράπεζες που είναι πιο κοντά στον πελάτη, πιο κοντά και τοπικά επίσης, αλλά και υπάρχει και ένα συσχετισμός δυνάμεων ενώ στην περίπτωση μιας πολύ μεγάλης τράπεζας η μικρομεσαία επιχείρηση αισθάνεται σαν ένας νάνος μέσα σε ένα κόσμο γεγάντων. Από την άλλη μεριά οι μεγάλες τράπεζες προσφέρουν μια ποικιλία υπηρεσιών που συχνά μπορεί να είναι χρήσιμες για τις ΜΜΕ. Το άλλο που πρέπει να εξετάσουμε και η ερώτησή σας άπτεται αυτού που είπα προηγουμένως αν η ε, ζώνη ευρώ είναι overbanked είναι λίγο πολύ η ίδια ερώτηση. Το άλλο θέμα λοιπόν που πρέπει να συζητηθεί είναι το κόστος του να διαθέτουμε ένα τραπεζικό σύστημα που συναπαρτίζεται κυρίως από μικρές τράπεζες αν εξετάσουμε ορισμένες χώρες που έχουν πολλές εκατοντάδες μικρών τραπεζών και κάθε μια από τις τράπεζες αυτές έχει ένα διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από 5 μέχρι 19 μέλη και συχνά μάλιστα τα διοικητικά σε αυτά συμβούλια είναι πολύ πολιτικοποιημένα. Η μισθή των μελών του Συμβουλίου είναι κάθε άλλο παρά μικρή. Φτάνουν και τις 100 και πλέον χιλιάδες. Και αυτά πληρώνονται τελικά από τον πελάτη. Είναι λοιπόν πολύ περίπλοκο το ερώτημα. Και είναι και ένα από τα θέματα που απασχολεί το Συμβούλιο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, λέει ο Πρόεδρος Γκουαλτιέρη. Θα περιμένουμε με μεγάλη ανυπομονησία το έργο σας για τα liquidity shocks τους κραδασμούς της ρευστότητας και τα άλλα αποτελέσματα των προσπαθειών σας. Η ημερομηνία της επόμενης συνάντησης με εσάς ως πρόεδρο του Συμβουλίου θα κοινοποιηθεί, από, ε, θα κοινοποιηθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Thank you, colleagues. Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε να περάσουμε στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Στη δεύτερη ακρόαση, μάλλον ακούσαμε περισσότερα νέα από ότι στο πρώτο. Δεν ξέρω, δημοσιογράφοι μπορούν να τα χάσανε, εμείς όχι. Λοιπόν, περνάμε στο σημείο 6 της ημερήσιας διάταξης. Έχουμε τη έκθεση για την νέα πολιτική ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συγητής μας είναι ο κύριος Μέσερ Σμιτ. Θα του δώσω ευθύ αμέσω το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως γνωρίζετε, η αρχική μας έκθεση έχει να κάνει με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πολιτική ανταγωνισμού για το 2013. Είμαστε μέσα βέβαια σε μεγάλους περιορισμούς για να ετοιμάσει κανείς μια ολοκληρωμένη έκθεση. Προσπάθησα πάντως να συμπεριλάβω όσο μπορούσα περισσότερο τα σημαντικά στοιχεία για μας. Πριν λοιπόν αναφερθώ στα επιμέρους θέματα, να σας πω ότι είχαμε καρποφόρες συνομιλίες με τους σκιώδεις εισηγητές και προσβλέπω σε συνάντηση και με τους υπόλοιπους συναδέρφους εδώ μέσα στις επόμενες εβδομάδες για να μπορούμε να καταλήξουμε σε έναν συμβιβασμό και να έχουμε όσο γίνεται ευρύτερη πλειοψηφία που θα στηρίξει την έκθεση αυτή. Όχι μόνο πολιτικά μιλώντας, αλλά και ρεαλιστικά αν το δείτε και πρακτικά. Τα θέματα αυτά είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι σημαντικό λοιπόν για μας να μπορούμε ε, παρόλα αυτά να εκφράσουμε τη δικιά μας άποψη. Γι' αυτό λοιπόν έχει μεγάλη σημασία να καταλήξουμε σε συμβιβασμό. Όπως ήδη σας είπα, συναντηθήκαμε με το νέο επίτροπο που είναι αρμόδιος για το χαρτοφυλάκιο αυτό. Είναι από τη χώρα μου. Και έτσι ίσως είναι και πιο εύκολο η επικοινωνία μεταξύ μας. Πράγματι πήρα το σχέδιο έδειξε ότι θέλει να ακούσει και να συνεργαστούμε. Λοιπόν, κατόπιν τούτων, ας δούμε τα επιμέρους θέματα που έχουμε να εξετάσουμε και που βρίσκονται στο σχέδιό μου. Το πρώτο θέμα που είναι ζωτική σημασία νομίζω είναι η εσωτερική κατανομή πόρων μέσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όλοι γνωρίζουμε ότι ο τομέας του ανταγωνισμού είναι πολύ σημαντικός προκειμένου να λειτουργεί ικανοποιητικά η Ευρώπη. Ξέρουμε επίσης ότι οι διάφοροι φορείς από τον ιδιωτικό τομέα, αν όχι ε, άπειρους, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουν τεράστιους πόρους να δαπανίσουν. Θυμάμαι και από την προηγούμενη φορά ότι υπήρχαν διάφορες ε, που λέγανε ότι ήταν ε, προτιμότερο να πληρώνει κανείς πρόστιμα παρά να μην κάνει αυτό που έκανε, ότι δηλαδή τα κέρδη είναι μεγαλύτερα από τα πρόστιμα που έπρεπε να πληρώνουν. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ασκεί τους ελέγχους όπως πρέπει να τους ασκεί για τις κρατικές επιδοτήσεις κλπ. Στο σημείο 2 της ε, έκθεσης, το αναφέρω αυτό επειδή πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κατόπιν τούτου είναι εξίσου σημαντικό να επικεντρωθούμε και στα θέματα των κρατικών ενισχύσεων. Στην έκθεση της Επιτροπής καταλαμβάνει ένα μεγάλο κομμάτι αυτό το θέμα. Και το θέμα των επιστροφών. Εδώ έχουμε να κάνουμε με τις τράπεζες, μετά μάλιστα την οικονομική κρίση. Αλλά υπάρχουν και νέα θέματα, όπως το σημείο 6 και μετά, πράγματα που έχει θέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων μέσω των διορθωτικών ταμείων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα έχει ετοιμάσει ένα, μια νέα δέσμη κανονισμών για την χρήση των κονδυλίων αυτών. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να κάνουμε αξιολόγηση για το πώς εφαρμόζονται όλα αυτά στην πραγματικότητα. Γενικά πάντως μιλώντα. ο τρόπος με τον οποίο οι χώρες και άλλε δημόσιες αρχές χρησιμοποιούν τα χρήματα έχει τεράστια σημασία για την εσωτερική αγορά και πρέπει να είναι ένα από τα βασικά ζητήματα που θίγει μια έκθεση σαν και αυτή. Αντιτράστ τώρα. Και αυτό ξέρω ότι απασχολεί πάρα πολλά μέλη της Επιτροπής μας. Εδώ, κυρίως στο σημείο 9, αναφέρω την ανάγκη για πιο συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές, για προθεσμίες, δικαιώματα και διαφάνεια στην όλη διαδικασία που εμπίπτει στην αρμοδιότητα αυτή. Σίγουρα για πράγματα όπως η υπόθεση που έχουμε τώρα με την Google ή άλλα για τα οποία θα θέλαμε να υπάρχει διαφάνεια για να εφαρμόζονται σωστά κανόνες. Σημείο 12. Θα δείτε ότι εδώ αρχίζει η ανάπτυξη ανατομέα. Όσον αφορά την ενέργεια πρώτα απ' όλα. Εδώ υπάρχει μεγάλο εμπόδιο με το unbundling σε ορισμένες χώρες, σε ορισμένες αγορές που αποφάσισαν να μην εφαρμόζουν το τρίτο ενεργειακό πακέτο. Άρα παραμένει μεγάλος κατακαιρματισμός στην ενεργειακή αγορά, κάτι απαράδεκτο. Ο κατακαιρματισμός της ενεργειακής αγοράς είναι σαν να κλείνουμε τους αυτοκινητοδρόμους μας. Είναι απαράδεκτο αν θέλουμε να έχουμε ίδιους όρους και συνθήκες για όλους. Δεύτερον, ψηφιακή αγορά. Όλοι γνωρίζουμε ότι έχει τεράστιο δυναμικό. Ήταν πάντα πολιτικό ζήτημα και κατά τη διάρκεια των ευρωπαϊκών εκλογών αλλά και, αξίζει να το αναφέρουμε, κατά την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ήταν ένα από τα θέματα τα οποία υπογράμμισε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη σημασία ακριβώ που έχει. Και το εξηγώ και εγώ πιο πολύ στην ιδεολογική μου σκέψη. δεδομένου ότι δεν είχα αρκετό χώρο για το να αναπτύξω περισσότερο στο κύριο σώμα της έκθεσης. Επανέρχομαι στις αρχικές μου παρατηρήσεις όσον αφορά τις αρμοδιότητές μας ή τις δυνατότητες που έχουμε να επηρεάσουμε την πολιτική της Ευρωπαϊκής Πολιτικής. Πιστεύω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συγγνώμη. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να μας ακούσει, θέλει να συναντηθεί μαζί μας όπως και με τον προηγούμενο επίτροπο εδώ, αλλά ίσως και κάποια άλλη σύνθεση σε μια ομάδα εργασίας να μπορούμε να συναντιόμαστε μαζί τους. Είναι κάτι που πρέπει να προσπαθήσουμε. Νομίζω ότι υπάρχει η βούληση από πλευράς του Επιτρόπου. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα τώρα. Από τώρα Έχουμε 10 μέρες, τώρα που έχουμε όλες μεταφράσεις, 10 μέρες για να προτείνουμε τροπολογίες. 27 Νοεμβρίου είναι η προθεσμία. Θα οργανώσω συνάντηση με τους κοιόδης εισηγητές και μετά το Δεκέμβριο είτε στις Βρυξέλλες είτε στο Στρασβούργο. Θα σας πω πότε. Μετά θα ψηφίσουμε εδώ στις 27 Ιανουαρίου. Και άρα θα πάμε στην Ολομέλεια του Φεβρουαρίου για να ψηφίσουμε την έκθεση αυτή. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ τον εισηγητή. Η Σκιώδης, παρακαλώ τώρα. Τρία λεπτά ο καθένας. Παρακαλώ, Μπέρναρ Λάγκε, ο πρώτος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η πολιτική ανταγωνισμού πράγματι είναι από τι εκτελεστικέ αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει μεγάλη σημασία. Και δεν είναι και επινόηση των τελευταίων ετών. Περιλαμβάνεται ήδη στις ιδρυτικές συνθήκες τη Ρώμης. Όμως έχει λησμονηθεί. Επανέρχεται στην συνειδητοποίηση των διαφόρων κρατικών επιπέδων μόνον εφόσον πρόκειται για υποθέσεις ανεπίτρεπτης επιδότησης. Γι' αυτό το πρώτο που πρέπει να ζητήσουμε είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βελτιώσει την επικοινωνιακή στρατηγική των αποφάσεών της και των νομικών βάσεων. Εγώ θα υποβάλω και σχετικές τροπολογίες. Ώστε δηλαδή να γίνουν περισσότερα πράγματα υπέρ μιας ενεργού πολιτικής του ανταγωνισμού. Που άλλωστε έτσι περιλαμβάνεται και στις ιδρυτικές συνθήκες. Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή λειτουργεί ως οικονομία της αγοράς με ελεύθερο ανταγωνισμό. Στο σχέδιο εκθέσεως του κ. Σμιτ δεν περιλαμβάνει τίποτε σχετικό και θα κάνω εγώ τις σχετικές συμπληρώσεις. Δεύτερο, έχουμε έγγραφα από τα τελευταία χρόνια και το καλύτερο από αυτά τα έγγραφα είναι το σχέδιο του εκθέσεως του κ. Ραμών Τρεμόζα Ιμπαλσές που ψηφίστηκε ήδη στο προηγούμενο κοινοβούλιο και που καλύπτει όλα τα ανοιχτά ερωτήματα που συζητούμε τα τελευταία χρόνια. Ένα χρόνο μετά καλούμαστε να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβεί σε μια απογραφή των όσων επιτέχθηκαν και των όσων εκκρεμούν ακόμη. Και για αυτά θα κάνω εγώ σχετικές τροπολογίες. Όσον αφορά την δόμηση και τα ανατομής θέματα. Ο κύριος Μέσο Σμιτ έχει καταστρώσει ένα πρώτο σχέδιο που ωστόσο χρήζει προσθήκων βελτιώσεων και συμπληρώσεων. Έχω κάνει πολλές τροπολογίες εγώ, έχω συντάξει δηλαδή πολλές τροπολογίες, διότι η απόφαση αυτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την πολιτική ανταγωνισμού αποτελεί τη δική μας τοποθέτηση για ένα σημαντικό τομέα της ε, ευρωπαϊκής πολιτικής, όπου δεν έχουμε νομοθετική αρμοδιότητα ή πάντως πολύ περιορισμένη. Γι' αυτό είναι σημαντικό να μπουν τα πράγματα αυτά στην έκθεση και ιδίως μια προτροπή προς την νέα Επίτροπο να καταβάλει προσπάθειες εξυγχρονισμού όχι μόνο σε συνεργασία με τις χώρες μέλη διότι βεβαίως επειδή το δίκαιο προέρχεται όπως είπα από τις αρχικές ιδρυτικές συνθήκες στηρίζεται κυρίως σε αποφάσεις των κυβερνήσεων. Όμως πρέπει να μπει τώρα και στη διαδικασία συναποφάσεων. Πρέπει λοιπόν να είναι η τακτική, η συνήθις διαδικασία για τις κατευθυντήριες γραμμές και για όλες τις σχετικές αποφάσεις. Έτσι λοιπόν και για το θέμα αυτό πρέπει να περιληφθούν σχετικές τροπολογίες στην έκθεση. Έχω και ένα άλλο θέμα. Πρέπει να δούμε τις τρεις διαστάσεις της πολιτικής ανταγωνισμού, των άρθρων 101 έως 109. Μίλησε για τις κρατικές επιδοτήσεις ο κ. Μπεσεσμίτ και σωστό. Σημαντικό θέμα διότι από αυτές προκαλούνται στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. Οι τοπικές αυτοδιοίκησεις δεν δέχονται παρέμβαση της Ευρώπης. Υπάρχουν δε πολλά παραδείγματα. Αυτά πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε μέσα στα πλαίσια των οδηγιών. Υπάρχει εξάλλου η απαγόρευση των συγχωνεύσεων και υπάρχει και η έννοια της σχετικής αγοράς, καθώς επίσης και η απαγόρευση καρτέλ, καθώς και σχετικών συμφωνιών. Υπενθυμίζω εδώ και πάλι την έκθεση του παρελθόντος έτους, που διαλαμβάνει πολλά θέματα από αυτά που συζητώ τώρα. Και τέλος, η κατανομή των κονδυλίων που περιλαμβάνει στην έκθεσή του ο εισηγητής. Ήδη η σχετική αρχή έχει χίλιους προσοντούχους ε, συνεργάτες. Δεν μπορούμε να ζητήσουμε ως πρώτο μέτρο την αύξηση του οργανογραμματός τους. Εγώ και δεν πρόκειται να συμφωνήσω. Γκουαλτιέρη, ευχαριστώ. Θα πρέπει ωστόσο να ζητήσω από όλες και όλους να σεβαστούν το όριο των τριών λεπτών, διότι κάποια στιγμή θα αποχωρήσουν οι διερμηνείς. Τίμπορ Σάνι, Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να τηρήσω το τρίλεπτο, το όριο που είπατε. Λέει ο κύριος Σάνι. Πάντως, δεν είναι θέμα ευγένειας, αλλά ουσιαστικά πρέπει να, να συγχαρούμε συγγνώμη, τον κύριο Μέσος για την εισήγησή του και ελπίζουμε ότι αυτή η έκθεση ε, θα είναι και στο τέλος όπως τώρα και στην αρχή της άρτια και ωραία. και όχι μόνο για μας εδώ στο Κοινοβούλιο αλλά και έξω. Νομίζω ότι σήμερα είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά. Αν σκεφτούμε πώς έχει σήμερα ο ανταγωνισμός στην Ευρώπη. έχετε πολλές βελτιώσει η κατάσταση του ανάγωνισμού στην Ευρώπη. Και τονίζω τα εξή τρία που θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ βασικά στους σοσιαλδημοκράτες. Πρώτα πρώτα. Να έχει όσο γίνεται πιο σημαντικό ρόλο η αγορά, η ψηφιακή. Να τη λάβουμε υπόψη όσο γίνεται περισσότερο γιατί θα είναι η ατμομηχανή, θα είναι η κινητήρια δύναμη για να ε, πάμε στην καινοτομία και σε περισσότερη απασχόληση. Επίσης, οι σοσιαλδημοκράτες δεν θέλουμε να προωθηθούν κάποιες πρωτοβουλίες που δεν θα λαμβάνουν υπόψη της ΜΜΕ και τα συμφέροντά τους. Αντίθετα, πρέπει να δούμε πώς θα του δώσουμε μια όθηση προ τον μπρο. Κατά δεύτερο λόγο, επίσης, θα πρέπει να καλύψουμε και το πρόβλημα της διαφθοράς. Είτε γίνεται στο δημόσιο, είτε γίνεται από πλευρά επιχειρήσεων. Κατά τρίτο λόγο και ίσω είναι το πιο σημαντικό, ο ανταγωνισμό δεν αφορά μόνο το να ευημερούν οι επιχειρήσεις. Θα πρέπει να εξυπηρετεί και την ευμάρεια, το συμφέροντων των καταναλωτών. Αυτό θα πρέπει να λέμε υπόψη πάνω απ' όλα. Αυτά θα ήθελα να καλυφθούν κατά κάποιο τρόπο στην έκθεση. Χέρι Ρεμόν Τρεμόσα. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρώτα πρώτα να ευχαριστήσουμε τον εισηγητή για το έργο του. Νομίζω ότι με την έκθεση αυτή θα έχουμε ενδιαφέρουσα συζήτηση για πολλά ζητήματα και όταν μελετήσουμε και στροπολογίες θα εμβαθύνουμε. Βεβαίω και συμφωνώ ότι θα πρέπει να γίνει καλύτερη χρήση των ανθρωπίνων πόρων από πλευράς Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού. Τα είπα πέρσι που είχα μία έκθεση. Οπότε δεν μπορώ να συμφωνήσω ότι συνεχίζεται εκεί που το άφησα εγώ το θέμα επίση. Δεν λέω να έχουμε λένε οι περισσότερου υπαλλήλου, απλώ θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε καλύτερα του ανθρώπινου πόρου γιατί είδαμε ότι σε πολλέ περιπτώσει κάποιε ερευνητικέ πολυεθνικέ έχουν περισσότερο προσωπικό από τη γενική μα διεύθυνση. Αυτά λέει η πολιτική μα ομάδα. Επίση, θα υποβάλω κάποιες τροπολογίες όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις προς τις τράπεζες και θα πρέπει να ασχοληθεί περισσότερο με αυτό η Γενική Διεύθυνση. Σε κάποια κρατημέλη έχουμε συγκέντρωση στον τραπεζικό κλάδο. Στην Ισπανία, Φερρυπίν, κατά την κρίση πολλές τραπεζές έκλεισαν και οι τρεις μεγαλύτερες ε, ε, κατέχουν το 80% σχεδόν της αγοράς. Οπότε μειώνονται οι πιστώσει, ο δανεισμό προ τι ΜΜΕ και έχουμε όμω λοιπόν όλε αυτέ τι πληροφορίε και αυτό, γι' αυτό πρέπει να, η Γενική Διεύθυνση να αναλύσει τη, τη σχέση μεταξύ ε, της του των πιστώσεων προ τι ΜΜΕ και τη συγκέντρωση στον τραπεζικό κλάδο. Άρα, να δούμε πώ αυτή η έκθεση θα καλύψει την πραγματική οικονομία πολλού κλάδου αυτή, να δούμε αν υπάρχει αρκετό ανταγωνισμό προ τούτο και γι' αυτό και πέρυσι στην έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης αναφέρθηκε ο κλάδος των μεταφορών διότι σε κάποια κρατημέλη το σύστημα των λιμένων και των αερολιμένων είναι κεντροκατευθυνόμενο και ελέγχεται από την κεντρική κυβέρνηση της χώρας. Οπότε και γι' αυτό και δεν έχουμε εκεί συνδίκες να στην Ευρώπη αεροδρόμια και λιμένες. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ τους. Ανταγωνίζονται βέβαια με άλλα έργα υποδομή, αλλά νομίζω τέλος πάντων ότι πρέπει η Γενική Διεύθυνση να το τσεκάρει. Το ίδιο και για τον ενεργειακό τομέα, εκεί όπου ε, επισημαίνουμε διαφορετικές και αυξητικές τάσεις τιμών σε κράτη-μέλη, γιατί και αυτό βέβαια πλήσει την ανταγωνιστικότητα. Και σε αυτό θα κατεβάσω μια τροπολογία. Και ελπίζω ότι η Γενική Διεύθυνση θα τα αναλύσει. Το ίδιο και όσον αφορά την οδηγία για τις υπερήμενες οφειλές. Ξέρετε, αυτή η προθεσμία των 30 ημερών δεν τηρείται από όλες τις κυβερνήσεις. Όπως και πέρσι θα κινηθώ για τις τροπολογίες. Θα τα, θα, θα, δεν θα είναι πολιτικά ορθώς, δηλαδή θα τα ανεβάσω στο Google και θα καλέσω να απαντήσουν μετά οι συνάδελφοι. Πολύ σημαντική η υπόθεση Google. Μια ΜΜΕ και για άλλες επιχειρήσεις. Αυτά θα πω για το Google. Το είπαμε και πέρσι. Και θυμάμαι ότι 604 ψήφους υπέρ η έκθεση. Όλες οι μεγάλες ομάδες. Άρα ας το λάβουμε αυτό υπόψη και γι' αυτό ας πορευτούμε ένα λόγο και φέτος. Καλησπέρα. Δύο πράγματα έχουμε να πούμε. Το πρώτο ότι υπάρχει διαφορά, υπάρχουν διαφορές όσον αφορά την πολιτική ανταγωνισμού. Το είπαμε και κατά την εκπόνηση της έκθεσης για την Ευρωπαϊκή Συνεργασία. Το κύριο εμπόδιο της ανάκαμψης δεν είναι προσφορά, είναι ζήτηση. Χωρίς αυτήν, ό,τι ρυθμίσεις και αν υιοθετήσουμε δεν οδηγούν σε ανάπτυξη. Η πολιτική ανταγωνισμού λοιπόν πρέπει να είναι συντονισμένη και να εξαρτάται και από τους άλλους στόχους. Την απασχόληση και την παραγωγική σύγκληση μεταξύ των χωρών. Δεν έχει νόημα να τιμωρούμε τις κρατικές επιθετήσεις στα ναυπηγεία ή στα ορυχεία όταν πρόκειται για σημαντικούς τομείς για τη διατήρηση της απασχόλησης σε περιοχές που έχουν πολύ υψηλή ανεργία όπως είναι η Ισπανία. Η ελευθέρωση μπορεί να έχει αποσταθεροτικές συνέπειες επί της οικονομίας. Είμαστε εναντίον λοιπόν να θεωρείται ο ανταγωνισμός φραγμός. Εμάς μας κάνει εντύπωση πώς αντιδρά στην οικονομική κρίση η Επιτροπή με ελευθέρωση και με διεθνείς συμφωνίες ή με μεγαλύτερη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Είμαστε κατά στοιχείων όπως είναι η επιδείνωση των εργασιακών συνθήκων ή τα άλλα που γίνονται στις μεταφορές και που διαπιστώνουμε τον τελευταίο καιρό. Επίσης στην έκθεση ε, δυστυχώς δεν αναφέρεται τίποτα για την παρέμβαση του 13 στο γεωργικό τομέα. Έγιναν καταχρήσεις δεσπόζουσας θέσης σε βάρος των αγροτών. Δεν έχει ερευνήσει επαρκώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ένα σαφές παράδειγμα το βλέπουμε με την διάσωση στην Ισπανία που τελικά κάλυψε σκάνδαλα Επίσης καταδικάζουμε την αδιαφορία που διαπιστώνουμε όσον αφορά τον ενεργειακό τομέα της Ισπανίας, όπως συσσωρεύονται σκάνδαλα, όπου παραβιάζεται η νομική ασφάλεια, οι επενδύσεις για την πράσινη οικονομία και υπάρχουν και άλλα παραδείγματα ολιγοπολίων στον ηλεκτρισμό και καταλήγουν να πληρώνουν οι πολίτες το τίμημα μέσω των ε, λογαριασμών ηλεκτρισμού. Φυσικά και έχω τροπολογίες και ευχαρίστω να τις συζητήσω με τον εισηγητή, όπως και με τους κοιόδες εισηγητές και εννοείται ότι θα σας στείλουμε τις τροπολογίες μας. Ευχαριστώ. σε ευχαριστούμε. Μισελ Ραϊμόντ. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω γερμανικά. Ευχαριστώ πρώτα τον εισηγητή για την έκθεση που υπέβαλε. Νομίζω πραγματικά μπορεί να αποτελέσει βάση για περαιτέρω συζήτηση. Βέβαια, ε, επιθυμώ να επιφέρω και ορισμένες βελτιώσεις. Χαίρομαι που περιλαμβάνει και τον τομέα των μεταφορών, όπου χρειάζεται μεγαλύτερο ανταγωνισμό μεταξύ των διαφορών εταιριών. Αυτό ισχύει και για τις μεταφορές μακρών αποστάσεων. Βεβαίω, το νόημα πρέπει να έχει ο ανταγωνισμό είναι να αποβαίνει προ όφελο των καταναλωτριών και καταναλωτών. Το ίδιο για τον τομέα του περιβάλλοντος. Στην τελευταία του εμφάνιση ενώπιον της παρούσας Επιτροπής, ο προηγούμενος αρμόδιος Επίτροπος είχε πει ότι δεν πρόκειται να ε, λάβει μέτρα για τον ανταγωνισμό μεταξύ των πυρηνικών σταθμών Νομίζω ότι πρόκειται για σημαντική στρέβλωση ωστόσο του ανταγωνισμού στον τομέα της ενέργειας και δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε. Είτε πρόκειται για την πυρηνική ενέργεια, είτε πρόκειται για επιδότηση υπέρ της ατομικής ενέργειας έτσι ώστε να αποβαίνει σε βάρος των ανώσιμων ενεργειών. Αυτό πρέπει να το συζητήσουμε. Το άλλο σημαντικό θέμα έχει σχέση με την φοροδιαφυγή. Περιλαμβάνεται εδώ. Ωστόσο δεν περιλαμβάνεται ο φορολογικός ανταγωνισμός στο μέτρο που είναι νόμος και επιτρεπτός. Αναφέρομαι βεβαίως στην περίπτωση του Λουξεμβούργου, αλλά όχι μόνο. Οποιαδήποτε πολιτική ανταγωνισμού ασκήσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χάνει τη σημασία της εφόσον καταστρέφει τις οικονομίες και τους προϋπολογισμούς των χωρών μελών ο φορολογικός ανταγωνισμός. Δεν μπορούμε να το αποδεχτούμε αυτό ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να τοποθετηθούμε, πρέπει να θεσπίσουμε τις απαραίτητες, απαραίτητα πλαίσια και αυτό πρέπει να μπει μέσα στην έκθεση το ίδιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρειάζεται επαρκή στελέχωση ώστε να μπορεί να αντιμετωπίζει επιθετικά τέτοιες υποθέσεις και ιδίως το νομικό της προσωπικό πρέπει να ενισχυθεί έτσι ώστε να μπορεί να δρά καταλήλως σε περιπτώσεις τέτοιων διαπιστώσεων. Μάλιστα, σας ευχαριστώ. Εσείς ε, ένα λεπτό. Κυρία Ιντφέλτ, μάλιστα θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Δύο ε, ζητήματα με απασχολούν στα οποία θα υποβάλω τροπολογίε. Πιο πολλοί ερωτήσει όμως είναι. Αυτές οι διαρροέ του Λουξεμβούργου για τις φορολογικέ υποθέσεις που διερευνά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα ω κρατικέ επιχορηγήσεις. Πολλές πολιτικές ανταγωνισμού έχουν αποκεντρωθεί στα αρμόδια όργανα. Πώς λειτουργεί όμως αυτό. Διερευνώνται οι σχετικές αποφάσεις των χωρών μελών και ένα άλλο θέμα προδιετίας. Είχαμε την απόφαση Μπόσμαν για τους ε, ποδοσφαιριστές, κάτι που δεν είναι απαραίτητα πολιτική ανταγωνισμού, πάντως έχει κάποια σχέση με την ελευθερία διακίνησης. Υπάρχουν και άλλες ε, περιπτώσεις ε, πιο χαμηλού προφίλ, λιγότερο σημαντικές ίσως, που έχουν σχέση ωστόσο με τον επαγγελματικό αθλητισμό που αποτελεί οικονομική δραστηριότητα και όπου ε, διεθνείς ομοσπονδίες αθλημάτων φαίνεται να βάζουν περιορισμούς πάνω στους αθλητές που είναι συνδεδεμένοι με αυτές. Και έχουν υποβληθεί παράπονα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία άραγε είναι διατεθειμένη να εξετάσει μια τέτοια υπόθεση που ενδεχομένω ε, θεωρεί ότι είναι ίσονο σημασία. Ευχαριστώ ο εισηγητή. Θα είμαι σύντομο. Λάγκεν. Τονίσατε πολλά σημαντικά θέματα που εν τέλει, επί των οποίων εν τέλει θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε. Δεν ξέρω αν θα έχουμε λόγο στις επικοινωνιακές πολιτικές της ε, Κομισιόν, αν όμως το επιθυμεί τόσο πολύ το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, εντάξει, να το βάλω μέσα. Για τα ταμεία, ομολογώ ότι επηρεάστηκα και τέθηκα στον πειρασμό από την, έκθεση, από την περσινή έκθεση και είναι σημαντικό να τοποθετηθεί με κάποια έμφαση αν συνεχίσουμε να συμφωνούμε επί των σχετικών διατυπώσεων, όπως πέρσι. Συμφωνώ εξάλλου ότι θα ήταν καλό να ερωτηθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να εξηγήσει τι έχει επιτύχει και τι όχι, ώστε να υπάρξει μια διαρκής αξιολόγηση του που βρισκόμαστε. Ευχαριστώ, δηλαδή, ευχαριστώ πάντως για τις ε, απόψεις που θέσατε υπόψη μου. Για τον Τιμπόρ ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Συμφωνώ με τα τρία θέματα που αναφέρατε. Για το ζήτημα της διαφθοράς πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τις διατυπώσεις μας. Είτε θα είμαστε πάρα πολύ συγκεκριμένοι είτε όχι. Δεν μπορεί ε, να είναι στο περίπου. Ή θα έχουμε συγκεκριμένε υποθέσεις που θα θέλουμε να τονίσουμε ή θα κάνουμε μια γενική παρατήρηση για προβλήματα διαφθοράς και τις επιπτώσεις που έχουν στις πολιτικές του αγωνισμού. Βεβαίως είμαι ε, πεπισμένος ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε συμβιβασμό που θα ικανοποιήσει ε, τους πάντες. Για τον Ραμόν. Πάλι το ίδιο θέμα, ποιον να κατονομάσουμε, ποιον όχι. Νομίζω και εδώ θα μπορέσουμε όπως και πέρσι να καταλήξουμε σε κάποιο σχετικό συμβιβασμό. Ενστικτοδός θα έλεγα ότι σε μια τέτοια έκθεση όταν εκφράζουμε γνώμη σε ένα χώρο που δεν έχουμε επισήμως αρμοδιότητα, την οποία έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι πιο σόφρον να μην, πιο σόφρον να μην προσπαθούμε να κρίνουμε επί συγκεκριμένων υποθέσεων. Ας δούμε όμως ποια ήταν η διατύπωση που χρησιμοποιήθηκε πέρσι. Από την άλλη μεριά, αν δεν έγινε και τίποτα από πέρσι, η διατύπωση να μην ήταν τόσο κατάλληλη. Θα δούμε πάντως πού μπορούμε να φτάσουμε. Για τον τομέα των μεταφορών που ανέφερε και ο Ραμόν αλλά και η Πράσινη περιλαμβάνεται μοναχά σε, δύο αιτιολογικές σκέψεις, 19 και 20 και απαντώντας ε, στις παρατηρήσεις του Τίμπορ ε, ε, ποιον θέλουμε να αναφερθούμε, σε ποιον θέλουμε να φτάσουμε, δηλαδή για κοινωνικό ντάμπινγκ και άλλα σχετικά θέματα. Αφού εκπροσωπούμε τους καταναλωτές, Νομίζω ότι είμαστε και πιο σημαντικοί εκπρόσωποι των καταναλωτών. Έτσι δεν είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Άρα βεβαίω μπορούμε να αναλάβουμε το καθήκον αυτό. Συμφωνώ λοιπόν και με αυτό. Για τον τομέα τη ενέργεια, συμφωνώ με την παράτηση που έγινε για τι καθυστερούμενε πληρωμέ και τη σχετική οδηγία μπορεί να έχει σχέση βεβαίω με το νομοθέτημα για τον ανταγωνισμό. Θα το συζητήσουμε αυτό μεταξύ των σκιωδών εισηγητών οι διαρροές του Λουξεμβούργου ε, δεν τις έχω βάλει διότι υπέβαλα το σχέδιό μου πριν να γίνει γνωστή η υπόθεση αυτή. Θα υπάρξει τοποθέτηση του Κοινοβουλίου και γι' αυτό και για την φοροδιαφυγή γενικότερα. κυρίως μέσα στο καθεστώς των κρατικών επιδοτήσεων ότι πράγματι πρέπει να γίνει μια πραγματική σε βάθος έρευνα κατά του Λουξεμβούργου και άλλων κρατών και να περιληφθούν και οι εφιστάμενες υποθέσεις αλλά και ενδεχόμενε νέε. Για την απόφαση Μπόσμαν, την οποία γνωρίζω καλά, δεν μου ήρθε στο μυαλό, αλλά ευχαρίστως να βάλω μια παράγραφο για τον επαγγελματικό αθλητισμό, κάπου θα συμφωνήσουμε δεν είναι απαραίτητα καλό να βάλουμε μέσα όσο το δυνατόν περισσότερους τομείς. Από αυτά που μου εξήγησε η γραμματεία, εγώ κατενόησα ότι είμαστε περιορισμένοι σε ό,τι αφορά τον αριθμό των σελίδων κτλ. Βέβαια αυτό δεν ισχύει ο περιορισμός, δεν ισχύει για τις τροπολογίες. Μπορούμε λοιπόν ενδεχομένω να βάλουμε και τέτοια πράγματα μέσα, ώστε να οριοθετήσουμε από την αρχή τη θέση μας. Ευχαριστώ για τις διάφορες παρεμβάσεις. Ναι, αλλά πρέπει να, να καταλήξουμε κύριε Λάγκεν προτείνω να διεξαχθεί νέα συζήτηση για το θέμα όταν θα έχουν κατατεθεί τροπολογίες και να μην, να μην συναντηθούν οι, σκιο, οι σκιώδεις πριν. Θα υποβληθούν τουλάχιστον 500 τροπολογίες. Κύριε Μέσα Σουμίτ, να αναβάλλετε την ε, έκθεση σας για του χρόνου. Ευχαριστώ. Ο πρόεδρος Γκουαλτιέρη, οκ, 27 Νοεμβρίου, 12η μεσημβρινή, προθεσμία κατάσταση τροπολογιών, οι οποίες θα συζητηθούν 21 Ιανουαρίου, θα ψηφιστεί στις 27 και ελπίζουμε στην Ολομέλεια να καταλήξει στις 25 Δευτέρου. Λίγη συνεδρίαση, η επόμενη συνεδρίαση την Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, 7.30 το βράδυ στο Στρασβούργο. Ευχαριστώ.